Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Άρχεται η συνεδρίαση. Οι αρχές αρμόδιες από την Πορτογαλία μου απίθυναν έτοιμα ανάκληση της άρσης ασυλίας του κυρίου Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες στο πλαίσιο ποινική διαδικασίας εις βάρος του από τις ε, αρχές δίωξης της πόλης του Πόρτο. Το σχετικό αίτημα έχει αναπεμφθεί στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη την κοινή συζήτηση για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο. Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. και δίνω το λόγο σε μία από τις συντάκτριες, την κυρία Γκαρσία Πέρες. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έλλειψη εκπροσώπησης ε, των γυναικών στα διάφορα πεδία της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής είναι ε, εκδήλωση της ανισότητας στην κοινωνία. Άρα χρειάζεται να προωθήσουμε την πολιτική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. <clears throat> το 2013 το κοινοβούλιο μας έλαβε θέση έναντι της ε, πρότασης της Επιτροπής για την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων ούτω ώστε να υπάρξουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις εκπροσώπησης των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο ούτω ώστε και στον οικονομικό τομέα λοιπόν να υπάρξει ίση εκπροσώπηση. Έκτοτε πέρασαν πέντε χρόνια. Πέρασαν διάφορες προεδρίες και το θέμα αυτό έχει μπλοκάρει στο Συμβούλιο. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να προωθήσουν μια πιο ίση Ευρώπη, καταλαβαίνοντας ότι μια Ευρώπη πιο ίση Πρέπει οπωσδήποτε να είναι μια Ευρώπη όπου είναι πραγματικότητα ίση εκπροσώπηση των γυναικών σε όλου του τομεί τη οικονομική ζωή. Έπρεπε να αλλάξει η κυβέρνηση στην Ισπανία για να δοθεί μια όθηση και στο Συμβούλιο ούτω ώστε να επιδιώξουμε επιτέλου να υπάρξει μια συμφωνία για το θέμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιούροβα για την όθηση που διαπιστώνω ότι δίνει, ούτω ώστε η Επιτροπή μαζί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να επιτρέψουν να ολοκληρωθεί πριν από το τέλο τη θητεία ή μια πρωτοβουλία για την ισότητα εκπροσώπηση που είναι θεμελιώδη. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε τα δικαιώματα των γυναικών να συνεχίσουν να καθυστερούν να εφαρμοστούν. Οι γυναίκε. πρέπει οπωσδήποτε να εκπροσωπούνται ισότιμα, να υπάρχει ισότητα ευκαιριών. Και το κοινοβούλιο μα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει σαφή θέση και να, να καλέσει την Ρουμανική Προεδρία να κάνει την τελευταία προσπάθεια, ούτω ώστε όπω ε, και η κυβέρνηση τη Ισπανία που προωθεί την ε, πρωτοβουλία αυτή, ούτω ώστε να καταφέρουμε οι γυναίκε να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Είναι θεμελιώδε για να προχωρήσουμε προ μια Ευρώπη πιο ίση και πιο δίκαιη. Σα ευχαριστώ πολύ. Συντάκτη επίση η κυρία Χάουταλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και είναι πιστεύω πολύ σημαντική στιγμή τώρα να διαπιστώσουμε πως ουδής λόγος μας αποτρέπει από την υιοθέτηση αυτής της οδηγίας του 2012, από την εισαγωγή αυτής της οδηγίας, που θα επέβαλε την υποχρέωση καταχωρημένες ε, ε, εταιρείε, επιχειρήσεις να φτάσουν στο 40% ποσοστό για τα μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Με καταπλήσει του γεγονό ότι ορισμένα κράτη-μέλη επικαλούνται ακόμη την επικουρικότητα. Πώ το κάνουν αυτό, Υπάρχουν ε, επιχειρήσει ευρωπαϊκέ που δρούν όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής. Επομένω, οπωσδήποτε είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, το αντικείμενο τη οδηγία. Και επίση είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφορά, η συμπερίληψη και η ποικιλία μεταξύ αυτής βέβαια και της διάστασης του φύλου και για την ε, διαφοροποίηση και την ανάπτυξη των στρατηγικών των επιχειρήσεων. Τρίτον, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν ικανές γυναίκες. Αυτό είναι μια πρόφαση μόνο μια ε, νοοτροπία στην οποία επικρατούν οι άντρε. Ναι, μπορεί να μην είναι ορατέ οι γυναίκε γιατί μερικέ φορέ δεν έχουν αυτή τη νοοτροπία ή τη συμπεριφορά που ε, προέρχεται από την ε, νοοτροπία όπου επικρατούν την ανδροκρατούμενη, αλλά πάντως είναι εξίσου ικανές με τους άντρες τουλάχιστον για να ανταποκριθούν σε προκλήσεις. Και έτσι πρέπει και σε αυτό το βαθμό να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις. Είχαμε πει αρχικά εθελοντικά, στην εισαγωγή των γυναικών, όπου διαπιστώσαμε στο το 17-18 ήταν μόνο το 26% των διοικητικών συμβουλίων γυναίκες, τις μεγαλύτερες από τις καταχωρισμένες επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλη διαφορά από το 7,5% στο 43% που αποδεικνύει πως χρειάζονται μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μας οδηγήσουν στην αναρμόνιση στη σημαντική αυτή πτυχή. Ευχαριστώ την Ισπανική κυβέρνηση, η οποία επιτέλους έριξε μια δεύτερη ματιά στην υπόθεση αυτή. Και ελπίζω ότι με την ε, Προεδρία της Ρουμανίας θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την πρόταση και πριν από τις ευρωεκλογές να μπορέσουμε να διακηρύξουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει ένεργα μια σύγχρονη και επιχειρηματική κουλτούρα και νοοτροπία με ισότιμη ε, προώθηση και ε, εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην συμβαίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους Συμβουλίου τώρα η Υφυπουργός κυρία Σότ την οποία και ευχαριστώ για την παρουσίαση της εδώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, μεγάλη χαρά που σας βλέπω εδώ σήμερα για αυτή τη σημαντική συζήτηση. Ξεκινώντας θέλω να πω πώς η ισότητα των φύλων εγγράφεται στο επίκεντρο του οράματος για την Ευρώπη του Συμβουλίου και σε πολλέ διακήρυξει του Συμβούλου έχει επιβεβαιώσει αυτή την προσήλωση, αλλά και στην νομοθεσία που αναπτύξαμε σύν το χρόνο από κοινού με το Κοινοβούλιο. Και επίσης θέλω να υπενθυμίσω τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που από κοινού ανεκήρυξαν Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017. Η ισότητα των φύλων λοιπόν έχει μεγάλη σημασία εδώ ισότητα των φύλων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να προάγεται σε κάθε τομέα συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσώπησης σε όρους αγοράς εργασίας και τις συνθήκες απασχόλησης και προαγωγής στη σταδιοδρομία. Άνδρες και γυναίκες έχουν δικαίωμα σε ίση αμοιβή για δουλειά ίσης αξίας. Αυτή η προσήλωση βεβαίως και καταχωρίζεται και προέρχεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες αλλά και από τις εθνικές μας νομοθεσίες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί το τελευταίο, την τελευταία πεντηκονταετία, αλλά και περισσότερο βλέπουμε ότι υπάρχουν πρακτικές των οποίων ακόμη δεν έχουμε τον έλεγχο ή την επιστασία. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω σαν παράδειγμα ότι υπάρχει ακόμα σημαντική διαφορά ως προς την αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, 16,2 ποσοστιαίες μονάδων και πάντα είναι χαμηλότερες οι αμοιβέ των γυναικών από, τους, από αυτές των ανδρών. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί ισότητα. Το ζήτημα λοιπόν της αμοιβή θα το ε, καλύψουμε σε συμπεράσματα του Συμβουλίου που αναμένουμε να υιοθετηθεί στον Συμβούλιο Άψικο τον Ιούνιο. Για να υλοποιηθούν όμως και οι άλλες ε, υποσχέσεις του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων χρειαζόμαστε δράση από την Επιτροπή, από τους συνομοθέτες, από τα κράτη-μέλη. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα μας ζητήσατε συγκεκριμένα να ε, σχολιάσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια οδηγία που θα βελτίωνε την ίση εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των ε, επιχειρήσεων. Με λύπη μου σας λέω σήμερα ότι δυστυχώς όπως όλους το γνωρίζετε υπάρχει ανασχετική μειοψηφία στο Συμβούλιο. Η τελευταία μας συνεδρίαση για το θέμα αυτό είχε λάβει χώρα υπό την Προεδρία της Μάλτας το 2017. Η συζήτηση δε δεν συζητήθηκε έκτοτε ε, επισήμω από το Συμβούλιο. Όπως έχει τώρα η κατάσταση παραμένει δηλαδή σε αδιέξοδο αυτή η υπόθεση. Πλην όμω ε, ευρεία είναι η συνένεση στην Ευρώπη ως προς την ανάγκη για προαγωγή της ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά Συμβούλια, όσο και αν έχουν διαφορετικέ προσεγγίσεις τα κράτη-μέλη, γιατί δεν αμφισβητείται η βάση αυτή τη στόχευση και έτσι η Ρουμανική Προεδρία στοχεύει να διευκολύνει τι συζητήσει και συνομιλίε επί του Συμβουλίου, προκειμένου να διερευνηθούν υπεραιτέρω ε, διάβλη για πρόοδο. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην πρόταση για μία οδηγία για, την, ε, για το συγκερασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου για γονείς ε, και εδώ θα ήθελα να πω ότι οι συνομιλίες μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου οδήγησαν σε μια προσωρινή συμφωνία στον έκτο τριμερή διάλογο που έλαβε χώρα στις 24 Ιανουαρίου. Επιτυχία η οποία κατέστη δυνατή και χάρη στην εξαιρετική πρόοδο που ε, οφείλουμε στη Βουλγαρική και Αυστριακή Προεδρία. Η διευκόλυνση λοιπόν του συνδυασμού οικογενειακού και επαγγελματικού βίου είναι τεράστιο πυλώνα τη πολιτική απασχόληση. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διευκολύνουμε του πολίτε μα να συγκεράσουν τον επαγγελματικό με τον οικογενειακό βίο, πράγμα το οποίο είναι ακόμη πιο σημαντικό και λόγω της δημογραφικής κατάστασης και των εξελίξεων στην αγορά εργασίας όμως. Αφενό λοιπόν πρέπει να καταστήσουμε να εξασφαλίσουμε πως η Ευρώπη θα έχει γυναίκες με την υψηλή τους κατάρτιση και τις δεξιότητές τους ικανές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας ε, πράγμα το οποίο έχει και οικονομική σημασία και αντίκτυπο ταυτόχρονα είναι και τα δικαιώματα και από την άλλη θα πρέπει οι γυναίκες και οι άνδρες να έχουν την δυνατότητα να κάνουν παιδιά χωρίς να πρέπει να κάνουν την επιλογή μεταξύ του να είναι γονείς ή να έχουν μια θέση εργασίας και βεβαίως επισημαίνω ότι πολύ πιο συχνά οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια τέτοια επιλογή. Έτσι λοιπόν, εάν οι εργαζόμενοι που έχουν οικογένεια έχουν κατάλληλα δικαιώματα για άδεια γονεακή ή άλλη και αυτά τα δικαιώματα ε, είναι κατανεμένα τόσο στους άντρες όπως και στις γυναίκες, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ωστόσο πρέπει και τα εθνικά συστήματα να τροποποιηθούν. Στη γυναίκα, στην Ευρώπη δεν μπορεί να πει κανεί ότι μία λύση μπορεί να ισχύει για, το, κάθε, για όλα τα κράτη αδιακρίτως. Ε, έτσι λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές πραγματικότητες και κοινωνικά συστήματα μεταξύ των κρατών μελών και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αλλά και να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Αυτές ήταν κάποιες από τις σκέψεις που εκλήθημε να συζητήσουμε κατά τις συνομιλίες για την οδηγία για την εξορόπιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Εύκολη δεν ήταν η συζήτηση, αλλά χαίρομαι ότι διότι ευρέθη μια λύση η οποία εξασφαλίζει με την βελτίωση των ε, απαιτήσεων και των προδιαγραφών τη δυνατότητα για την εξορρόπηση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου και ελπίζουμε και το Κοινοβούλιο είναι ικανοποιημένο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Τώρα την, το λόγο θα λάβει η Επίτροπος κυρία Γεωρόβα, την οποία και ευχαριστώ για την παρουσία της. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο επειδή έθεσε το σημαντικό αυτό θέμα στην σημερινή μερίσια διάταξη. Είμαι ευγνώμων για την ε, στήριξή σας στην ε, πρόταση της Κομισιόν που στόχο έχει να βελτιώσει την ισορροπία των δύο φύλων σε εταιρικά διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών. Εδώ και πέντε χρόνια σχεδόν είμαι τώρα Επίτροπος για την ισότητα των φύλων και είμαι υπερήφανη για την συλλογική μας δουλειά ειδικά για την ε, οριστικοποίηση του πακέτου για την ισορροπία μεταξύ εργασιακού και οικογενειακού βίου, ανησυχώ όταν το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα λέει στην ε, τελευταία του έκθεση, στον δίκτυ του, ότι σε κάποιου τομεί ε, πηγαίνουμε πάρα πολύ αργά. Όταν ε, δημοσίευσαμε τα πιο πρόσφατα νούμερα, δεν έκρυψα την απογοήτευσή μου για τις εξελίξεις αυτές, παρόλες τις προσπάθειες που κάνουμε. Ο δείκτης ισότητας των φύλων δείχνει πως η ισότητα στην λήψη αποφάσεων εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλότερα από όλους τους άλλους τομείς που αξιολογήθηκαν στον δείκτη παρά την νομοθεσία σε κάποια κράτη που εντωμεταξύ εγκρίθηκε. Όλοι γνωρίζουμε τις μελέτες που δείχνουν σαφώς τα ωφέλη της ποικιλομορφία ε, στα διοικητικά συμβούλια ωφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία βεβαίως. Η Κομισιόν βεβαίως παραμένει προσιλωμένη στην οδηγία αυτή. Οι γυναίκες παρά τις ικανότητες τους συνεχίζουν να έχουν να αντιμετωπίσουν εμπόδια στην είσοδό τους ε, στα διοικητικά συμβουλία και σε ηγετικές θέσεις. Η οδηγία αυτή θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε την πρόσβαση ταλαντούχων γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις και να επιταχύνουμε την οικονομική ανάπτυξη. Όταν αποκτήσουν εξουσία οι γυναίκες θα έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο θα διευρύνει την ισότητα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως πρόκειται για μια πρόταση αναλογική και ευέλικτη, φιλική προς την επικουρικότητα που δίνει μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη για το πώς θα επιτευχθεί αυτή η πρόοδος. Επίσης, είναι ένα νομοθέτημα το οποίο είναι ουδέτερο ως προς τα φύλλα. Αφορά το φύλλο το οποίο υποεκπροσωπείται ε, όταν έχει ανάλογα προσόντα, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες. Και βεβαίως ε, τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να διατηρήσουν τα υφιστάμενα μέτρα που έχουν για να βελτιώσουν την ισορροπία των φύλων στα ΔΣ. Σύμφωνα με τους αριθμούς μας, τα κράτη τα οποία έχουν περάσει την νομοθεσία σημειώνουν κάποια πρόοδο. Όσα δεν έχουν την νομοθεσία έχουν απλά κολλήσει. Βλέπουμε λοιπόν τον θετικό αντίκτυπο της νομοθεσίας αυτής σε πολλά παραδείγματα. Η πρόταση της Κομισιόν έχει ευρία στήριξη από το Κοινοβούλιο και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι και επίσης έχει την στήριξη της πλειοψηφίας των κρατών μελών. Κατά την απόψή μου μπορούμε να καταλήξουμε σε μια γενική προσέγγιση και θα επαναλάβω αυτό το οποίο υπόθηκε ότι υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη από την Ισπανική κυβέρνηση ε, τους οποίους είχα επισκεφθεί ούτως ή άλλως πρόσφατα και αυτό μας δείχνει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για να πείσει και τις ε, χώρες εκείνες που ακόμα είναι αντίθετες. Και επίσης ε, βασιζόμαστε ιδιαίτερα και στην Ρουμανική Προεδρία που επίσης είναι πολύ αποφασισμένη. Εν ώψη του Συμβουλίου του Μαρτίου σκοπεύουμε να ξεμπλοκάρουν οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο και η υπουργό ανέφερε και το Συμβούλιο του Ιουνίου που πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το επέσχυντο αυτό ζήτημα του μισθολογικού χάσματος. Οπότε η Κομισιόν ελπίζει ότι η Ρουμανική Προεδρία θα καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για το θέμα αυτό για να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ακούμε τις ε, πολιτικές ομάδες. Σε αυτή τη φάση δεν δεχόμαστε μπλε κάρτα διότι δεν μας το επιτρέπει ο χρόνος. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η κυρία Κοσλόφσκα Ράγεβιτς. Δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Άκουσα όλα όσα υπόθηκαν και φαίνεται ότι όλοι συμφωνούμε. Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Κομισιόν, όλοι υποστηρίζουν την οδηγία επιπλέον. Κανένα κράτος μέλος δεν αμφισβητεί του στόχου τη οδηγία. Οπότε η ερώτησή μου είναι γιατί δεν έχει ακόμα τεθεί ενισχύ και γιατί σε κάποια κράτη-μέλη η παρουσία γυναικών σε εισηγμένε εταιρείε στα ΔΣ είναι μόλις 7%. Εάν το επιχείρημα της επικουρικότητας ήταν σοβαρό, τότε τα κράτη-μέλη θα πρότειναν κάποιες λύσεις για να αλλάξει η κατάσταση. Γιατί δεν νομίζω ότι κανείς με κοινή λογική θεωρεί ότι η διαφορά 7 με 43% είναι κάτι το σωστό. Το ίδιο επίσης ε, και για τα υπόλοιπα ζητήματα. Είναι προφανές ότι δεν είναι ζήτημα ικανοτήτων. Άλλοι μηχανισμοί λειτουργούν. Πρέπει να αντιδράσουμε λοιπόν σε επίπεδο κρατών μελών. Γι' αυτό κάποια αντίδραση πρέπει να υπάρξει. Εγώ στηρίζω αυτή την φανταστική οδηγία της Επιτρόπου της κυρίας Ρέντινγκ και έχει φτάσει πια η στιγμή οι ικανότητες να κρίνουν ποιος θα είναι διευθύνων ή διευθύνουσα σύμβουλος και ποιος θα είναι στο ΔΣ. Πρέπει να έχουμε σαφή κριτήρια και να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Δεν θα πρέπει αυτοί οι οποίοι ορίζουν τα μέλη του ΔΣ να ορίζουν τους κολλητούς τους που τους ξέρουν χρόνια. Εξ ονόματος του ΕΛΚ θα ήθελα να πω ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω της έλλειψης ε, υποδομών ε, για τα παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ε, ζωής. Θα πρέπει λοιπόν να συγχαρούμε την Προεδρία για το αποτέλεσμα του διαλόγου που μόλις ολοκληρώθηκε και να στηρίξουμε την οδηγία στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρέγνη, στους Δημοκράτες, δύο λεπτά. Μικρόφωνο, μικρόφωνο. Ωραία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε χρειαζόμαστε ικανές, έξυπνες γυναίκες και άνδρες στην κεφαλή των ε, επιχειρήσεων, των ΔΣ. Πριν από 7 χρόνια, 7 χρόνια έφερε την πρόταση η Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Διαπιστώσαμε ότι χρειαζόμαστε αντικειμενικά κριτήρια επιλογής και να είμαστε και πρακτικοί. Κοιτάμε τι γίνεται στις ε, χώρες ποια χώρα έχει περάσει ανάλογους νόμους, ε, ποια έχει κάνει πρόοδο με θελοντικά μέτρα. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδείχθηκε πάρα πολύ πρακτικό ότι χρειάζονται αντικειμενικά κριτήρια τα οποία μετά θα πρέπει να εφαρμοστούν. Δεν πάμε πουθενά με τον προαιρετικό χαρακτήρα. Χρειάζεται να είναι κάτι το υποχρεωτικό και με κυρώσεις η ισότητα είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει τόσο μεγάλη πρόοδος σε τόσες πολλές χώρες. Είναι δηλαδή κάτι το θαυμάσιο για τις επιχειρήσεις και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Και τι συμβαίνει τώρα, πάρα πολλές χώρες κρύβονται πίσω από την νομική βάση. Ε, τι σημαίνει αυτό δηλαδή είναι δεδομένη η νομική βάση, γιατί μόνο οι χώρες εκείνες οι οποίες δεν έχουν επιτύχει καμία πρόοδο κρύβονται. Γι' αυτό ζητώ από την Ρουμανική Προεδρία την οποία χαιρετίζω καθώς επιτέλους ε, φέρνει αυτό το θέμα στο προσκήνιο να τραβήξει την κουρτίνα πίσω από την οποία κρύβονται κάποιες χώρες, χώρες όπως η Ουγγαρία που βλέπουμε τι γίνεται. Υπάρχει μάλιστα οπισθοχώρηση εκεί. Γι' αυτό ζητάω επιτέλους από την Προεδρία του Συμβουλίου να ζητήσει να μάθει αυτές οι χώρες επιτέλους τι έκαναν και να ψηφίσουν επιτέλους στο Συμβούλιο γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εδώ πέρα μια πολύ ισχυρή θέση είναι ενωμένο και χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι επανήλθε επιτέλους αυτή η πρόταση. Βυσνιεύσκα, παρακαλώ για δύο λεπτά και να σέβεστε το χρόνο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εάν δούμε τον δίκτυ ισότητας, βλέπουμε ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα ΔΣ εταιριών στις υψηλόβαθμες ε, θέσεις. Γιατί οι γυναίκες είναι ικανότατες, ε, έχουν προσόντα, θέλουν να δουλέψουν, είναι φιλόδοξες. Σαφώς ε, δεν έχουν λιγότερο ταλέντο. Γιατί λοιπόν τόσο λίγες γυναίκες είναι σε αυτές τις υψηλόβαθμες θέσεις. Για εμένα ο βασικός λόγος είναι ότι η σταδιοδρομία τους ε, εξελίσσεται με πιο αργό ρυθμό. Θέλουν όχι μόνο να τις εκτιμούν στη δουλειά, αλλά και ως μητέρες. Πρέπει να συνδυάσουν ε, τη δουλειά με την οικογενειακή ζωή, θέλουν να γίνουν μητέρες, να φροντίζουν τα παιδιά τους. Γι' αυτό μένει πίσω η σταδιοδρομία τους. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στα Δέλτα σίγμα, αλλά όχι με τεχνητό τρόπο με οδηγίες αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να προτείνουμε λύσεις που θα δώσουν στις ε, γυναίκες την δυνατότητα να συνδυάσουν την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή γιατί χρειαζόμαστε λύσεις ε, που θα μπορέσουν να εγγυηθούν αυτήν την ισορροπία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και θεωρώ ότι οι λύσεις αυτές προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι πολύ πιο επιτυχής. Η Eurostat μας λέει πως ε, το μισολογικό χάσμα διαφέρει πολύ ανάλογα με το κράτος μέλος, αλλά υπάρχουν χώρες όπου είναι πολύ ψηλό. Ευτυχώς η Πολωνία είναι μεταξύ των πέντε κρατών μελών ε, με το χαμηλότερο μισολογικό χάσμα και ευτυχώς ε, τελευταία έχουμε όλο και περισσότερες γυναίκες σε υψηλές ε, θέσεις χωρίς να ληφθούν τέτοια τέχνητα μέτρα. Σας ευχαριστώ. Μπιλμπάο Μπαραντίκα, δύο λεπτά για την Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλε τι προσπάθειε και για τη δέσμευσή σα για τι πρωτοβουλίε αυτέ. Βλέποντα το περιεχόμενο αυτών των ερωτήσεων και βλέποντα πώ έχουν φρακάρει στο Συμβούλιο αυτέ οι προτάσει για να υπάρξει ισότητα στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, θέλω να ζητήσω τρία πράγματα από τι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει. Συνέπεια, μακρόπνο όραμα και θάρρο, Πρώτα απ' όλα συνέπεια. Μα εδώ μας λένε συνέχεια για την ευφυή ανάπτυξη, για μια οικονομία που θα βασίζεται στο ταλέντο. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε το μισό ταλέντο που διαθέτουμε, που είμαστε εμεί οι γυναίκε, να μην φτάνει εκεί που μπορεί να βοηθήσει πιο πολύ. Στα διοικητικά συμβούλια, στα κέντρα λήψη αποφάσεων. Ο, και όπω αποδεικνύουν όλε οι μελέτε, αποδίδει περισσότερο. Εκεί θα επιτύχει, όπως το διαπιστώνουν όλες οι εμπειρίες που κάναμε σε ορισμένες, όλες μελέτες που κάναμε σε ορισμένα κράτη-μέλη. Να έχετε το θάρρος να δείτε αυτή την πρόταση από την πλευρά της αποδοτικότητας. Ε, εφόσον φοβάστε να το δείτε από την πλευρά της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ε, ίσης ευκαιρίας. Μακρόπνο όραμα τώρα. Η Ευρώπη είναι μία από τις περιοχές του κόσμου που προωθούν πολιτικέ ε, πολιτικές ισότητας. Ας αξιοποιήσουμε αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Άλλε περιοχές ε, ασχολούνται τώρα με ιδέες που εδώ και χρόνια τις ε, προωθούμε. Α κάνουμε το τελευταίο βήμα. Όπως είπαμε, όχι μόνο είναι δίκαιο και δημοκρατικό, αποδίδει, είναι κερδοφόρο. Όλα τα ωφέλη που θα ε, εξαγάγουμε από την πρόθεση αυτού του ταλέντου θα μας κάνει πιο ανταγωνιστικού. Επίσης, θάρρος. Πολλοί άνδρες σκέφτονται μόνο με αρσενικό τρόπο έναντι αυτού του φρακαρίσματος. να ξεπεράσετε τον φόβο σα. θα κερδίσετε. Είναι πολύ σημαντικό να ασχολείται κανεί με τα παιδιά, με του ηλικιωμένου. Είναι καταπληκτικό να έχει κανεί αυτή τη μαγική ευκαιρία να κάνει μια, έναν υπόθηκο δάνειο σε ένα σπίτι. Έτσι θα αξιοποιήσετε αυτό το τμήμα τη ζωή σα. Θα σα βοηθήσει να εξασκήσετε την συναισθηματική σα ε, νοημοσύνη. Θα σα συνδέσει με άτομα, με τι εμπειρίε, με τα προβλήματα, με τι ε, ευθύνε που αιώνε αποφεύγεται. Είμαι πεπισμένη ότι ένα κόσμο όπου και οι άνδρες θα αναλάβουν αυτές τις προκλήσεις θα είναι πολύ καλύτερος. Ευχαριστώ πολύ. Γουρτασούν για τους πράσινους. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε το διέξοδο για αυτή την οδηγία. Δεν έχει προωθηθεί το θέμα αυτό. Θα έπρεπε η Ρουμανική Προεδρία και το Συμβούλιο να προωθήσει αυτό το θέμα μέχρι το τέλος της θητείας. Γιατί όπως είπαμε έχει φρακάρει από το 2012. Θα πρέπει να υπάρχει 40% ποσόστοση για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Είναι απαραίτητο αυτό. Είναι απαραίτητο γιατί η οικονομική ισχύ είναι βασική για την ισότητα φίλων και έχει λειτουργήσει πολύ θετικά. Δεν τα επέλυσε όλα τα προβλήματα, αλλά τι επιχειρήσει που είναι στα χρηματιστήρια υπάρχει ψηλό ποσοστό γυναικών. Και δεν είναι θέμα όπου μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από την επικουρικότητα, όπω κάνουν πολλά κράτη-μέλη. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η ισότητα φύλου είναι στόχος που αναφέρεται στις συνθήκες και η οικονομική δύναμη είναι βασικό θέμα για να υπάρχει ισότητα. Και δεύτερον, γιατί οι ανισότητες στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ορισμένε χώρε 7,4 μόνο, με 63% σε άλλε. Στα διοικητικά συμβούλια είναι τεράστια αυτή η ανισότητα, τεράστιο αυτό το χάσμα. Χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να επιτρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το χάσμα. Όπω είπαμε, η Νορβηγία είναι σίγουρα επιτυχία, δεν τα επέλυσε όλα και μπορούμε να, τα, να εξαγάγουμε ε, πορίσματα. Αλλά τα πορίσματα είναι τα εξή. Ένα είναι να είναι γυναίκε στα δυτικά συμβούλια, το βασικό όμω είναι να είναι και στι ανώτερε θέσει. Το να φτάσουμε στο πρώτο δεν σημαίνει πω επιτυγχάνουμε και το δεύτερο. Και αυτό που μα διδάσκει η εμπειρία τη Νορβηγία είναι ότι και η εφαρμογή δημιουργεί προβλήματα. Όμω από το 2013 το Κοινοβούλιο είπε να υπάρχουν κυρώσει για τι επιχειρήσει που δεν θα επιτυγχάνουν αυτού του στόχου. Για παράδειγμα, να μην συμμετέχουν στι δημόσιε προμήθειε, αν δεν έχουν φτάσει στο 40% που ανέφερε η οδηγία. Οπότε, είναι ένα βασικό τμήμα τη ε, νομοθεσία για να υπάρξει ισότητα. Εγώ θα ήθελα και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να επιχειρήσουν να μα στείλουν καλέ ειδήσει για το θέμα αυτό. Γιατί εμεί εδώ νομίζω ότι ομόφωνα σε αυτή την αίθουσα υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Εκ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Γιατί λοιπόν μόνο 24 ε, από τις 400 ε, θέσεις ε, στις επιχειρήσεις στη Γερμανία που είναι στο χρηματιστήρια υπάρχουν γυναίκες και δεν υπάρχει καμία πρόεδρος. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε φτάσει σε κάτι καλύτερο. Αυτό είναι ντροπή. Και παγκόσμια δεν είναι καθόλου καλύτερη η κατάσταση. Από τις 500 ε, μεγαλύτερε επιχειρήσεις, μόνο τρει γυναίκες είναι επικεφαλής. Είμαστε στο 2019 και το συζητάμε ακόμη. Αυτό είναι ντροπή. Μας λέτε ότι είμαστε τόσο προοδευτικοί, αλλά υπάρχουν πολλοί που έχουν ε, ξεπερασμένες ε, αντιλήψεις ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι στο σπίτι ή σε ε, χαμηλόμιστε δουλειέ. γιατί δεν είναι κατάλληλε, λένε, για τι ε, ηγητικέ θέσει ε, στην οικονομία. Μα πόσο θα κρατήσει αυτή η κατάσταση. Αν δεν υπάρξουν δεσμευτικοί κανόνε, δεν θα επιτύχουμε τα ποσοστά που θέλουμε ε, για τι γυναίκε τα διοικητικά συμβούλια και τα υποπτικά συμβούλια. Δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω συζητήσει. Ο κόσμο δεν είναι κόσμο των ανδρών. Είναι κόσμο για όλα τα φύλλα. Σε οποιοδήποτε φύλλο και να ανήκετε. Πρέπει να πούμε σε αυτούς που είναι κατά των γυναικών και έχουν αναχρονιστικές αντιλήψεις ε, στις διοικητικέ θέσεις ότι έχει περάσει η εποχή τους. Παρακαλώ, Πάρκερ, για δύο μισή λεπτά. Η FTT. Η οδηγία για τις γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο όχι μόνο είναι προσβλητική, αλλά είναι και πατερναλιστική έναντι των γυναικών αυτών, οι οποίες κέρδισαν με το σπαθί τους και την αξία τους τις θέσεις τους. Δηλαδή μια γυναίκα η οποία διαπιστώνει ότι έχει επιλεγεί μια ποσόστοση στη θέση της και όχι μέσω λόγω των δεξιοτήτων της, αποδεικνύει ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες και δεν μπορούν να επιτύχουν μόνο τους την επιτυχία. Πώς ε, δικαιολογείται όμως η κατάσταση σε σχέση με τις γυναίκες που είναι σε χαμηλότερα επίπεδα των, ε, της ιεραρχίας της επιχειρήσης και που δεν τις πρόχνει κανείς να πάνε πιο πάνω ή τα καταφέρουν μόνες τους. Είδαμε ότι και με την Ορβηγία ακόμα και στα συστήματα αυτά μόνο 7% των γυναικών έφτασαν στα διοικητικά συμβούλια. Αυτή η ιστορία με τις ποσοστώσεις Πού θα σταματήσει. Πρώτα μιλήσατε για ποσοστώσεις για γυναίκες και άντρες. Μετά θα συνεχίσουμε πάντα με κατηγοριοποιήσεις και με ποσοστώσεις ατελείωτες. Για άλλη μια φορά, ακόμα περισσότερη παρέμβαση και επέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρώπη. Ναι, οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να βρουν μια δουλειά και να την κρατήσουν, αλλά εδώ επιβάλλεται μια σειρά από και απειλές και αυτό είναι μεγάλη απογοήτευση για τι επιχειρήσει. Ε, μπορεί να οδηγήσει μεγάλα προβλήματα τι επιχειρήσει οι οποίε δεν καλύπτουν τι ποσοστώσει. Οι ποσοστώσει δεν λύνουν κανένα πρόβλημα ανισότητα. Και είναι πράγματι αντιπαραγωγικέ. ΕΝΦ, Σόλτεκ, 2.30. Πρόεδρε. Αυτή η φεμινιστική παράνοια βλέπω να συνεχίζεται. Τι γυναίκες θέλουμε να τι κάνουμε άντρε και τους άντρε γυναίκες. Δεν καταλαβαίνω. Αρρώστια είναι, είναι τίποτα άλλο. Αλλά και ενώ κάποτε ήταν και φεδρό, όπως όταν ψηφίσαμε για το θέμα των γυναικών στη γεωργία που δεν είναι αρκετές ε, οι βοσκοπούλες μπορεί να ήταν εφεδρό. Αλλά όταν μιλούμε για γυναίκες ε, στα διοικητικά συμβούλια των συγκεκριμένων επιχειρήσεων ε, τότε γίνεται επικίνδυνο και ανοησία. Ας βγουν μερικοί άντρες να πούνε ότι είναι γυναίκες και έτσι καλύπτεται και το θέμα της ισορροπίας των φύλων. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό όμως και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Ε, βέβαια, όλη την νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο δίνει μόνο το τυποθήτο και τελικά είναι πολύ κακή η νομοθεσία και όσο πιο κακή είναι τόσο πιο υπεύθυνο είναι και το κοινοβούλιο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με νομοθεσία η οποία παρεμβαίνει στην οικονομική ελευθερία των επιχειρήσεων αλλά και στην εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Βλέπουμε διάφορες τέτοια, διάφορα τέτοια ψηφίσματα ανόητα, παράλογα, άχρηστα να βγαίνουν από το Κοινοβούλιο. Πάντα όμως θα μιλάνε ή για μετανάστες ή για ομοφιλόφιλους ή για φεμινιστές που φαίνεται να είναι καλύτεροι από τους απλούς πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια αρρώστια. Ώρα να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν νομίζω ότι χωρεί μεταρρύθμιση. Και απευθύνομαι και στι άλλες χώρε. Ας ακολουθήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο. Ας βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας προετοιμαστούμε γι' αυτό και ας χτίσουμε μια νέα Ευρώπη όπως την είχαν οραματιστεί οι ιδρυτές που δεν θα παρεμβαίνει στην οικογενειακή πολιτική, δεν θα προσπαθεί να αλλάξει το ρόλο της γυναίκας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς θα πρέπει να κάνει τη διαχείριση μιας σωστής νομοθεσίας, μιας καλής νομοθεσίας σε περιορισμένο βαθμό. Και ελπίζω πραγματικά και εγώ να ζήσω να το δω αυτό, αυτή τη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω πει δυστυχώ εξ αρχή ότι δεν δέχομαι μπλε κάρτα. Σόσνιε, ένα λεπτό έχετε, παρακαλώ. Ε, państwo, że ε, postaram się Wam coś Proszę Mam... Ευχαριστώ. Να επιχειρήσω, κυρίε και κύριοι, να σα εξηγήσω κάτι. Σα παρακαλώ, α εστιάσουμε τα πορίσματά σα ε, είναι λανθασμένα γιατί το σημείο εκκίνησης είναι λανθασμένο. Λέτε ότι οι γυναίκε έχουν ε, τα ίδια προσόντα, τι ίδιε ικανότητες με του άνδρες. Αυτό είναι εντελώ λάθο. Μετά διαμαρτύρεστε ότι δεν υπάρχει ίση εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια και σε θέσει λήψη αποφάσεων. Και θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία, ότι υπάρχει κάποια πατριαρχική συνωμοσία που εμποδίζει τι γυναίκε από την ανάληψη τέτοιων ευθυνών. Αλλά κοιτάξτε, Κοιτάξτε στην οικονομική δραστηριότητα. Αν οι γυναίκε δεν θέλουν να αναλάβουν τέτοιε ευθύνε, ή αν δεν θέλουν να απασχοληθούν καθόλου, είναι επειδή δεν έχουν ίσω τα προσόντα, ή επειδή δεν επιθυμούν μια τέτοια σταδιοδρομία. Ενώ, όπω ξέρετε, οι άνδρε ζουν λιγότερο από τι γυναίκε. Πώ θα του ε, ε, ανταμείψουμε για το γεγονό ότι πεθαίνουν ε, νεότεροι. Σα το λέει η αγορά οι γυναίκες δεν είναι σε αυτές τις θέσει και δεν υπάρχει καμία συνωμοσία ανδρών. Ακούσαμε όλες τις πολιτικές ομάδες. Τώρα, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση, οι ομιλητές, η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ πολύ, κύρια Επίτροπε. Ζούμε σε έναν κόσμο και σε μια κοινωνία όπου δεν είναι δυνατόν να αμφισβητείται η ισότητα ανδρών και γυναικών. Παρόλα αυτά, στα διοικητικά και υποπτικά συμβούλια δεν υπάρχουν επαρκεί γυναίκε. Οι γυναίκε είναι ο μισό πληθυσμό. Παρόλα αυτά, είναι πολύ λίγε σε αυτέ τι θέσει. Ιδιαίτερα για τι επιχειρήσει ε, που είναι τι εισηγμένε. Στην Τσεχία, για παράδειγμα, είναι μόνο 9%. Ενώ οι γυναίκε σίγουρα έχουν τα ίδια προσόντα τις ίδιες ικανότητες, αν όχι περισσότερες, γιατί οι γυναίκες έχουν υψηλότερο ποσοστό, υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και έχουν την ίδια φιλοδοξία. Παρά όλα αυτά δεν είναι επαρκής ο αριθμός των γυναικών σε αυτές τις θέσεις. Γιατί, γιατί οι γυναίκες είναι πολύ σημαντικές ως μητέρες και για να φροντίζουν ε, τους ηλικιωμένους. Οπότε ξεκινάνε αργότερα τη σταδιοδρομία τους. Δεν θα βοηθήσουν οι ποσοστώσεις να προωθήσουμε και να επιταχύνουμε την σταδιοδρομία των γυναικών. Πρέπει να βοηθήσουμε τι ίδιε τι γυναίκε να μπορούν να συνδυάζουν την επαγγελματική με οικογενειακή ζωή. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό είναι σημαντικό το Συμβούλιο επιτέλους να συμφωνήσει με αυτή την οδηγία. Ούτως ώστε επιτέλους να εφαρμοστεί, ούτως ώστε αυτή η οδηγία να βοηθήσει τον συνδυασμό της ε, επαγγελματική και οικογενειακή ζωής. Επιτέλους να γίνει, να εγκριθεί και να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Και σα ρωτώ, τι εμποδίζει τα κράτη-μέλη μέσω τη δικής τους ε, νομοθεσία να προωθήσουν την ισότητα των γυναικών. Για παράδειγμα, η Ισπανία. Πιστεύω ότι αυτό που έκανε η Ισπανική κυβέρνηση Μπορεί να το κάνει και σε εθνικό επίπεδο. Να αποφασίσει εγώ ω χώρα θα προωθήσω αυτά τα μέτρα που επιχειρώ να προωθήσω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όποιο θέλει μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Και φυσικά και η Ένωση μπορεί να δώσει καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ, Γκούτελεντ. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πάνω από το 65% των πτυχιούχων είναι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν τις γνώσεις για να καταλάβουν τις ε, κορυφαίες θέσεις στα ΔΣ. Και όμως ακόμα ε, δεν το κάνουν. Είναι απαράδεκτο. Δεν είναι μόνο άδικο, είναι και βλακώδες. Σημαίνει ότι χάνουμε γνώση. Δεν υπάρχει καινοτομία. Ε, βλέπουμε ότι σε πολλές εταιρείες οι γυναίκες είναι πολύ πιο καινοτόμες από τους άνδρες και οι εταιρείε που έχουν περισσότερες γυναίκες από άνδρες ε, παρέχουν πολύ καλύτερες δυνατότητες για τις εταιρείες αυτές. Παρόλα αυτά, πολλές εταιρείες και πολιτικοί εξακολουθούν ε, να μάχονται αυτήν την ιδέα ότι τουλάχιστον 40% των μη εκτελεστικών μελών θα πρέπει να είναι από το φύλλο που εκπροσωπείται. Γι' αυτό ακριβώς είναι περίεργο να βλέπουμε την Ισπανία να ε, μεταβάλει στάση στο Συμβούλιο. Δεν θέλουμε άλλα ωραία λόγια. Θέλουμε επιτέλους να γίνει κάτι στην πράξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά τις ε, γυναίκες στα Δέλτα Σίγμα, ας δούμε εδώ πέρα τι γίνεται σε Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν. Είχαμε 12 πρόεδρους ε, της Κομισιόν, ε, καμία γυναίκα. 30 πρόεδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μία γυναίκα και 78 πρόεδρους του Συμβουλίου, σε νέα γυναίκες. Λοιπόν, ε, γιατί δεν το βλέπουμε, γιατί δεν ζητάνε συγγνώμη οι άντρε ε, πρόεδροι για αυτό το γεγονό. Δηλαδή χρειάζεται πραγματικά οδηγία. Όλοι είναι ίσοι ε, ενώπιον του νόμου, στην πολιτική, στην οικονομία, στην κοινωνία. Έτσι τα έχουμε ρυθμίσει στο Σύνταγμα της Πολωνίας. Έχουμε μια κοινωνία στην οποία θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση, γιατί είμαστε όλοι ίσοι. Ε, ενώπιον του νόμου. Αυτή είναι η εντολή και πρέπει να την σεβόμαστε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπέτσερα Μπαστερετσέα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη στήριξή σας κύριε Επίτροπε και για την αποφασιστικότητά σας. Σήμερα ορισμένοι λένε ότι οι γυναίκες δεν είναι σε τέτοιες ηγετικέ θέσεις γιατί δεν το επιδιώκουν. Όμως το ποσοστό γυναικών των εισηγμένων ε, ευρωπαϊκών εταιριών από 10% το 2005 πέρασε στο 22% το 2015. Άρα κάτι γίνεται. Ορισμένοι λένε ότι δεν χρειάζεται εφόσον αλλάζει η κατάσταση πρωτοβουλία αυτή για την ίση εκπροσώπηση. Όμω οι γυναίκε ε, είναι επικεφαλής μόνο στο 7% των εισηγμένων και μόνο το 6% ε, στις κυριότερες επιχειρήσεις. Εξακολουθεί να υπάρχει η γυάλινη οροφή Υπάρχουν εμπόδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Για να γίνει αυτό πρέπει το Συμβούλιο να προωθήσει αυτήν την οδηγία. Η ίση εκπροσώπηση είναι θετική για όλους, για τις επιχειρήσεις, για τις γυναίκες. Οι επιχειρήσεις που έχουν γυναίκες έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Πρέπει να ε, καταλάβουμε ότι είναι το πιο λογικό να υπάρχει αυτή η ισότητα. Πρέπει να προχωρήσει αυτή η οδηγία, να αναλάβει την ε, προώθησε αυτέ τι ιδέε που απαιτούν οι Ευρωπαίοι και ελπίζω η Ρουμανία να παίξει το ρόλο τη. Κυρία Φορέντσα, για ένα λεπτό, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, των ε, Πρασίνων και των Σοσιαλιστών Δημοκρατών που κατέθεσαν αυτή την προφορική ερώτηση, τις προφορικές ερωτήσεις σε σχέση με την ενσωμάτωση της δεύτερης των φύλων ε, και με την συνσηγήτρια έχουμε εργαστεί προς την κατεύθυνση. Θα ήθελα να επισημάνω ωστόσο ότι εδώ αντιμετωπίζουμε, κοιτάμε να αντιμετωπίσουμε ένα σύμπτωμα αυτής της διακριτικής μεταχείρισης. Εδώ θα έπρεπε να προβλέψουμε και να προλάβουμε τις εξελίξεις αυτές που μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερες ακόμη διακρίσεις. Το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει λοιπόν απαντήσεις αποφασιστικές όχι μόνο για αυτή την ε, γυάλινη οροφή που αφορά τις γυναίκες και επιτρέπει μόνο στο 1% να την ξεπεράσουν σε όλες τις ε, διακρίσεις βάρος τους και εις βάρος ουδήποτε, είτε πρόκειται για φίλο, φιλή, ε, προέλευση κτλ. Πρέπει να καταπολεμείται κάθε διάκριση και πρέπει το Κοινοβούλιο να δώσει ένα έναυσμα σοβαρό προ την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ του συναδέλφου λοιπόν που κατέθεσαν τι προφορικέ ερωτήσει. Αλλά βλέπω ότι έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε και όπω υπενθύμησε και η κυρία Ορτασούν, θα μπορούσε, θα είχε, θα μπορούσε η περίοδο η βουλευτική αυτή να είχε κάνει πολύ περισσότερα ε, για τα θέματα τη ισότητας και τη απαγόρευσης των διακρίσεων. Η κυρία Αγιούτο για ένα λεπτό. Ε, το 2012, χρόνια πριν, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια πρώτη πρόταση για σχέδιο οδηγίας ε, για τις θέσεις των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων που έμεινε σε αδιέξοδο στο Συμβούλιο και στόχο είχε να εξασφαλίσει περισσότερη ισότητα στις, ε, στην παρουσία των γυναικών, ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Βέβαια ξέρουμε ότι αυτό, αυτή η ισότητα, ο στόχος ισότητας μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο όταν στο πεδίο τη δράση μπορούμε να αποδείξουμε την αξία μα, την αξία μα, που εμεί οι γυναίκε έχουμε και θέλω να διαβεβαιώσω τον συνάδελφο. Λυπούμε βέβαια για λογαριασμό του, αλλά είναι αποδεδειγμένο πως οι γυναίκες έχουν και περισσότερα πτυχία και δεξιότητες προς τους από του άντρες ε, και τα, το σημείο εκείνης αυτής της οδηγίας και των προτάσεων που είχε καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σχετικές διαπιστώσεις γιατί μόνο 13,20% κατέλαμβαναν στις υψηλές θέσεις γυναίκες και εδώ θέλω να ρωτήσω τη Ρωμανική Προεδρία τι είδους μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να ε, σπάσει αυτή τη γυάλινη οροφή επιτέλους και εάν σκοπεύει να καταστεί εκπρόσωπος της φωνής των γυναικών, εσείς κυρία Υφυπουργέ, εκπρόσωπος της φωνής των γυναικών στο Συμβούλιο. Ο κύριος Σκέλη, παρακαλώ ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι γνωστό ότι οι ή υπερπροσωπούνται στα ΔΣ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα το 2017 οι γυναίκε ήταν μόλι το 1 τέταρτο των μελών των ΔΣ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στην Ένωση. Το 2015 υπήρχαν περισσότεροι ε, Δέλτα ε, περισσότεροι, με συγχωρείτε, διευθύνοντες ε, σύμβουλοι που λεγόταν Τζον παρά γυναίκες. Λοιπόν, ε, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο τα ΔΣ. Από εκεί θα διαχυθεί σε ολόκληρη την ε, ιεραρχία. Ε, οι γυναίκες συχνά βρίσκονται σε άλλους ρόλους εντός των εταιριών, ενώ οι άντρες βρίσκονται σε θέσεις οι οποίες θεωρούνται πιο σοβαρές. Οι γυναίκες είναι στο ανθρώπινο δυναμικό, δημόσιες σχέσεις κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να αντικατοπτρίζονται ολόκληρε όλες οι απόψεις ε, που υπάρχουν στην κοινωνία. Αλλιώς ε, συνεχώς ε, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα ΔΣ θα προάγουν τους ομοίους τους. Δηλαδή αν υπάρχουν ήδη περισσότεροι άντρες θα προάγονται περισσότεροι άντρες. Αυτό δεν έχει νόημα. Σύμφωνα με το Διεθνές Ταμείο μια τέτοια πρακτική θα προωθούσε αυξημένη παραγωγικότητα και ισότητα στα εισοδήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κοφεράτη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συχνά στις συζητήσει μας ε, επενθυμίζουμε ότι η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά βέβαια στη συμπεριφορά, την πρακτική, έχουμε διαφορετικό προσανατολισμό, όπως ε, άλλωστε αποδεικνύει και η σημερινή συζήτηση. Αυτό που κάνει το Συμβούλιο είναι πονίδιστο πραγματικά, γιατί βρισκόμαστε ενώπιον μια οδηγία που έχει με ευρύτατη πλειοψηφία εγκριθεί πριν 10 χρόνια και περισσότερο και δεν έχει προχωρήσει ούτε βήμα το συμβόλιο. Εδώ δεν πρόκειται για κάτι το εξαιρετικά απαιτητικό ή ρηξικέλευθο αυτό που στάει η οδηγία. Ένα 40% για παρουσία των γυναικών, μια αντίστοιχη ποσόστοση για τις ε, θέσεις ε, της ε, ιεραρχίας παραμένει ανοιχτό το θέμα εξάλλου και της ισότιμη ε, αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και αυτό που ζητούσαμε εμείς ήταν ένα μικρό βήμα, ένα μικρό βήμα προς σωστή κατεύθυνση που θα επέδεικνυε μόνο απλώς καλές προθέσεις. Ελπίζω το Συμβούλιο να επιδείξει τη βούληση και να αποδείξει ότι σκοπεύει να το κάνει, να αλλάξει προς την ορθή κατεύθυνση, δηλαδή να δείξει σεβασμό και να ε, προωθήσει και την οδηγία αυτή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κούνεβα, ένα λεπτό σε μια κοινωνία χωρίς ισότητα αλήθεια τι αρμονία και τι ομορφιά μπορεί να επικρατήσει αναρωτιόταν ο Τζον Μίλτον. Το ίδιο αναρωτιέμαι και εγώ. Το γυάλινο ταβάνι που εμποδίζει την σταδιοδρομία χιλιάδων εργαζομένων γυναικών ανατρέπει τις ζωές τους. Εργαζόμενες με εμπειρία, σποντές και κατάρτιση αποκλέονται από διευθυντικές θέσεις αμείβονται λιγότερο τιμωρούνται αν έχουν ή αν θέλουν οικογένεια δέχονται παρενοχλήσεις διάφορων μορφών. Η πρόταση οδηγίας είναι σίγουρη, σίγουρα μια ακόμα ευκαιρία να διορθώσουμε ανισότητες που επικρατούν. Όμως, γιατί αργεί η υιοθέτησή της. Ρωτώ το Συμβούλιο ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο του η υάλινου ταβανιού στις επιχειρήσεις και πώς σκοπεύει να προάγει την ισότητα των φύλων κατά τη διάρκεια της Ρωμανικής Προεδρίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κούνεβα. Ο κύριος Ντουαχ δεν είναι εδώ και έτσι προχωρώ στη διαδικασία Catch Παρακαλώ με προσοχή στο χρόνο. Κινήσει ένα λεπτό. Έλα Κατερίνα. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε το 2017 ήταν ένα τέταρτο μόνο των μελών των, συμβουλίων, των διοικητικών συμβουλίων των εισηγμένων στα χρηματιστήρια ευρωπαϊκών επιχειρήσεων οι γυναίκες και όμως ακόμα τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ε, στα, στην εκπροσώπηση του στα διάφορα κράτη μέσα στην Ένωση. Οι ικανότητε βεβαίω των γυναικών είναι αμφισβήτητε και οι δεξιότητε του. Είναι απαράδεκτη λοιπόν αυτή η διάκριση ει βάρο του για λόγου στερεοτύπων, που ταυτόχρονα όμω ε, προξενεί προβλήματα και στην αγορά εργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσει μια καλύτερη ισότητα φύλων, εκπροσώπηση των φύλων η πιο ισόρροπη, χρειάζεται να εισαχθούν και νομοθετικά μέτρα. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Έστω και με ποσοστώσει υπέρ των γυναικών. Έγινε στην πατρίδα μου την Ιταλία, παραδείγμα την μια τέτοια πρωτοβουλία η οποία έφτασε να, ξεπερα... να εξασφαλίσει πάνω από το 33% των ε, γυναικών στου... στα διοικητικά συμβούλια και έτσι να, υπάρχουν πολύ καλύτερη... να υπάρχει πολύ καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών. Καλό λοιπόν τη Ρουμανική Προεδρία το ταχύτερο δυνατό να εξασφαλίσει πρόοδο για την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων επιχειρήσεων. Η κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό το συζητάμε εδώ και 7 χρόνια. Το είπαν όλοι οι συνάδελφοι. Εγώ θέλω να απευθώ κυρίως στους άνδρες που αναφέρθηκαν σε ανισότητες. Γιατί υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι δουλεύουν στο σπίτι και αισθάνονται μειονεκτικοί. Ε, κοιτάξτε, οι γυναίκες ε, και βιολογικά είναι παντού οι καλύτερες και στις ε, επιχειρήσεις και στο σπίτι γιατί περισσότερες έχουν ούτως ή δύο δουλειές και μια επαγγελματική δραστηριότητα και κάνουν τη δουλειά στο σπίτι και είναι οι καλύτερες για τα δικαιωτικά συμβούλια μπορούν να κάνουν δύο πράγματα την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν επαγγέλματα που είναι μόνο για άνδρες ή μόνο για γυναίκες και ελπίζω κυρία Υπουργέ και κυρία Επίτροπε να μπορέσουμε να υπερβούμε αυτή την ε, ε, μειοψηφία άρνηση κυρία στο Συμβούλιο. Λυπάμαι που πρέπει να υπάρχουν ε, ποσοστό, αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Αν η κοινωνία δεν καταλαβαίνει πώ πρέπει να προωθηθούν οι γυναίκε, πρέπει να παρέμβουμε. Συμφωνώ, κύριε Επίτροπε, η οδηγία για, την, για το συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και όλα τα άλλα που είπατε, όλες οι μελέτες το αποδεικνύουν, όλα αυτά πρέπει να γίνουν πραγματικότητα γιατί θα κερδίσει η κοινωνία. Ο κύριος Μαριάς για ένα λεπτό γυναικών και στην κοινωνία και στις ε, βασικές θέσεις και στην οικονομία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και προφανώς πρέπει αυτό να αλλάξει και φυσικά θα πρέπει οι γυναίκες να εκπροσωπηθούν και στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων αλλά η κοινωνική μηχανική το social engineering το οποίο επιχειρεί η ευρωπαϊκή ένωση δεν νομίζω ότι μπορεί να πετύχει στον τομέα αυτό ούτε μπορεί να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάνουν κάτι διαφορετικό. μπορεί όμως η ευρωπαϊκή ένωση να κάνει κάτι άλλο και επειδή είναι εδώ και ο κύριος Γιούγκερ και ακούω λέω το εξής 140 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 70 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 2,5 τρισεκατομμύρια έχει δώσει ο κύριος Ντράγκη λέω λοιπόν να μην γίνεται καμία χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια ούτε από δάνεια ούτε να αγοράζονται ομόλογα από την κεντρική τράπεζα εάν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν έχουν την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. να δείτε πώς αμέσως μόνες τους οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν και θα αλλάξουν την τακτική και θα έχουν την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια διότι δεν θα έχουν πρόσβαση ούτε στην οικονομία ούτε στα ομόλογα ούτε βεβαίως στα χρήματα που είναι και από το ε, πρόγραμμα juncker. με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια απάντηση και αναγκάζουμε τις επιχειρήσεις να έρθουν σε αυτά τα οποία εμείς επιθυμούμε. ευχαριστώ. Σας παρακαλώ να είμαστε όλοι αυστηροί με το χρόνο. Από εδώ και μπρος όποιος ξεπερνάει το λεπτό του θα ε, χάνει το μικρόφωνο. Σπίνα παρακαλώ. Πρόεδρε, ναι, αυτή η συζήτηση σήμερα νομίζω δείχνει μια μεγάλη σύγκληση του Κοινοβουλίου προς την υποστήριξη της ε, οδηγίας αυτής και σας παρακαλώ προσέξτε το δεν λέει τίποτε το καταπληκτικό ένα μικρό βήμα που όμως πάει προς σωστή κατεύθυνση γιατί δεν επιβάλλει την παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εδώ αυτή η οδηγία. Απλώς καταγράφεται πως δεν είναι δυνατόν να εκπροσωπείται μόνο το 50% δηλαδή ο ανδρικός κόσμος στη διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων των εισηγμένων και ότι χρειάζεται και η εκπροσώπηση των γυναικών. Μια πραγματικότητα. Το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι όπως πάντα το Συμβούλιο και το λέω αυτό με μεγάλη πικρία αλλά και μεγάλη ανησυχία διότι βλέπουμε εκεί μια στάση Έχουμε από τη μία πλευρά μια στάση του Κοινοβουλίου που θέλει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάποια βήματα προόδου. Ενώ από την άλλη έχουμε τη συμπεριφορά και στάση του Συμβουλίου και, που το οποίο δυστυχώς πολύ συχνά Πρόεδρε παρεμποδίζει αποφάσεις και επιλογές που βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως και η προτεραιότητα πρέπει να είναι αυτή η ισότητα και χρειάζεται δράση. Ευχαριστώ πολύ. Μάη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για αυτήν την οδηγία και για την συζήτηση για διάφορους λόγους. Είναι καλό το ότι συμμετέχουν όλο και περισσότεροι άντρες γιατί πρέπει από κοινού να επιτύχουμε την ισότητα για τις γυναίκες και την εκπροσώπησή τους σε όλους τους τομείς γιατί είναι αρκετά καλές όσο και οι άντρες και αναφέρθηκε το μισθολογικό χάσμα ξέρω ότι στη Γερμανία είναι υψηλότερο από σε άλλες ε, χώρες συζητάμε ήδη σε μας ένα νόμο περί ισότητας με διαφορετικές προσεγγίσεις. Κάποια έχουν τέτοιους ε, νόμους για το φύλλο που υποεκπροσωπείται. Είναι κρίμα το ότι το συζητάμε ακόμα. Έπρεπε να υπάρχει ήδη. Και χαίρομαι που η συναρφός Ρέγνερ λέει ότι είναι επιτέλους το ευρωπαϊκό DNA. Γι' αυτό ελπίζω να υπάρχει ευρεία ε, στήριξη και να καταλήξουμε κάποτε σε ένα αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ η κυρία Ward για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Είναι εκπληκτικό να βλέπουμε πως ε, η πρωτοβουλία αυτή για την ισότητα μπλοκάρει στο Συμβούλιο μετά από πέντε χρόνια. Πραγματικά δείχνει πόσο συντηρητικές είναι οι κυβερνήσεις των ε, κρατών μελών. Είναι ανισχυτικό το ότι είναι τόσο αμφιλεγόμενη αυτή η πρωτοβουλία. Και βλέπουμε ότι βεβαίως η ισότητα, αν και είναι σημαντική κυρίως, απευθύνεται σε προνομιούχες γυναίκες και δεν ασχολούμαστε με τις μη προνομιούχες. Στον κόσμο των επιχειρήσεων οι γυναίκες υφίστανται πολλές διακρίσεις, αντιμετωπίζουν φοβερές προκλήσεις, μαύρες, Ρωμά, μετανάστες, ανάπηρες, ε, ξεχνιούνται και στην πολιτική και στις επιχειρήσεις μετά από την συμφωνία που επετέφθη την προηγούμενη εβδομάδα στην οδηγία για την ισορροπία οικογενειακής ε, και επαγγελματικής ζωής ζητάω από την Προεδρία να επιτύχει επιτέλους μια συνένεση για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Μιράντα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση εδώ που επικρατεί στο Συμβούλιο νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική. Αρκεί να δούμε μια φωτογραφία του Συμβουλίου. Λίγες οι γυναίκες στο διοικητικό, στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων της Ευρώπης. Στην ε, Σουηδία το πολύ να φτάσουν στο 36%. Όμως είναι πολύ μακριά τα ποσοστά αυτά από τα επίπεδα που ζητεί η οδηγία. Έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, σε προηγούμενη σύνθεση του Κοινοβουλίου, το ίδιο θέμα. Και δυστυχώ βλέπουμε ότι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση πάντα και δεν γίνονται σεβαστέ οι οδηγίε. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία παρέμβαση. Dear President, dear Commission... Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, εγώ ως ε, ε, Ευρωβουλευτή από την Ρουμανία, καλωσορίζω το γεγονό ότι αυτή η οδηγία είναι μία από τι προτεραιότητε τη Προεδρία μου για την ισότητα των φύλων. Σε κάποια κράτη-μέλη άλλαξε η κατάσταση πρόσφατα και ε, έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι θα προχωρήσει η διαπραγμάτευση για το θέμα αυτό. Ο λόγος υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικέ θέσεις ε, είναι περίπλοκος. Υπάρχει βεβαίως ε, η νοοτροπία που υπάρχει και σε διοικητικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Η Γιάννη οροφή στην οτροπία των επιχειρήσεων όχι μόνο υποτιμά την συμβολή των γυναικών στη δίκη των επιχειρήσεων, αλλά αποθαρρύνει και τι γυναίκε από την προσπάθεια να προωθήσουν τη σταδιοδρομία του και να αναπτύξουν τι δυνατότητέ του στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Η δική μου εμπειρία μου επιτρέπει να σα πω ότι οι γυναίκε όταν αναλαμβάνουν την ηγεσία κάποιων επιχειρήσεων προσθέτουν αξία και αυξάνεται η επιχείρηση, κάνει καλύτερε προτεραιότητε για, για τι ανάγκε των γυναικών και αλλάζει την οτροπία τη επιχείρηση. Εκφράζω λοιπόν τη στήριξή μου για τι προσπάθειε Ρουμανική Προεδρία ούτω ώστε να συνεχιστεί η συζήτηση για αυτή την οδηγία. Σα ευχαριστώ πολύ. Ωραία, έκλεισε η συζήτηση. Για να απαντήσει τώρα η κυρία Γιούροβα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την αποφασιστικότητα και την στήριξη του Ευρωπαϊκού του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, όπως φάνηκε στην συζήτηση και χαιρόμαι που υπάρχει και ενδιαφέρον των ΜΜΕ. Θα ήθελα να καταλήξω λέγοντας ε, λίγα λόγια. Πέρα από την σαφή στήριξη της Κομισιόν που ήδη εξέφρασα, θα ήθελα να σας πω πως ε, δεν ε, περιμένουμε να ξεμπλοκαριστεί το θέμα αυτό στο Συμβούλιο, γιατί υπάρχει πολλή δουλειά που μπορεί να γίνει για να στηρίξουμε την ε, μεγαλύτερη ισότητα ε, όχι μόνο στον κόσμο των επιχειρήσεων. Θα ήθελα και πάλι να αναφέρω κάποια στατιστικά στοιχεία. Οι γυναίκες είναι πάνω από το 50%. 62% των πτυχιούχων. Οπότε θα έλεγε κανείς πως ε, το φυσιολογικό θα ήταν να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση των γυναικών σε διάφορους τομείς. Ας συγκρίνουμε τους αριθμούς όμως. Έχουμε 22% γυναικών στα ΔΣ. Μόλις 6% των ε, διευθύνων των συμβούλων. 20% γυναικών βουλευτών. Έχουμε κάποιες ε, κυβερνήσεις ε, στα κράτη-μέλη με μία ή δύο γυναίκες. Πρόσφατα είχαμε κυβέρνηση χωρίς γυναίκα. Ας δούμε τώρα τα θετικά παραδείγματα. Στην ε, Κομισιόν ήδη φτάνουμε το 40% στις θέσεις τις διευθυντικές. Μια πολύ έξυπνη διαδικασία η οποία εγγυάται τον ε, δίκαιο ανταγωνισμό χωρίς ε, προκαταλήψεις ε, που βλέπουμε αλλού και χωρίς εμπόδια. Και να αντιδράσω σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ζόλταξ. Ε, πίστεψε με, ε, ως γυναίκα εντός κομψιών. δεν χρειάστηκε να γίνω άντρα για να φτάσω σε αυτήν την θέση και να συνεισφέρω στην λήψη των αποφάσεων. νομίζω πως... Κατά σύμπτωση είναι εδώ και ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, αλλά ε, υπάρχουν τουλάχιστον 9 γυναίκες στην Κομισιόν και όλοι οι συνάδελφοι νομίζω κάνουν ε, πολύ σωστή δουλειά με το να μεταφέρουν την οπτική των ε, γυναικών στην λήψη των αποφάσεων. Όταν συγκρίνουμε αυτούς τους αριθμούς λοιπόν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Γι' αυτό ακριβώς ε, εργαζόμαστε σκληρά για να το αλλάξουμε. Και δεν ε, περιμένουμε μόνο... Δεν ξεμπλοκάρουμε μόνο αυτή την οδηγία. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω κυρία Πάρκερ να διαβάσετε την ε, τωρινή εκδοχή της οδηγίας. Τίποτα δεν λέει ότι το μόνο προσόν είναι να είναι κανείς γυναίκα. Ζητάμε απλά δίκαιο ανταγωνισμό και συνεργασία. Καλό είναι να ε, δείτε την ε, τελευταία έκδοση την οποία προωθούμε. Αυτή τη στιγμή ήδη τα μισά κρατημέλη έχουν σχετική νομοθεσία, οπότε προσεχώς θα έχουμε και τα υπόλοιπα. Και γεγονός είναι ότι τα κρατημέλη μπορούν να δράσουν από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να περιμένουν να ξεμπλοκάρει η οδηγία γιατί από αυτά εξαρτάται να κινηθούν. Εν τω μεταξύ η Κομισιόν δεν περιμένει κάνουμε και μη νομοθετικό έργο στηρίζουμε την ε, χάρτα της ποικιλομορφία, ε, την οποία έχουν συνυπογράψει 10.000 ε, μεταξύ των οποίων μεγάλες εταιρείες η Sodexo, IBM, Siemens πολυεθνικές που προωθούν την ιδέα αυτή η οποία είναι υποφελής ε, για τις επιχειρήσεις ε, πολλά κρατημέλη ε, και όπου δεν υπάρχει νομοθεσία εξάγουν και διαδίδουν αυτό το θετικό μήνυμα. Χρηματοδοτούμε και πολλά έργα τα οποία προωθούν ακριβώς την ποικιλομορφία. Είναι λοιπόν ένα σχέδιο Β αν θέλετε να μην ε, περιμένουμε την νομοθεσία κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα αλλά θα ήθελα να επαναλάβω πώς ε, θεωρούμε πώς ε, θα εγκριθεί τελικά αυτό το νομοθέτημα και πάλι θα ήθελα να επαναλάβω ότι ελπίζουμε ότι η Ρουμανική Προεδρία θα κάνει πολύ καλή δουλειά σας ευχαριστώ η κυρία Τσότ για το Συμβουλίο Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε κυρίες και κύριοι βουλευτές κυρίες και κύριοι. ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Όπως είπα και στις αγωγικές μου παρατηρήσεις η προσήλωση του Συμβουλίου στην ισότητα των φίλων, είναι πραγματική και απαρασάλευτη. Η Προεδρία της Ρουμανίας οργανώνει διμερείς συνομιλίες με την ανασχετική μειοψηφία για να αναζητήσει δυνατότητες λύσης. Έχουμε σχεδιάσει ακόμη ε, συνεδριάσεις σε επίπεδο ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό. Δεν πρέπει όμω και να λησμονούμε ότι η Προεδρία είναι στα χέρια και υπό τον έλεγχο των κρατών μελών. Απαιτείται λοιπόν μια ειδική πλειοψηφία για την πρόθεση αυτού του έργου. Ε, επιπλέον των όσων έχουμε κάνει σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο για να προαγάγουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πάντως, όπως είπα και νωρίτερα, προετοιμάζουμε και μια σειρά συμπερασμάτων για την ε, διαφορά στις αμοιβέ μεταξύ ανδρών και γυναικών και τις πολιτικές ε, συγκερασμού του οικογενειακού και του επαγγελματικού βίου. Ελπίζουμε ότι αυτά τα συμπεράσματα θα εγκριθούν στο Συμβούλιο Άψικο στις 13 Ιουνίου και θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι η Ρουμανική Προεδρία ε, θα υποδεχθεί στο Βουκουρέστι το Φεβρουάριο την ε, ομάδα εργασίας για την ε, ισότιμη εκπροσώπηση, για την ενσωμάτωση σα του φίλου καλύτερα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε και τους υπουργούς, ε, τους αρμόδιους άψκο στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα σήμερα εδώ. Με την κοινή δουλειά τους το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να θέσουν ένα τέρμα στην, στις διακρίσεις και την αδικία και να εξασφαλίσουν ε, ως πραγματικότητα για όλες τις γυναίκες και τους άντρες την ισότιμη μεταχείριση σε μια περίοδο μετάβασης, σε μια περίοδο κλειδονισμών όπου αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις. Το μέλλον όμως είναι η ισότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την κυρία Σότ και τώρα ολοκληρώνεται έτσι η κοινή συζήτηση. Δε ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Φινλανδίας για το μέλλον της Ευρώπη Κάνουμε μια διακοπή ενός λεπτού. Καταρχά, θέλω να ευχαριστώ τον Φιλανδό, τον Φιλανδό Πρωθυπουργό που είναι εδώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τι ε, διαφορέ θέσει των, των διάφορων χωρών ε, για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισημάνει δύο-τρία περισσότερα σημαντικά θέματα και θέλουμε περισσότερε εξουσίε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Θέλουμε να ενισχύσουμε και όχι να καταστρέψουμε την Ευρώπη. Στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θέλουμε την αλλαγή από το 1,1 στο 1,3 του όγκου του. Έχουμε επίσης ε, προτίμηση για τους ιδίους πόρους. Ε, μετανάστευση είναι πολύ σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη μεταρρύθμιση των κανόνων του Δουβλίνου και θέλουμε να δούμε απόφαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εχθές και σήμερα στο επίκεντρο των συνομιλιών μας μάλιστα έθεσαμε δύο κέρια ζητήματα, το Brexit και τη Βενεζουέλα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για μα να ενημερωθούμε για τι ιδέε σα για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ποιε είναι οι θέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε ποιε είναι οι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίω, τα κράτη-μέλη έχουν το καθένα τι δικέ του θέσει και τώρα είναι σημαντικό να ακούσουμε ποιε είναι οι θέσει τη Φιλανδία. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να δώσετε τώρα τις, ε, τον εκδηλώσετε τον ενδιαφέρον σας για το Catch the αμέσως μετά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού θα κλείσουμε τον κατάλογο των αγορητών. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σας φέρνω τους χαιρετισμού από την πολύ κρύα Φιλανδία. Ήμουν στη Βόρεια Φιλανδία την προηγούμενη εβδομάδα, εκεί μένω. Η θερμοκρασία ήταν μείον 30 και είχαμε ένα μέτρο περίπου χιόνι. Έχουμε βαρύ χειμώνα. Ε, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι και εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στα πλαίσια των ε, πολύ δύσκολων ε, καταστάσεων. Οι συζητήσει για το μέλλον της Ένωσης είναι ουσιώδης για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, για να εκπληρώσουμε το όραμα της διακήρυξης της Ρώμης, πρέπει να συζητήσουμε πώς θα επιτύχουμε επαρκή ενότητα για να λαμβάνονται αποφάσεις και να εφαρμόζονται. Δεύτερον, Πρέπει να συζητήσουμε για να διαπιστώσουμε τις ε, προτεραιότητες των ΜΕΝ και των ΔΕ για τη δράση και τον προπολογισμό της Ένωσης. Οι χώρες της Ένωσης είναι κάτι που γνώρισα όταν ήμουν επιχειρηματίας. Είχαμε θηγατρικέ σε διάφορες χώρες τη Ευρώπης. Όταν ήμουν 30 και κάτι, θυμάμαι ότι ταξίδευα για να συναντήσω τον επικεφαλή μια μεγάλη ε, γαλλική εταιρεία. Στο αεροπλάνο διάβασα έναν ταξιδιωτικό οδηγό που, είχε, που δανειστεί η γυναίκα μου από, ένα, από μια βιβλιοθήκη. Έλεγε ότι δεν θα πρέπει ποτέ να κάνεις ερωτήσεις για την οικογένεια όταν ε, ε συναντάς ένα Γάλλο για επαγγελματικού λόγους. Όταν έφτασα στην ε, συνεδρίαση, ε, στην, συγγνώμη, στο δείπνο, ο επικεφαλής ήταν με τη γυναίκα και την κόρη του και η πρώτη ερώτηση που με έκανε ήταν «Πες μου για την οικογένειά σου». Τότε κατάλαβα ότι εμείς οι Ευρωπαίοι Έχουμε πολλά κοινά και μπορούμε να συνοηθούμε. Έχουμε περισσότερα κοινά από όσα νομίζουμε. Ήδη το 1920 ο ιδεολογικό πρόδρομο και ιδρυτής ε, του κεντρικού του κέντρου τη της Φινλανδίας, ο Σάντρι Άλκιο, έγραψε ότι για να υπάρξει ειρήνη στην Ευρώπη, η Ήπειρος θα πρέπει να οδηγηθεί προ τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη. Ανέφερε ακόμη και ένα κοινωνόμισμα. Ήταν πρωτεργάτης από πολλές ε, απόψεις. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, η διεθνή συνεργασία και η προώθηση της ειρήνης και της οικονομικής ανάπτυξης έχει υπάρξει φάρος για τη Φιλανδία. Αγαπητοί φίλοι, τα τελευταία χρόνια όμως ε, είδαμε πολύ λαϊκισμό στην Ευρώπη. Είδαμε τι συμβαίνει όταν, και που οδηγεί ο λαϊκισμός όταν προτείνονται υπεραπλουστευμένες λύσεις για περίπλοκα θέματα. Στο τέλος κάνει δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Αυτό συνέβη και στον Ηνωμένο Βασίλειο και τα αποτελέσματα είναι ενώπιον όλων μας. Αλλά δεν είναι μόνο το Brexit όπου βλέπουμε τα αποτελέσματα του λαϊκισμού. Βλέπουμε ότι μειώνεται το κράτος δικαίου, η ελευθερία των μέσων και τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτά δεν θα τα περιμέναμε. στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει τις κοινέ αξίες της μέσω της εξωτερικής της πολιτικής αν δεν μπορεί να τις προωθήσει στο εσωτερικό της. Οι κοινέ αξίες όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, ασφάλειας και ευημερίας της Υπήρου μας. Αυτές οι αξίες πρέπει να ε, συνενώνουν τα κράτη-μέλη. Πρέπει να γεφυρώσουμε τις ε, εσωτερικές διαιρέσεις της Ευρώπης. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει κανένας συμβασμός στην εφαρμογή του κράτους δικαίου. Η Φιλανδία καλωσορίζει θερμά τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σύνδεση του πολιτού ε, δημοσιονομικού πλαισίου με το κράτο δικαίου. Είμαι πεπισμένο ότι υπάρχει τρόπο να δημιουργηθεί ένας ε, ισορροπημένος μηχανισμός για να εφαρμοστεί αυτή η αρχή. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ο πιο σημαντικό ακρογωνιαίο λήθο που καθορίζει τη θέση τη Φιλανδία όσον αφορά την εξέλιξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νομισματική Ένωση είναι ο σεβασμό των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί και να υπάρξει ε, αποτελεσματική εφαρμογή τους. Στηρίζουμε ισχυρά μια Ευρώπη που επιτυγχάνει αξιοπιστία μέσω συγκεκριμένη δράση. Το 2015 η κυβέρνησή μου ανέλαβε ενώ είχαμε ένα δημόσιο έλλειμμα περίπου 3,5% σε σχέση με το ΑΕΠ. Το κατεβάσαμε στο 2% μέσω ε, εποδίνων εξοικονομήσεων σε σχέση με το ΑΕΠ πάντα το 2%. Βελτιώσαμε τα δημοσιονομικά μέσω μεταρρύθμισης ε, των συντάξεων και της ε, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και άλλων κοινωνικών μέτρων. Η εσωτερική υποτίμηση το 4% έγινε μέσω προώθησης της ε, απασχόλησης και της ανάπτυξης. Συμφωνήσαμε με τα συνδικάτα για πάγωμα των μισθών και για περικοπές. Επεκτείναμε κατά 24 ώρες τον ετήσιο χρόνο εργασίας και μειώσαμε τις εισφορές των εργοδοτών στην κοινωνική πρόνοια. Αυτέ είναι μόνο ε, κάποιε από τι πρωτοβουλίε μα. Μπορείτε να καταλάβετε, αυτέ μα οι ενέργειε δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλεί. Ωστόσο, τώρα, μετά από τρία χρόνια, δεν έχουμε πλέον δημόσιο έλλειμμα. Ο προπολογισμό είναι ισοσκελισμένο και η απασχόλησή μα είναι η υψηλότερη εδώ και 30 χρόνια. Οπότε, η ιδέα ότι πρέπει να λύνονται αυτά τα προβλήματα μέσω μονίμων δημοσιονομικών μεταφορών είναι απαράδεκτη για μας. Η καλύτερη εγγύηση κατά των ε, οικονομικών σοκ είναι ισοσκελισμένοι προπολογισμοί και χαμηλό χρέος. Πολλές φορές τα χρόνια αυτά θυμάμαι αυτό που είπε ο Ζωάν Κλοντ Ιούνκερ. Όλοι ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς να επανεκλεγούμε ε, αφού θα το έχουμε κάνει. Εγώ ε, θα ελέγξω στην πράξη αυτό στις ε, περχόμενες εκλογές τον Απρίλιο. Για να δούμε. Τι εννοώ. Παρά τον κίνδυνο, τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν και να εφαρμόζουν αποφάσεις. Η αποτελεσματική εφαρμογή είναι η μακράν καλύτερη μέθοδος για να αποκριθούμε στις ε, σημερινές και μελλοντικέ προκλήσεις. Θέλουμε εφαρμογή της ενιαίας αγοράς και πολιτικών για την έρευνα, ανάπτυξη και την καινοτομία. Θέλουμε εφαρμογή των ε, πολιτικών εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Θέλουμε εφαρμογή των μεταναστευτικών πολιτικών και εφαρμογή των πολιτικών για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Η καλύτερη εφαρμογή είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή λαϊκισμού και για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κύριοι, η Φιλανδία θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμεινο του έτους. Θα αναφέρω λοιπόν κάποια σημεία που θα μας απασχολήσουν στην Προεδρία μας. Είναι επίσης ε, θέματα στα οποία θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί στενότερα και να κάνει και τα όσα λέει. Θα ξεκινήσω από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το βασικό εργαλείο εφαρμογής της πολιτικής. Κατά την άποψη της ε, Φιλανδίας, το συνολικό επίπεδο του ΠΔΠ πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τωρινό ποσοστό. Πρέπει να εστιάσουμε στους τομείς όπου έχει τις καλύτερες δυνατότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετανάστευση, ασφάλεια, ενιαία αγορά, καινοτομία, ψηφιοποίηση και κλίμα. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανάγκη να υπάρξει μια ανακατανομή των κονδυλίων της αγροτικής ανάπτυξης εντό του προπολογισμού. Η κοινή αγροτική πολιτική μας δίνει την δυνατότητα να δώσουμε ασφαλή και προσιτά τρόφιμα στους πολίτες και να μπορούν βεβαίως να ζήσουν από τη δουλειά τους και οι αγρότες. Ταυτόχρονα η πολιτική συνοχής δημιουργεί πιο ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ κρατών και εντός των κρατών Είμαι πεπισμένος ότι θα καταφέρουμε να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των παραδοσιακών πολιτικών της Ένωσης και των νέων προκλήσεων. Είμαι επίσης πεπισμένος ότι μπορεί αυτό να γίνει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Φιλανδίας. Δεύτερον, χρειάζεται μια μεταναστευτική πολιτική με μια συνολική προσέγγιση. Πρώτα, οι αιτίε της μετανάστευσης που πρέπει να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά. Πέρα από την αναπτυξιακή συνεργασία και ανθρωπιστική βοήθεια απαιτούνται το εμπόριο και οι επενδύσεις για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να γίνει πιο αποτελεσματική πολιτική των επιστροφών. Η εσωτερική πτυχή της μετανάστευσης είναι στα χέρια μας. Πρέπει να διαχειριστούμε την ε, μετανάστευση μέσω άμεσων μετεγκαταστάσεων από τα στρατόπεδα προσφύγων. Αυτό θα σημάνει μικρότερη πίεση στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και λιγότερη λαθρέα διακίνηση. Ταυτόχρονα, η διαχείριση των εξωτερικών σύνορων μας θα πρέπει να ενισχυθεί. Επίσης, υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε με τα πιο πολύπλοκα πολιτικά ζητήματα, όπως ένας μηχανισμός αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια των κρίσεων πρέπει να το συμφωνήσουμε αυτό εκ των προτέρων και όχι εν το μέσο μιας κρίσης όπως κάναμε το 2015. Τρίτον, η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια που είναι επίσης σημαντική και πρέπει να ενταθεί. Η Φιλανδία ζητά ενεργά μια φιλόδοξη πρόοδο σε ζητήματα Ασφάλεια και Άμυνας μαζί με τη Γαλλία. Είναι καλοδεχούμενη λοιπόν αυτή η πρόοδο. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου και της ε, ΠΕΣΚΟ επίση είναι βήματα προ σωστή κατεύθυνση. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ε, εφαρμογή και στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει ενισχύσει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει υβριδικές απειλές. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπισης Υβριδικών Απειλών στο Ελσίνκι συνεισφέρει στην ετοιμότητα των χωρών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις 19 ε, χώρες που συμμετέχουν, 16 από τις οποίες είναι κράτη-μέλη της Ένωσης, για την ε, προσήλωσή τους ε, σε αυτό. Επίσης, καλώς ορίζω και τα υπόλοιπα κρατημέλη αν θέλουν να ενταχθούν. Τέταρτον, πρέπει να βελτιωθεί η ενιαία αγορά. Είμαστε η καλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο. Πέρα από τις καινοτομίε και το εμπόριο, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος δημιουργίας θέσεων εργασίας. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, ειδικά στις υπηρεσίες και τα ψηφιακά προϊόντα. Η βελτίωση της κατάστασης εξαρτάται από εμάς. Σας ε, ζητώ λοιπόν να καταλήξετε σε μια κοινή αντίληψη για να περάσουν οι 35 προτάσεις που είναι ακόμα αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Κοιτώντας προς το μέλλον, ελπίζω η νέα Κομισιόν να έχει μια πιο γενική προσέγγιση όπου θα συνδέονται καλύτερα η ενιαία αγορά, η ψηφιοποίηση, η βιομηχανική πολιτική και η ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ανάπτυξη που θα κοιτάει προς το μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κινητικότητα δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη και άλλα. Επίσης, πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα εφαρμόζοντας τις αρχές του κοινωνικού πυλώνα Παραδείγματο χάρη έχει μεγάλη σημασία να προωθηθεί η ισότητα στον χώρο εργασία και να ενισχυθεί το επίπεδο εκπαίδευση όλων των πολιτών. Πέμπτον, η εμπορική πολιτική έχει μεγάλη σημασία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νέες θέσεις εργασίας. Όσον αφορά τις συμφωνίες ελευθέριου εμπορίου, Είμαι ικανοποιημένο από τα τελευταία επιτεύγματα που είχαμε, τη σύναψη συμφωνιών με Ιαπωνία, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, Μεξικό και Καναδά. Και εύχομαι να ολοκληρωθούν ε, σύντομα οι διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται. Όμως, είναι επιβλαβές εάν οι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν να υψώνουν εμπορικά τείχη, τα οποία πρέπει να ρίξουμε ειδικά από την σκοπιά των μικρότερων χωρών ε, η ζημιά μπορεί να είναι μοιραία. Πρέπει να σεβόμαστε τους κοινούς κανόνες του εμπορίου. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή. Η έκθεση του Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή μας υπενθύμησε και πάλι πως ε, πλέον απειλείται η ζωή στη γη. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα συμπεράσματα της επιστήμης. Ε, πέρα από τις απειλές βλέπω πάρα πολλές ευκαιρίες. Ως μηχανικός σκέφτομαι και προσανατολίζομαι προς λύσεις και προς την τεχνολογία. Είμαι σίγουρος πως ε, καθώς ο κόσμος προχωρά προς ανάπτυξη με χαμηλό άνθρακα θα είμαστε στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, φιλόδοξης κλιματικής πολιτικής και έτσι θα έχουμε και νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Πρέπει να ληφθούν μέτρα σε τρία μέτωπα. Εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα και ε, απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακα και νέες τεχνολογίες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ε, σκανδιναβική συνάντηση για το κλίμα στο Ελσίνκι. Και οι σκανδιναβικές χώρες υποσχέθηκαν να αυξήσουν το επίπεδο φιλοδοξίας μέχρι το 2020. Θέλουμε να παίξουμε έναν καταλητικό ρόλο για να περιοριστεί η παγκόσμια θέρμανση στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Επίσης, κατά τη διάρκεια συζητήσεων στο Κοινοβούλιο της Φιλανδίας, 8 κόμματα της χώρας έθεσαν τον στόχο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς τον άνθρακα πριν το 2050. Αυτό απαιτεί αυστηροποίηση των υποχρεώσεων ε, που έχουμε για το 2030 στο 55% τουλάχιστον του επίπεδου του 1990. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εκπομπών είναι το πιο οικονομικό και αποτελεσματικό σύστημα για την ε, μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα έχει δημιουργήσει το σύστημα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να καθοδηγεί τους ε, παραγωγούς προς τη μείωση των ε, εκπομπών κατά τρόπο αποτελεσματικό. Έχουμε προτείνει, έχουμε πει ότι νέοι τομείς, ε, η ψήξη και η θέρμανση δηλαδή των κτηρίων πρέπει να περιληφθούν στο σύστημα ITS, το σύστημα των ανταλλαγών. Επίσης, ε, πρέπει να επιταχύνουμε τη μετάβαση προς μια κυκλική και βιοοικονομική δραστηριότητα. Ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα δράση για τη βιοοικονομία πρέπει άνευ καθυστερήσεως να υλοποιηθεί. Μια μικρή λεπτομέρεια. Η κυβέρνησή μου αποφάσισε να μην ε, ετοιμάσει δωράκια της Προεδρίας, αλλά να κάνει τη σχετική εξοικονόμηση από τους ε, πόρους σε άνθρακα που θα προξενούσαν τα ταξίδια τα αεροπορικά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Επίσης, πρέπει να μιλήσουμε για τις δεξαμενές άνθρακα. Καταβόθρες άνθρακα. Έχουμε 4 εκατομμύρια εκτάρια δασών και 5 ε, δισεκατομμύρια εκτάρια δασών και 5 δισεκατομμύρια ε, εκτάρια ε, καλλιεργήσιμης γης. Με ξαφνιάζει λοιπόν το πόσο πολλοί άνθρακα θα μπορούσαμε να συγκρατήσουμε από τα χωράφια εάν κάναμε αλλαγέ στον τρόπο με τον οποίο τα καλλιεργούμε 100 γεωργοί άνθρακα, ανθρακογεωργοί θα μπορούσαμε να τους πούμε, μπορούν να δοκιμάσουν τώρα τις νέες αυτές πρακτικές στη γεωργία και μπορούμε να, το, να κάνουμε αντίστοιχους σχεδιασμούς και για τα δάση. Μόνο η Αφρική ε, χάνει 2 εκατομμύρια εκτάρια δασών κάθε χρόνο, όσο είναι δηλαδή ολόκληρη η έκταση της Σλοβενίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων μας λέει στην έκθεση για, τα παγκόσμια, για την κατάσταση των δασών στον κόσμο ότι πρέπει να ε, εστιαστούμε περισσότερο στα δάση αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Ένα συγκεκριμένο βήμα θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την εξωτερική χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση των συνολικών ε, καταβοθρών ε, ή δεξαμενών άνθρακα. Έχει προτείνει λοιπόν ένα, ένα ευρωπαϊκό ε, ταμείο για τα δάση της Αφρικής η Φινλανδία με αντίστοιχες επενδύσεις που θα είχαν σημαντικές σημαντικό αντίκτυπο για, για το κλίμα αλλά και για τις γεωργικές θέσεις εργασίας. Ε, πιστεύουμε λοιπόν ότι έχουμε το τεχνικό δυναμικό για να συγκρατούμε περισσότερο άξα, άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα και να το μετατρέπουμε σε άλλα προϊόντα. Έχουμε τεράστιο δυναμικό έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομία στον τομέα αυτό. Επίσης πρέπει να στραφούμε με καινοτόμους τρόπους για να αναζητήσουμε νέες, ε, νέα κίνητρα και νέες μεθόδους με εφαρμογές στην αγορά που θα εξασφαλίσουν την αύξηση των δεξαμένων άνθρακα. Το κύριο μήνυμα που θέλω να απευθύνω είναι ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα και πρέπει να τα κάνουμε ταχύτερα. Πρέπει να μειώσουμε εκπομπέ, πρέπει να ενισχύσουμε τι ε, καταπόθρε άνθρακα και να υιοθετήσουμε νέε τεχνολογίε για τη συγκράτηση του οξυδίου του άνθρακα από τον ατμοσφαιρικό αέρα ή, ίσω και αμέσω από, την από την πηγή τη εκπομπή. Αγαπητοί Ευρωπαίοι συμπατριώτε, Αμέσως μετά τις ε, ευρωεκλογέ θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταλήξει συμφωνία για το φιλόδοξο και πλήρες ε, σχέδιο που ονομάζεται ε, θεματολόγιο για τη στρατηγική. Πέραν των θεμάτων του κλίματος θα πρέπει να σταθούμε και στην ανάπτυξη και την ασφάλεια. Βεβαίως και τα θέματα του κράτους δικαίου παραμένουν κρίσιμη σημασία. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν και απευθύνω μία έκκληση για πιο συγκεκριμένες δράσεις ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση με ουσιαστική υλοποίηση του δικαίου και με περισσότερες ευθύνες. Ευθύνες που σημαίνει και εγώ αναλαμβάνω ευθύνη για τον εαυτό μου, αλλά αναλαμβάνω ευθύνη και για τους γύρω μου και για το περιβάλλον μου και άρα και για ολόκληρο τον ε, πλανήτη όπως και για την οικονομία. Α θυμόμαστε ότι εμεί έχουμε εδώ ως ρόλο να διαφυλάξουμε ένα καλύτερο μέλο για του νέου μα και για τι επόμενε γενιές για το δικό τους το καλό. Για το μέλλον απαιτείται να έχουμε μια αποφασισμένη, αποφασιστική, αποτελεσματική και ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως απαραίτητο είναι να επιδείξουμε έργο. Δεν μπορώ παρά να τονίσω αυτή τη σημασία και γι' αυτό τη λέξη implementation, εφαρμογή, υλοποίηση, την έχω επαναλάβει τόσες φορές μέσα στην ομιλία μου. Οι δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης θα ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών λαμβάνοντας αποφάσεις και υλοποιώντας τόσο στο ιστορικό τους όσο και εδώ στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον ε, Πρωθυπουργό Σίπηλα για την ομιλία του οποίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρακαλώ τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Ζαν Κλοντ Ιουνκέρ, να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και ο Γύρκη, κατά έναν και εγώ, με μεγάλη χαρά συναντούμε τον φίλο Πρωθυπουργό της Φινλανδίας. Η Φινλανδία το 1995 κατέστη μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατατύχει την ίδια χρονιά και την ίδια μέρα ανέλαβε εγώ καθήκοντα ως Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. Από τότε μέχρι σήμερα, ε, πότε, πότε δουλεύει η Ευρώπη ικανοποιητικά. Και Σημείωσα εξ αρχής, διαπίστωσα εξ αρχής ότι από την πρώτη μέρα της ένταξής της η Φινλανδία είχε στάση και συμπεριφορά σαν να ήταν ιδρυτικό μέλος, σαν να ήταν ανέκαθεν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να πω ότι ορισμένα από τα ιδρυτικά μέλη θα μπορούσαν πολλά να αποκομίσουν αν ακολούθησαν το παράδειγμα της Φινλανδίας και ακολουθούσαν αυτή τη συμπεριφορά. Η Φινλανδία από την ε, ένταξή της έδειξε πάντα μία τάση να αφουγκράζεται οι κυβερνήσει της όλες ήξεραν να τίνουν ευικονούς η Φινλανδία αφουγκράζεται, αντιλαμβάνεται αυτό που ακούει και μετατρέπει σε πράξη αυτό που έχει αντιληφθεί στην πολιτική. Έχοντας ξεκινήσει με τον Παύλο Λίπον ως Πρωθυπουργό, με τον Κατάινεν μετά, με σένα εδώ. Να, αργότερα πάλι τρει πρωθυπουργού σήμερα από την Φιλανδική Προεδρία, ε, Φιλανδική ημέρα σήμερα, σπάνιο μεν, αλλά χρήσιμο. Τρει Φιλανδοί θα περάσουν από την ε, Επιτροπή σήμερα. Και έχουμε λοιπόν και την επόμενη Φιλανδική Προεδρία στον ορίζοντα, μια Προεδρία με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, καθώς ξεκινάει η Προεδρία της Φινλανδίας μετά τις ευρωεκλογέ. πριν από, την, από τον διορισμό του υποψηφίου Προέδρου της Επιτροπής και της Επιτροπής Λογικά και του νέου διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, αναλαμβάνεται καθήκοντα ως Προεδρία σε μια περίοδο που χρειάζεται πολύ επιδεξιότητα στη διαχείριση των Ευρωπαϊκών και τη ε, προεδρία. Όπω άλλωστε έχει αποδείξει η Φιλανδία ότι μπορεί να πράξει. Το έχει αποδείξει και σε προηγούμενε ε, Προεδρίες τη. Όσον αφορά τη σχέση Φιλανδία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καλύτερε δεν θα μπορούσαν να είναι. Έχουμε σχέση απόλυτη εμπιστοσύνη στη συνεργασία μα, όπω άλλωστε είδαμε και κατά την εγκαθίδρυση του Μηχανισμού ασφάλεια και Άμυνα όπω άλλωστε συμβαίνει και στον τομέα τη ενέργεια και των κλιματικών αλλαγών, όπω άλλωστε άλλωστε συμβαίνει και στην ανάπτυξη των υποδομών ε, διασυνδεσιμότητας στην υπεθρο ε, της Φινλανδίας και εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα, χάρη στην ε, ευκαιρία που μας δίνει η ανάληψη της Προεδρίας από την Φιλανδία, να αναπτυχθεί περισσότερο η διάσταση του ε, βόρειο αρκτικού κύκλου. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ε, μια περιοχή στο βορειοαρκτικό κύκλο που παρουσιάζεται διπλάσια αύξηση θερμοκρασίας από ό,τι στην υπόλοιπη φίλιο. Και άρα πρέπει να, υπάρχει, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, άλλωστε υπάρχει και σχετικό συμβούλιο. Τον Νοέμβριο που ήρθα στη Φινλανδία, συζήτησα με τον ε, Πρωθυπουργό την ιδέα για μια σύνοδο κορυφής των χωρών του Βόρειου Αρκτικού Κύκλου, διότι θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε η περιοχή αυτή, ο Βόρειος Αρκτικός, να μπει ως κύρια προτεραιότητα στην, ε, στο θεματολόγιο των ευρωπαϊκών εργασιών. Ταυτόχρονα όμως έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαία πράγματα η Φινλανδία και ως Προεδρία και μπορεί να κάνει και αυτό ελπίζω να συμβεί με την εμβάθυνση και της Νομισματικής Ένωσης κατά τη διάρκεια της ε, Φινλανδικής Προεδρίας, με την Τραπεζική Ένωση, με την ολοκλήρωση της κεφαλαϊκής αγοράς που μπορεί να μας εξασφαλίσει η Φιλανδική Προεδρία. Υπό τη Φιλανδική Προεδρία πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε και, αυτό είναι στο επίκεντρο αυτής της, αυτού του προγραμματισμού, και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή είναι η μεγάλη δουλειά, η σκληρή δουλειά που έχει μπροστά της Φιλανδική Προεδρία, στην οποία πιστεύω ότι μπορεί να στηριχθεί απολύτως στην ε, βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οτιδήποτε χρειάζεστε θα το προσφέρουμε έτσι ώστε στο Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό του Οκτωβρίου να ολοκληρωθεί αυτό το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει εφέτος να ολοκληρωθεί, να κλείσει δηλαδή ως συμφωνία. Ιδάλλως χάνουμε πολλές ευκαιρίες για κατάθεση προτάσεων προγραμμάτων και χρηματοδότησή τους. Θα ήμουν επίσης ευγνώμων προς τη Φιλανδική Προεδρία και μέσα στο πλαίσιο του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου αλλά και στον τομέα της εμβάθυνσης οικονομικής και νομισματικής ένωσης θα παρακαλούσα να ε, εισακούσει τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των διαδροτικών μέσων και τη σταθεροποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης αλλά και της ανταγωνιστικότητάς της και της ε, στεναρότητάς της, της έναντι εξωτερικών κλειδονισμών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε μπροστά μας Έχουμε ένα ζήτημα για το οποίο ο πολίτης περιμένει να έχει τη δυνατότητα η Οικονομική και Νομισματική Ένωση να είναι σε θέση να αντιδράσει καλύτερα στην επόμενη κρίση που θα βρούμε μπροστά μας. Και θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τη Φιλανδική Προεδρία, προ την Φιλανδική Κυβέρνηση, γιατί βλέπω ότι σκοπεύει να αποδώσει μεγάλη σημασία στο επενδυτικό σχέδιο του Γύρκη και το δικό μου. Ε, έχουμε αυτή τη στιγμή ήδη ξεκινήσει με την υλοποίηση περί τα 8 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Φινλανδία. Ελπίζω να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και σας εύχομαι κάθε επιτυχία τον Απρίλιο, κάθε επιτυχία για την ανάληψη της Φιλανδικής Προεδρίας στη συνέχεια. Κάθε επιτυχία για το μέλλον. Ευχαριστώ. Θα ήθελε άλλος βουλευτής να εγγραφεί στο κατάλογο για τη διαδικασία cars the Παρακαλώ, εάν ναι, παρακαλώ να το πράξετε αμέσως. Ιδάλλως θα κλείσω τον κατάλογο της ηλεκτρονικής εγγραφή, την ηλεκτρονική εγγραφή στον κατάλογο και παρακαλώ τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της ε, ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κύριο Μάνφρετ Βέμπερ, να λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώ ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια κρίσιμη συγκυρία όπου τον Απρίλιο θα εκφραστεί ο λαός σας και η Ευρωπαϊκή Λαή τον Μάιο. Θα έχουμε δημοκρατικές λοιπόν εκλογές του επόμενου τους επόμενους Ξέρετε ότι η πρωτεύουσά σας, ε, το Ελσίνκι, είναι για εμένα και για το κόμμα μας ε, ζωτική σημασία. Εκεί πήρα το χρήσμα του υποψηφίου στο συνέδριό μας. Και αυτό ακριβώς αναμένουν οι πολίτες να έχουμε συζητήσεις, να υπάρχουν υποψηφιότητες και μετά θα επιλέξουν οι πολίτες για το μέλλον μας και την κατεύθυνση της πορείας μας. Αυτέ είναι οι αρχέ τη εθνική και τη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Θα είναι στο κέντρο των εξελίξεων των επόμενων μηνών. Θέλω να συμμεριστώ μερικά σημεία τα οποία αναφέρατε. Να σας συμμεριστώ τις γνώσεις, τη σκέψη μου δηλαδή. Στηρίζουμε αυτά που λέτε για τη δημοσιονομική πειθαρχία. Μπορεί να φαίνεται τεχνικό αυτό το θέμα. Μπορεί να έχει να κάνει με τι αγορέ. Μπορεί να φαίνεται τεχνοκρατικό και ότι αφορά μόνο τι επιχειρήσει. Όχι. Είναι το μέλλον των παιδιών μα. Είναι θέμα βιαισιμότητα όταν αναφερόμαστε στην δημοσιονομική πειθαρχία. Και το ΕΛΚ και σε εθνικό επίπεδο με τον κύριο Όρπα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εμά και ο Γύρ και βεβαίω κατά είναι, είναι στο πλευρό σα. Θα μα έχετε πάντα στο πλευρό σα αν θέλετε να επιδιώξετε αυτήν τη βιωσιμότητα. Γιατί η βιωσιμότητα σημαίνει μέλλον. Δεύτερον, αντιδρώντα στην ε, ομιλία σα για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, εδώ θα σα επικρίνω κάπω. Γιατί ξεκινήσατε την ε, αναφορά σα στο πολιτέ πλαίσιο λέγοντα ότι πρέπει να καθοριστεί το ποσό. Αυτό μα λένε πάντα οι εθνικοί ηγέτες. Νομίζω πω δεν είναι σωστή προσέγγιση αυτή. Η σωστή προσέγγιση είναι ποιοι είναι οι στόχοι, ποια είναι τα καθήκοντά μα. ε, τι απαιτήσει υπάρχουν έναντι τη Ένωση. Πολλοί ηγέτε λένε πρέπει να καθορίσουμε του πόρου, αλλά μετά θέλουμε ισχυρού ελέγχου στα σύνορα, θέλουμε κυβερνοασφάλεια, θέλουμε περισσότερη καινοτομία στην Ένωση. Αν αυτέ είναι απαιτήσει έναντι τη Ευρώπη, τότε τα κράτη-μέλη πρέπει να δράσουν σωστά. Πρέπει να συμβάλλουν στον προπολογισμό. Πρέπει να υπάρξει επαρκή χρηματοδότηση για να ανταποκριθούμε στι προκλήσει των καιρών. Πρέπει λοιπόν πρώτα να αναφερθούμε στι προκλήσει των καιρών. Το τρίτο σημείο που θα αναφέρω στη σύντομη παρουσίασή μου είναι το πιο δύσκολο για όλου μα. Αυτό μας είπαν και 35.000 παιδιά όταν ε, διαδήλωσαν τι προηγούμενε εβδομάδε στην Ευρώπη. Καλή και ο Πάπας ε, Φραγκίσκο για να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια τη γη. Είναι η καταπολέμηση τη ε, κλιματική αλλαγή. Αναφερθήκατε αναλυτικά σε αυτό. Υπογραμμίζω. Ποιε πρέπει να είναι οι αρχέ που εμεί ω ΕΛΚ θεωρούμε ότι πρέπει να κυριαρχήσουν σε αυτή την αντιμετώπιση. Μία αρχή είναι ότι η αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή δεν είναι να απαγορεύουμε διάφορε δραστηριότητε και προϊόντα. Δεν είναι δυνατόν να λέμε στου πολίτε ότι δεν μπορούν να πάρουν το αεροπλάνο και να πάνε στη Μαγιόρκα για διακοπέ γιατί αυτό αυξάνει το αποτύπωμα άνθρακα. Όχι, δεν είναι η δική μα προσέγγιση. Ελπίζουμε στο μέλλον να πηγαίνουν ε, οι ταξιδιώτε στη Μαγιόρκα με αεροπλάνα που δεν θα μολύνουν. Αυτή είναι η προσέγγιση. Δεν μπορούμε να πούμε στι αναπτυσσόμενε χώρε ή στι αναδυόμενε οικονομίε ότι θα πρέπει να μην αναπτυχθούν περισσότερο. Δεν είναι απάντηση αυτό. Η απάντηση είναι ότι εμεί ω Ευρωπαίοι πρέπει να του παράσχουμε σε αυτέ τι αναπτυσσόμενε χώρε τι αναγκαίε τεχνολογίε, ούτω ώστε η ανάπτυξή του να μην έχει επίπτωση στο κλίμα. Αυτή είναι η απάντηση. Η καινοτομία είναι η βασική αρχή για μα. Δεύτερο σημείο. Για το διοξείδιο του άνθρακα. Πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτε τι κάνουμε. Οι πολίτε πρέπει να υιοθετήσουν τι αλλαγέ. Για παράδειγμα, στην αυτοκινοβιομηχανία. Πολλοί ανησυχούν για αυτέ τι αλλαγέ. Βλέπετε τις διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία και πολύ και εδώ στην αίθουσα. Μπορούμε να πληρώσουμε υψηλότερε τιμέ ενέργεια, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν όλοι οι συμπολίτε μα. Πρέπει λοιπόν να επέλθουν αυτέ τι αλλαγέ με τέτοιο τρόπο που να τι αποδεχθούν οι πολίτε. Να ενστερνιστούν την άποψή μα. Πρέπει να κερδίζουμε από αυτήν την αλλαγή και όχι να χάνουν κάποιοι. Και τέλο, για την κλιματική αλλαγή του δεξιού του άνθρακα, μαζί μπορούμε να δράσουμε. Εμεί καταστήσαμε δυνατή τη Συμφωνία των Παρισίων, εμεί κάναμε τα βήματα για να μειωθούν οι εκπομπές καυσαερίων από τα αυτοκίνητα, διοξιδίου του άνθρακα. Εμείς είμαστε πρωτοπορία παγκοσμίω στην καταπολέμηση στη μείωση δηλαδή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και αποκινούμε του πολίτε τους ε, πολίτες μας μπορούμε να επιτύχουμε πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο ομιλητής, Κόφοντ για τη σοσιαλιστική ομάδα Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Η πατρίδα σας Ιφλανδές είναι ηγετική δύναμη σε πολλού τομεί την καθαρή ενέργεια, την ισότητα των φύλων, τα κοινωνικά θέματα. Η Transparency International ε, κατέταξε στην υψηλότερη βαθμίδα διαφάνειας και μη διαφθορά στην Φινλανδία στον κόσμο. Ε, βεβαίως πρέπει να πω ότι μας έχετε προλάβει εμάς σε ορισμένα θέματα όπως είναι η ενέργεια, έστω τους Ουδανούς δηλαδή. Πάντως η Δανία, η Φινλανδία δείχνει ότι μπορεί μια μικρή χώρα να ε, βρίσκεται μπροστά στον κόσμο, έστω και αν γεωγραφικά είναι πιο απομακρυσμένη. Θα ήθελα όμως ε, να πω ότι δεν είδα σε εσά στην ομιλία σας αυτή τη φιλοδοξία να καταστείτε πρωτεργάτης, να ηγηθείτε, να σπρώξετε την Ευρώπη προς την βιώσιμη ανάπτυξη, την δίκαιη ανάπτυξη, την ε, ανοιχτή σε όλους ανάπτυξη. Πού ήταν τα λόγια που θα λέγανε θα κάνω τη ζωή των Ευρωπαίων καλύτερη τα όσα μας είπατε περισσότερο μου θύμισαν τα νεοφιλελεύθερα σλόγγαν της ε, χθεσινής μέρας και όχι τα φιλόδοξα σχέδια για το αύριο. Εμείς ε, οι σοσιαλιστές έχουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την Ευρώπη. Ε, πιστεύουμε ότι η γη μας... Η πόροι μας κινδυνεύουν από την ε, ρήπανση, από την κλιματική αλλαγή. Ο ατμοσφαιρικός αέρας που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, το χώμα πάνω στο οποίο περπατάμε είναι το μέλλον των παιδιών μας και έχουμε καθήκον να τα υπερασπιστούμε. Ωστόσο και οι πολίτες μας και οι εργαζόμενοι έχουν κουραστεί να πληρώνουν αυτό το λογαριασμό ενός πιο βιώσιμου τρόπου αναπαραγωγής και με δυσφορία βλέπουν ότι οι μεγάλες πολυεθνητές ρηπαίνουν χωρίς όμως να πληρώνουν το μερίδιο που τους αναλογεί σε δίκαιους φόρου. Πρέπει αυτό να αλλάξει πια. Πρέπει να αλλάξει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης να καταστεί ένας, ένα πραγματικό σύμφωνο βιωσιμότητας για την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν και έχουμε εμείς ένα σχέδιο για να προχωρήσουμε πιο μια προβιώσιμη, ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής για να είναι πιο ε, δίκαιες συνθήκες και η μετάβαση για τον πολίτη και την Ευρώπη. Και σήμερα Καλό τη Φινλανδία να ενώσει τις δυνάμεις της σε αυτό το σημαντικό αγώνα, να έρθει κοντά μας. Πρέπει εμείς να διαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση όπως εμείς την εννοούμε και όχι να αφήσουμε να επικρατήσουν οι δυνάμεις της καταστροφής. Πρέπει εμείς να ορίσουμε τους κανόνες και τους όρους του παιχνιδιού. Η απληστία ορισμένων ελίτ και ο αν η ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση μας οδηγούν στην καταστροφή. Μόνο έτσι λοιπόν με την κατάλληλη φορολόγηση, με τις συνθήκες εργασίας για όλους ισότιμες και τον κοινωνικό πυλώνα που δεν άκουσα ούτε κουβέντα να ξοδέψετε για αυτόν που με τόση δυσκολία υιοθετήσαμε εδώ στην Ευρώπη. Κύριε Πρωθυπουργέ, η δίκαιη φορολόγηση είναι το θεμέλιο του κράτους ε, προνοίας της Ευρώπης που είναι άλλωστε μοντέλο το ε, κοινωνικό κράτος στη Βόρεια Ευρώπη, στη Φιλανδία και τις άλλες χώρες. Ε, είδαμε από μία μελέτη την προηγούμενη εβδομάδα από τον καθηγητή Μέρφυ ότι 800 85 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το, το κενό στην χρηματοδότηση που χάνεται, στους σπόρους που χάνεται από την ε, φορολογία που δεν καταβάλλεται από τις μεγάλες πολυεθνικές. Έχουμε τεράστιο δυναμικό λοιπόν να αντλήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουν οι κατάλογοι με τους παραδείσους φορολογικούς ε, όχι μόνο έξω από την Ευρώπη αλλά και μέσα στην Ευρώπη. Γιατί ο πολίτης δεν καταλαβαίνει πως είναι δυνατόν εμείς οι πολίτες να πληρώνουμε όλο και πιο υψηλούς φόρους όταν η Facebook, η Google και άλλοι μεγάλοι μεγάλη ε, κόλωση, ε, πληρώνουν ελάχιστος και καθόλου φόρου στην Ευρώπη. Πρέπει να αλλάξει αυτό, πρέπει να προστατέψουμε το κράτος προνοίας, ε, όχι μόνο για να είναι ελεύθερος ο ανταγωνισμός, αλλά και δίκαιος ο ανταγωνισμός, θεμητός ο ανταγωνισμός για όλους αυτούς. Πρέπει να διωχθούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτοί οι οποίοι αποφεύγουν την καταβολή φόρου. Η ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων και της ιατροφαρμακής θρησκευτικής ε, πρόνοιας ε, και περίθαλψης κύριε Πρωθυπουργέ δεν θα είχε ε, ίσως ε, πραγματοποιηθεί στη Φινλανδία εάν υπήρχαν οι πόροι αυτοί που έχουν εξεφύγει. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε να μείνει κανείς έξω κύριε Πρωθυπουργέ. Βλέπουμε κάποιες δυνάμεις προσπαθούν να διαλύσουν την Ευρώπη. Χρειάζονται όμως αυτές οι ριζικές αλλαγέ που θα οδηγήσουν στην κοινωνική δικαιοσύνη. ω είναι ο αγώνας μας εμάς των Σελιδημοκρατών της Ευρώπης. Ελπίζουμε ότι οι φιλελεύθεροι και οι άλλοι προοδευτικοί θα ενωθούν στον αγώνα αυτό. Ευχαριστώ per il gruppo dei conservatori Τους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές ε, τον λόγο έχει η κυρία Ρόχναν Λέρνερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κοινό μας στόχος ε, είναι σίγουρα να αυξηθεί η ευημερία. Η αύξηση της ευρωπαϊκής ευημερίας και αυτό θα ήθελα ακριβώς να τονίσω το θέμα της μετανάστευσης, την ασφάλεια των πολιτών, την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και την προστασία των πληροφοριοδοτών. Κύριε Πρωθυπουργέ, είχατε δηλώσει δημοσίως το 2015 πως ε, θα θέσετε στην διάθεση των τον άσυλο τη μονοκατοικία σας με τις εννέα κρεβατοκάμαρες. Αλλά αυτό αναπαράχθηκε από τα ΜΜΕ και πολλοί νέοι από το Ιράκ είπαν ότι το άκουσαν αυτό και επέλεξαν ειδικά τη Φιλανδία. Πέρα από αυτό Ε, διάβαζαν ε, τις διάφορες ε, περιγραφές για την δωρεάν παροχή υγείας, εκπαίδευσης, την καθαρή φύση, τις ωραίες γυναίκες που τους περιμένουν, όλα αυτά στο Αλαράμπια που ήταν σαν τα του παραδείσου. Λοιπόν, εσείς απευθύνατε αυτήν την πρόκληση, έκτοτε έχουμε σεξουαλικά εγκλήματα και το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών έχει επιδεινωθεί. Αναγνωρίζετε τώρα ότι η πρόσκλησή σας αυτή οδήγησε στο να έρθουν πολλοί άνθρωποι που τελικά δεν έχουν κάποια βάση για να λάβουν άσυλο. Τα προβλήματα στις χώρες προέλευσης δεν μπορούν να λυθούν με το να μετακινηθεί ο πληθυσμός του στην Ευρώπη. Τα προβλήματα πρέπει να λυθούν εκεί. Δεν μπορεί η Ευρώπη να γίνει το Ταμείο Ενεργείας του πλανήτη. Λοιπόν, συζητάμε επίσης για την φροντίδα των ηλικιωμένων και ιδιαίτερα για μια εταιρεία που προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες. Μια τέτοια εταιρεία εξοικονόμησε πάρα πολύ κόστη με το να παραμελεί τους ε, ασθενείς ε, και πολλοί προσπάθησαν να αποφύγουν τους ε, φόρους και μετέφεραν το κεφάλαιο του φορολογικούς παραδείσους. Έχουμε λοιπόν πολλά προβλήματα που εμφανίζονται. Πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν μια κουλτούρα όπου όλα τα εγκλήματα, παραδείγματο χάρη η παραμέληση αυτών των ηλικιωμένων, η φοροαποφυγή και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα θα πρέπει να δηλώνονται αμέσως στις αρχές όταν παρατηρεί κανείς ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να θεωρούνται υπέρμαχοι του δημοσίου συμφέροντος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ε, κάποια κανάλια που θα τους επιτρέπουν να το κάνουν αυτό με τρόπο εύκολο και ανώνυμο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στη Φιλανδία. Τον λόγο τώρα έχει ο πρόεδρος των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, ο κύριος Φερχοφστάτ. Κύριε Πρωθυπουργέ, και εγώ ξεκίνησα ως Πρωθυπουργό Ζων Κλοντ Ιουνκέρ στη Φινλανδία, θα θυμάσαι ίσως. Η πρώτη σύνοδος κορυφή στην οποία έλαβα μέρο ο Πρωθυπουργός ήταν το Τάμπερε. Να, 98, τα θυμάμαι πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα ότι είχαμε τάρανδο στο μενού στη σύνοδο και επίση ότι εκεί αποφασίστηκε μια κοινή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ακόμα αγωνιζόμαστε να πείσουμε τα κράτη-μέλη για το σκοπό αυτόν. Χάρηκα από τα όσα είπατε, γιατί ξεκινήσατε στην ομιλία σας με τον Άκιο και έχω κι εγώ μια παράθεση των λόγων του, με βοήθησε ο Νίλς βέβαια, ο συμπατριώτης σας, που λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει τις ιδέες της κοινωνίας των εθνών και να χτίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στη δεκαετία του 20. Τα είπε αυτά. Ένα εγχείρημα υπέροχο, ένα εγχείρημα που πρέπει να οικοδομηθεί και βεβαίως στην ε, παρέμβαση σας άκουσα τρία σημαντικά θέματα στα οποία θέλω να σταθώ. Καταρχάς, Ευρωζώνη και διακυβέρνησή της και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν χρειάζεται μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση για να αντικατασταθεί η δουλειά που δεν κάνουν στο ιστορικό τα κράτη-μέλη από την εισαγωγή νέων μέτρων. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει, να κάνουν τη δουλειά που έχουν να κάνουν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα νέο νόμισμα βεβαίω, το οποίο όμω χρειάζεται και την δημοσιονομική δυνατότητα με τα ε, ασφαλή στοιχεία ενεργητικού σε με παγκόσμια απήχηση που θα κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο που θα αποτελεί ταυτόχρονα όμως και την ασφάλειά μας έναντι των λεγόμενων ασυμμετρικών ε, κλειδονισμών. Γιατί αυτό δεν μπορούν μόνο τους τα κράτη-μέλη το καθένα να τα αντιμετωπίσει. Δηλαδή συμφωνώ μαζί σας μεν, αλλά το ένα συμπέρασμα αντιφάσει και με το άλλο. Και το δεύτερο, εσωτερική αγορά. Λέτε ότι έχουμε την καλύτερη εσωτερική αγορά του κόσμου. Να το διορθώσω λίγο. Θα μπορούσαμε ίσως να είχαμε την καλύτερη εσωτερική αγορά του κόσμου. Εάν είχαμε μια ενιαία αγορά και στους τομείς της, ψηφιακής αγοράς, των κεφαλαίων, της ενέργειας. Και σε αυτό χρειάζεται ένας ρυθμιστής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άπαξ και υπάρξει αυτό, αυτομάτως θα δούμε να αναδύεται η εσωτερική αγορά, η ενιαία αγορά για τα ψηφιακά, για τα κεφάλαια, για την ενέργεια. Η άμυνα, τρίτη παρατήρηση η μεγαλύτερη διασπάθηση κονδυλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται αυτή τη στιγμή στο ότι δεν υπάρχει μια γνήσια ευρωπαϊκή άμυνα. Δαπανούμε χρήματα και για την άμυνα των... Ε, χρήματα περισσότερα από ότι οι Αμερικανοί, ακόμα και οι Ρώσοι, αλλά δεν έχουμε την αμυντική δυνατότητα. Γιατί, Γιατί επαναλαμβάνουμε τέτοια πράγματα επί 28 και ελπίζω ότι θα καταστεί η Ένωση Αμυντική προτεραιότητα της Φιλανδικής Προεδρίας. Τώρα η συμπρόεδρος... κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ που ήρθατε στη συζήτηση αυτή για το μέλλον της Ευρώπης. Στιγμή αυτή που μιλάμε, 10.000 ε, μαθητές κάνουν πορεία στους δρόμους ε, εδώ πέρα και στη Φιλανδία και μας δείχνουν πραγματικά ότι πρέπει οι άνθρωποι και ο πλανήτης ε, να προηγηθούν ε, των κερδών. Λοιπόν, σας παρακαλώ να δεσμευτείτε για το μέλλον, να ακούσετε τους νέους και να επενδύσετε στο μέλλον όταν μιλάμε για την προστασία του κλίματος, την εκπαίδευση και την συνεργασία των Ευρωπαίων. Στην προστασία του κλίματος η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια τεράστια ευθύνη και κάθε κράτος μέλος πρέπει να παίξει τον ρόλο του. Και χαίρομαι που αναφέρατε το ότι είστε προσιλωμένο σε αυτό, θέλετε να έχουμε πιο φιλόδοξου στόχου. ωραία πράγματα και αναφέρατε και την σημασία των καταβοθρών διοξιδίου του άνθρακα και η Φιλανδία βεβαίως είναι ευτυχής που έχει κάτι τέτοιο τα ωραιότατα φιλανδικά δάση και κυρίως χάρη στα δάση της η Φιλανδία έχει γίνει το κράτος πρόνοιας που είναι σήμερα αλλά υπάρχει και ένα σημαντικός παράγοντας στην κλιματική πολιτική ε, εχμαλωτίζουν το ισοδύναμο 20 εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα κάθε χρόνο. Οπότε είναι προς το κοινό συμφέρον μας να τα διαχειριστούμε με αηφόρο τρόπο. Αλλά σε αντίθεση με τα όσα μας λέτε εδώ πέρα, η κυβέρνησή σας προγραμματίζει υλοτομία στα δάση αυτά, ε, η οποία δεν είναι αηφόρος και είναι ιδιαίτερος υπερβολική. Και έτσι κινδυνεύει αυτός ο πλούτος που έχετε. Ελπίζω λοιπόν μετά την πολύ ωραία σας ομιλία σήμερα η κυβέρνησή σας να αναστρέψει αυτήν την ε, θέση της ε, για να διατηρήσει την κληρονομιά σας και τον ρόλο της ως καταβόθρας διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί εάν είναι να έχουμε μια οικονομία ουδέτερη ω προ το διοξίδιο του άνθρακα, χρειαζόμαστε περισσότερα δάση. Αντί να λέμε στου άλλου να έχουν περισσότερα δάση, πρέπει να διατηρήσουμε τα δικά μα. Χαίρομαι λοιπόν που αναφέρατε ότι θέλετε πιο φιλόδοξους στόχους. Είμαστε στο πλευρό σας. Και χαίρομαι που το κάνετε αυτό και στο Σκανδιναβικό Συμβούλιο. Ε, φέρετε το όμως και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους άλλους πρωθυπουργού για να προχωρήσει στην Ευρώπη. Αυτό θα είναι αποτελεσματική εφαρμογή και οι νέοι τους οποίους ανέφερα αυτοί θα διευθύνουν τις χώρες μας, ε, τις ε, κοινωνίες, την οικονομία προσεχώς και ελπίζω πολύ σύντομα. Και πρέπει να τους προετοιμάσουμε γι' αυτό και η Φιλανδία είναι διάσημη για το εκπαιδευτικό τους ε, σύστημα. Όλοι ήρθαν στη Φιλανδία για να αντιγράψουν ε, τα φιλανδικά σχολεία, αλλά λυπούμε για το ότι η κυβέρνησή σας ε, πλέον κόβει ένα δισεκατομμύριο ευρώ από την εκπαίδευση και την έρευνα. Χρειάζεται περισσότερη επένδυση σε αυτούς το όχι λιγότερη. Και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε όταν μιλάμε για το ΠΔΠ στο ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να συνεισφέρει στην ευημερία όλων των πολιτών και όχι μόνο σε όσων έχουν τα μέσα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχει πολύ περισσότερα καθήκοντα η Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα χρειάζεται και επαρκείς πόρους. Δεν θα δεχτούμε λοιπόν μείωση του προϋπολογισμού. Μόνο έτσι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τα όσα έχει αναλάβει. Επίση, αναφέρατε πόσο σημαντικές είναι οι κοινέ αξίες, το κράτο δικαίου και η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη και αναφέρατε τον κίνδυνο του λαϊκισμού και συμφωνώ. Όμως ε, και εσείς ε, συνεργάζεστε με δεξιούς ε, λαϊκιστές, ε, κάποιους από τους οποίους μόλις ε, ακούσαμε, οπότε νομίζω ότι γνωρίζετε πλήρως τις κοινέ προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρός μας. Εθνικιστικά και ακροδεξιά κινήματα κερδίζουν στήριξη στην Ευρώπη μέσω παραπληροφόρησης ε, στις, ε, καλά είναι λοιπόν τα λόγια, αλλά οι πράξεις έχουν σημασία. Εκεί πέρα δείχνουμε ότι είμαστε σοβαροί, ότι θέλουμε ακριβώς να οικοδομήσουμε αυτό το καλύτερο μέλλον μαζί. Καθώς λοιπόν θα έχουμε τη Φιλανδική Προεδρία αυτό το καλοκαίρι, ελπίζω η χώρα σας μετά να είναι στην προοδευτική πλευρά, να μας οδηγήσει προς τα ευρώς για μια ενωμένη και δίκαιη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Για την ΓΚΟΕ, NGL, τον λόγο έχει ο κύριος Ηλικιώτης. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζω από μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, της Βόρειας Πράσης Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Συζητάμε σήμερα για ακόμα μια φορά το μέλλον της Ένωσης. Ένα μέλλον που καθορίζεται όμως από τη συνέχιση των ίδιων αδιέξοδων και αντιλαϊκών πολιτικών. Των πολιτικών εκείνων που προωθούν τη φτωχοποίηση, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, προκαλούν την καταστροφή του περιβάλλοντος προωθούν τη στρατιωτικοποίηση αλλά και το φλερτ των κυρίαρχων πολιτικών κύκλων με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. πόσο πιο δυνατά χρειάζεται να το πούν οι λαοί τη Ένωση, πώ χρειάζεται ρήξη με τι νεοφιλεύθερε πολιτικέ λιτότητα, ρήξη με τι πολιτικέ σε βάρο του περιβάλλοντο, ρήξη με τι πολιτικέ του κοινωνικού κράτου. Μόλι την προηγούμενη εβδομάδα ξεχύθηκα στου δρόμου του Βρυξελό δεκάδε χιλιάδε μαθητέ, και εργαζόμενοι για αλλαγή της πορείας των πολιτικών για το κλίμα. στη γαλλία και αλλού οι εργαζόμενοι εκφράζουν το θυμό και την αγανάκτησή τους για τις πολιτικές οι οποίες τους στοχοποιούν. ακόμα και στη φιλανδία που αποτέλεσε παράδειγμα κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης η κοινωνία παρακολουθεί παγωμένη σκάνδαλα που ήταν αποτέλεσμα των ιδιωτικοποιήσεων και της απορρίθμισης στον τομέα της υγείας υποστελέχωση στις στέγες ηλικιωμένων λόγω ιδιωτικοποιήσεων ακατάλληλα φάρμακα στους ηλικιωμένους για αύξηση του κέρδους των εταιριών φροντίδας. Πριν από δύο χρόνια, από αυτό εδώ το βήμα, ο πρόεδρος Γιούνκερ αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει τον κοινωνικό της χαρακτήρα και κινδυνεύει να γίνει η άγρια δύση του κοινωνικού τάμπινγκ. Δεν παραδέχθηκε όμως και πολιτικές οδήγησαν εδώ. Οι πολιτικές που παράγουν την νεανική ανεργία, τη φτώχεια τι περιφερειακέ και κοινωνικέ ανισότητε, ενώ ταυτόχρονα λιένεται το έδαφο για την άνοδο τη ακροδεξιά, του ρατσισμού και τη ξενοφοβία. Όσοι δεν αναγνωρίζουν την αιτία προφανώ θα συνεχίσουν με τι ίδιε συνταγέ και στον ίδιο δρόμο. Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική αλληλεγγύη. Χρειάζεται να ανακατανέμεται ε, δίκαια ο παραγόμενο πλούτο για κοινωνική δικαιοσύνη όχι για τι τράπεζε και τι πολυεθνικέ. ένα άλλο δρόμο ανάπτυξη που να δημιουργεί μόνιμε αξιοπρεπεί εργασία και πλήρη εργασιακά δικαιώματα. να προασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα των στρατηγικών τομέων και υπηρεσιών κάθε χώρα. να ενισχύει την κοινωνική προστασία για του αδύναμου και όχι να διανέμει ευχολόγια χωρί μια δεσμευτική ισχύ όπω είναι ο περιβόητο ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα ούτε να δίνει πακτολό χρημάτων στο ταμείο για την άμυνα ενώ αποκόπτονται από τι κοινωνικέ δαπάνε την παιδεία και την υγεία. Πώ να μην διορωτούνται οι πολίτε τη Ένωση γιατί υπάρχουν 38,5 δισεκατομμύρια ευρώ για το νέο ταμείο για την άμυνα ενώ κλείνουν τα γεροκομεία στη Φιλανδία. Η Ένωση χρειάζεται μια τολμηρή πολιτική για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή σήμερα η βιομηχανία καθορίζει τι πολιτικέ για το κλίμα σύμφωνα με τι δικέ της ανάγκε. οι λαοί όμω απαιτούν πραγματικέ λύσει απαιτούν πολιτικέ αποφάσει που να θέτουν φραγμό στην ανεξέλεκτη και ασίδωτη δράση των πολυεθνικών επιχειρήσεων και δεσμευτικού στόχου για προστασία του περιβάλλοντο και αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. ακόμα πιο φιλόδοξου στόχου από τη συμφωνία του παρισιού τέλος η ευρώπη χρειάζεται μια πολιτική ασύλου και μετανάστευσης βασισμένη στο διεθνές δίκαιο στην ανθρωπιστική αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες αλλά και την αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη μέλη. χρειάζεται να δημιουργεί ένας μόνιμος μηχανισμός για τη φιλοξενία όλων των προσφύγων σε όλα τα κράτη μέλη ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός. κύριε πρωθυπουργέ για να γίνουν αυτά χρειαζόμαστε μια άλλη ευρώπη την ευρώπη για την οποία η αριστερά παλεύει την ευρώπη της ειρήνης της πραγματικής αλληλεγγύης της κοινωνικής δικαιοσύνης την ευρώπη των λαών. ευχαριστώ πρόεδρε. Ευρώπη για τη Δημοκρατία και την ε, Άμεση Δημοκρατία, η κυρία Νταμάτο, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περάσει από μια ριζική διαδικασία αλλαγής, αυτή που απαιτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες όλο και πιο έντονο, έντονα. Είναι παντού ορατά τα μηνύματα, οι δυνάμεις του κατεστημένου, τα κόμματα, τα φιλελεύθερα και τα σοσιαλιστικά χάνουν διαρκώς τις εκλογικές αναμετρήσεις. Οι πολίτες έχουν πλέον κουραστεί από την ε, αδικία, από τη ε, λιτότητα, από την διαφθορά και θέλουν την αλλαγή πλέον στις κυβερνήσεις των χωρών τους. Ε, έχουν στείλει λοιπόν πολλές φορές τους ε, προηγούμενους ηγέτες ε, στα σπίτια τους. Στην Ιταλία λοιπόν, η... για να σας δώσω μια εικόνα, η οικονομική πολιτική ήταν ισοδύναμη με μια οικονομική σφαγή, με μια καταστροφή. Όμως εμείς τώρα κάνουμε προϋπολογισμό ο οποίος δίνει δύναμη στον πολίτη, ο οποίος δίνει νέες επενδύσεις, ο οποίος περιορίζει της, την διασπάθηση χρήματος. Έχουμε ένα επίδομα κατώτατο στήριξης των εισοδημάτων, το οποίο η Φιλανδία το γνωρίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε πολιτική πρόνοια, γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε την αγορά εργασίας, αλλά θέλουμε να μειώσουμε και τη φτώχεια. Πάνω από 5 εκατομμύρια είναι η φτωχή στην ε, Ιταλία νέες δεξιότητες θα εξασφαλίσουμε για αυτούς που δεν έχουν θέση εργασίας και έτσι θα, αυξήσουμε την απασχόληση με ένα πιο εξειδικευμένο ε, εργατικό δυναμικό που θα διευκολύνεται έτσι και η πρόσληψή του. Θα ενισχυθεί χάρη σε αυτή την ενίσχυση εισοδήματο ε, και ιστορική κατανάλωση. Μια Ιταλία λοιπόν ενωμένη, μια Ευρώπη ενωμένη αλλά και αλληλέγγυα. Ε, ήταν πολλοί οι ψευτοπροφήτες της αλλαγής, ε, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτοί ε, οι οποίοι υποτάσσονταν στα λόμπι, όπως ο Μακρόν, παραδείγματι, όπως το θέμα της γλυφοζάτης στην Γεωργία που δεν θα, το, δεν θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτό πριν από μερικά χρόνια. Δεν μπόρεσε να μας κοροϊδέψει. Ο Μακρόν ακολούθησε τις υποδείξεις της ε, Μέρκελ και ε, ενέκρινε την παράταση χρήση του ισκλιφοζάτη ε, για λογαριασμό της Bayer που εξαγόρασε τη Μονσάντο το 2018. Α σταματήσει λοιπόν αυτή η υποκρισία, Ο πολίτη θέλει να δει πραγματικά και πράξει, γεγονότα. Θέλει μια Ευρώπη που θα έχει παγκόσμια αντανάκλαση, θα μιλάει με μια ενωμένη φωνή, μια μόνη φωνή. Και βεβαίω χρειάζεται μια ε, έδρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Ασφαλεία. Αλλά η Μέρκελ και ο Μακρόν κάθονται χώρια και συζητούν μόνοι του για το μέλλον το οποίο θέλουν να χαράξουν οι δυο του, ενώ θα το πληρώνουν οι 27. Και έτσι αποκλείουν τα 50 τα 500 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Αλλά δεν μπορούν αυτοί οι δύο να φτιάξουν, έστω και αν φτιάξουν ενότητα άμυνας, ένωση άμυνας, την ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται η συμμετοχή ολόκληρης της ε, Υπήρου. Η Ιταλία χωρίς να έχει ηγεμονικές διαθέσεις είναι η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη, είναι όμως εγγυήτρια ε, στην Ευρώπη για την ε, ενότητα, για την αλληλεγγύη. Και έτσι θέλουμε μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να περιλάβει και ε, τα θεσμικά όργανα, χωρίς όμως παρεμβατισμό, χωρίς διευθυντική συμπεριφορά που θα εξασφαλίζουν την ενότητα που δεν θα κρατάνε τις Βεξέλλες μακριά από τον πολίτη γιατί αυτό το έλλειμμα δημοκρατίας πρέπει να το αντιμετωπίζουμε όχι φτιάχνοντας ακόμα ένα χωριστό κύκλο λήψη αποφάσεων αλλά επαναφέροντας την διαδικασία λήψη αποφάσεων στο μόνο άμεσα εκλεγμένο όργανο που εκπροσωπεί τον πολίτη, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θέλει να αλλάξει η Ευρώπη πρέπει και να εγκαταλείψει τις πολιτικές λιτότητας που καταστρέφουν την εκπαίδευση, την υγεία, τη δημόσια, τα δικαιώματα και να σταματήσουν οι αυτοκριτικές, οι ψεύτικες του Γιουνκέρ για τα λάθη γιατί οι δρόμοι που ακολουθείτε είναι πάντα οι ίδιοι και απευθύνω έκκληση σας αγαπητοί συνάδελφοι ας ας, απορρίψουμε τη μακροοικονομική ε, προσέγγιση, την μακροπροληπτική προσέγγιση. Ας αφήσουμε κατά μέρο αυτές τις υποδείξεις των Βρυξελών, ας προστατέψουμε περισσότερο τους πολίτες. Είναι απαραίτητο αυτό και για την ανάπτυξη των χωρών μας, των περιοχών μας, για την ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων των περιβαλλοντικών. Πρέπει η Ευρώπη και μπορεί να αλλάξει αν είναι στο πλευρό του πολίτη και αν μπορεί να τους δίνει απαντήσεις και όχι προβλήματα συνέχεια και κολάφους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποργέτσιο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε. Φαντάζομαι ότι σας ε, ξαφνιάζει λίγο αυτή η συμπάθεια που δείχνουν όλοι οι Ευρωπαίοι προς την ε, χώρα σας όπως εκφράστηκε εδώ μέσα και ίσως πρέπει να κοιτάξουμε ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι, αυτούς που εσείς ονομάζετε λαϊκιστές, έχουν κάποιες επιφυλάξεις, γιατί όταν λέτε ότι είστε σε θέση να υποδεχθείτε 20-25 χιλιάδες πρόσφυγες, τη δική μας δουλειά κάνετε, γιατί βλέπουμε ότι ε, αυξάνεται η συνείδηση του πολίτη που δεν είναι ρατσιστής, που δεν είναι ξενόφοβος, αλλά που βλέπει ότι αυτή η άτακτη μετανάστευση αποτελεί ε, πηγή ανασφάλειας, δυσκολιών στην κοινωνική ένταξη, προβλημάτων τρομακτικών και ίσως θα ήταν πολύ πιο ευφυές και φρόνιμο να πει κανείς, όπως άλλωστε έχουν πει και κάποιοι από την ηγεσία του Κοινοβουλίου, θα ήταν καλό να προχωρήσουμε σε ένα σχέδιο Μάρσαλ για την Αφρική. Για τη σωστή λύση, η σωστή συνταγή δεν είναι η υποδοχή στις δικές μας χώρες και κοινωνίες, με μια διαδικασία ένταξης που είναι πολύ αργή αλλά και αδύνατη μερικές φορές αν αναφερθούμε σε ορισμένους που προέρχονται από περιοχές και πολιτισμό μουσουλμανικό επί παραδείγματι, που είναι πολύ δύσκολο να ενταχθούν στις κοινωνίες μας, αλλά θα ήθελα ιδιαίτερος ε, για εσά που εκπροσωπείτε εκπροσωπείται μια χώρα πλούσια και ένα μεγάλο λαό, ε, τη Φιλανδία, ε, να μας πείτε τι έχετε να πείτε για ένα σχέδιο Marshall που θα μπορούσε να εισαχθεί. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Αυτή η Ευρώπη η οποία έχει χάσει κάπως το δρόμο της είναι κάπως υποτίθεται ε, λαϊκιστική όπως λέγεται ε, δημαγωγική που όμως αναζητεί ένα ρόλο ιστορικό που της ανήκει να βοηθήσει τους αφρικανικούς λαούς όχι όπως το παρελθόν όμως χρηματοδοτώντας πολέμους και κερδοσκοπία αλλά με πραγματική γνήσια υποστήριξη που ίσως να περάσει και από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αυτού αυτού που, τους επιχειρηματίες που ξέρουν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητες του με σωστό τρόπο και που έτσι μπορούν να ξεριζώσουν και το πρόβλημα της μετανάστευση. και συγχωρέστε μου την έκφραση δημαγωγική ήταν η δική σα η προσέγγιση στην ε, μετανάστευση ήταν δημαγωγική όλη αυτή και αν εγώ ήμουν πραγματικός ε, Φινλανδός θα είχα επιλέξει να αλλάξω δρόμο. Αυτό που έχουν κάνει κάποιοι άλλοι με θάρρος στην Ευρώπη που μπορεί να κατηγορηθούν για ανεξογονοφοβία και ρατσισμό αλλά στην πραγματικότητα να ζητούν το γνήσιο δρόμο, το στον πραγματικό δρόμο, το δρόμο των δικών μας ιεραποστόλων που πήγαν μέχρι την Αφρική για να τους προσφέρουν πολιτισμό και εκπαίδευση να τους δείξουν το δρόμο. Ο Ντόν Μπόσκο, ο ιερέας που αν ζούσε ακόμα σήμερα όπως έγινε στο 19ο αιώνα στην ε, ε, η Ιταλία θα είχε δείξει τον τρόπο να δουλεύουμε, να αρχίζουμε να κάνουμε επιχειρήσεις και όχι να ερχόμαστε, να έρχονται εδώ στη χώρα μας, στις χώρες μας, να κλέψουν και να βιάσουν γιατί ποτέ αυτοί οι άνθρωποι στην Αφρική δεν έμαθαν να δουλεύουν σωστά και αυτό είναι το το σφάλμα, η υπετιότητα των εγκλημάτων που διαπράττουν αυτοί οι μετανάστε είναι δική σα, εσεί που ποτέ δεν δώσατε την εκπαίδευση σε αυτούς τους λαούς. Ο κύριο Φοντούλη με εγγεγραμμένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πρωθυπουργέ, αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Το κυριότερο όμω είναι η πατερναλιστική αντίληψη που τίνει να εδρεωθεί σε πολλέ από τι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει και στου ευρωπαϊκού θεσμού. Οι ηγέτε τη Ενώσεω λειτουργούν σαν να κατέχουν εκείνη την απόλυτη αλήθεια και προσπαθούν να επιβάλλουν την ιδεολογία του πολίτε πολλέ από τι αποφάσει των ηγετών είναι μη αναστρέψιμε δημιουργώντα στου πολίτε την αίσθηση πω ο δημοκρατικό έλεγχο μέσω των εκλογών είναι ανώφελο. χαρακτηριστικό και πολύ πρόσφατο παράδειγμα η συμφωνία των πρεσπών η οποία μάλιστα χαιρετίστηκε από το σύνολο των ευρωπαίων ηγετών. ο ελληνικό λαό εξέφρασε την ξεκάθαρη αντίθεσή του όμω η κυβέρνηση τσίπρα αδιαφόρησε δημιουργώντα τελεσμένα. συντασσόμενη η ευρώπη πίσω από τη συμφωνία αυτή περιφρονεί τη βούληση των ελλήνων εμφανίζεται ως εχθρική προς τα ελληνικά συμφέροντα. θα ήθελα να υπενθυμίσω τόσο σε εσά όσο και στους υπόλοιπους ηγέτες της ενώσεως και ιδιαίτερο στον κύριο τσίπρα πως η εξουσία σας πηγάζει από το λαό και έχει ισχύ μόνο όσο ο λαός συνεχίζει να την εγκρίνει. σύντομα όμως θα διαπιστώσετε πως η εκ μέρους σας απαξίωση των ευρωπαϊκών εθνών θα αφυπνίσει τους πολίτες και θα τους κάνει να σκεφτούν εθνικά. ευχαριστώ. Και τώρα έχει το λόγο για να απαντήσει στα ερωτήματα που το απευθύνθηκαν ο Πρωθυπουργό Φιλανδία. Παρακαλώ. Mr. President, thank you Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ομιλίες. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις σύντομα. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ Ζαν Κλόντ και Γιούρκη για τα καλά σας λόγια και βεβαίω και εγώ να σου πω πως ήταν μεγάλη μου ευχαρίστηση η συνεργασία με την Κομισιόν. Η γεγονό είναι πως ε, θα είναι δύσκολη η στιγμή που θα αναλάβουμε την Προεδρία. Θα έχουμε μια Κομισιόν, ε, θα έχουν γίνει ευρωεκλογέ, θα έχουν γίνει και οι δικές μας εκλογές πριν. Πριν από αυτό θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις του ΠΔΠ, το Brexit, ε, ο ΝΕ και τα λοιπά. Μεγάλα θέματα. Ζαν Κλοντ, ε, επίσης ε, είχατε δίκιο για τα ζητήματα της Αρκτικής ε, και την κλιματική αλλαγή. Εμείς είμαστε έτοιμοι για την Αρκτική Σύνοδο Κορυφής σε λίγες εβδομάδες. Το επενδυτικό ταμείο του Γιούρκη Κατάινεν είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς ε, μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο και στη Φιλανδία. Κύριε Βέμπερ, συγχαρητήρια για τον ε, ορισμό σας. Η συνεδρίαση του ΕΛΚ στο Ελσίνκι ήταν θετική και για εμένα καθώς ε, συνάντησα γύρω στους 10 συναδέλφους ταυτόχρονα. Συμφωνώ μαζί σας για τις οικονομικές αρχές για το ΠΔΠ το έχω ήδη συζητήσει με 17 συναδέλφους ε, για την κατάσταση που επικρατεί εκεί και οπωσδήποτε θα βρεθεί μια συμβαστική λύση κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Για την κλιματική αλλαγή συμφωνώ ότι θα πρέπει να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για να μπορεί ο κόσμος ε, να την δεχτεί και Τονίζω ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να κάνουν περισσότερα από ό,τι νομίζαμε. Π.χ. υπάρχει η δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχει ένα μικρό πανεπιστήμιο εκεί στην ε, Λαπωνία. Ε, πιάνουν το διοξίδιο του άνθρακα από τον αέρα και φτιάχνουν προϊόντα διάφορα. Και επίσης ε, και η χαμηλή τιμή της ηλιακής ενέργειας έχει μεγάλη σημασία. Σκεφτείτε λοιπόν το τι δυνατότητες δίνει αυτό στην ε, Αφρική. Κύριε Κόφοντ, μάθε φιλανδικά νομίζω στην ομάδα σας. Έχετε κάποιους φιλανδούς. Καλό είναι αυτό. η ευτυχέστερη χώρα στον κόσμο η Φιλανδία μπορεί να είναι αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι είμαστε και αυτοί που το κρύβουμε καλύτερα αν δείτε τις συζητήσεις στο εσωτερικό μας. Ανέφερα τον κοινωνικό πυλώνα. Επίσης, οι προτεραιότητες μας είναι η ισότητα των φίλων ε, Έχουμε παίξει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτών με τον ε, Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που δώσαν πολιτικά δικαιώματα στις ε, γυναίκες. Φορολογική παράδειση. Συμφωνώ πλήρω με αυτά τα οποία είπατε. Πρέπει αυτό να αφορά όλες τις εταιρείε και όλους τους πολίτες, ε, δηλαδή να πληρώνουν όλοι φόρους εκεί όπου παράγονται τα κέρδη. Αυτή είναι μια βασική αρχή. Κύριε Ρούχονεν θα απαντήσω στα φιλανδικά, αν θέλετε. Και σε αυτό το φόρουμ ε, είναι καλό νομίζω να ε, επαναλάβω το τι εννοούσα όταν είπα ότι διαθέτω το σπίτι μου. Ξέρετε ότι ε, είχα μια οικογένεια την οποία φιλοξένησα πράγματι γιατί είχε κάποια συνεργασία με το εξωτερικό στη χώρα της και ήταν χριστιανή σε μουσουλμανική χώρα και κινδύνευε η ζωή τους ε, κάθε μέρα. Ε, δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς ζούσαν πριν φύγουν η οικογένεια αυτή ήθελε να ε, έρθει να εγκατασταθεί στο σπίτι μου και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φτάναμε στην Φινλανδία σε μια τέτοια ατμόσφαιρα όπου θα έπρεπε τελικά να ανακαλέσω αυτή την οικογένεια για να την απόφαση για να προστατεύσω την οικογένεια αυτή γιατί μου είπε η αστυνομία ότι δεν ήταν ασφαλής η οικογένεια αυτή στο σπίτι μου. Γι' αυτό τελικά αναγκάστηκαν να μετακομίσουν αλλού. Μετά... Α, άλλος... Χοφστατ έχει και δουλειές. Λοιπόν, να απαντήσω στην ε, κυρία Κέλλερ. Έχω εργαστεί και σε προσωπικό επίπεδο για τα ζητήματα κλιματικής ε, αλλαγής και έχω υποσχεθεί η οικογένειά μου θα είναι ουδέτερη ως προς το διοξείδιο του άνθρακα στο τέλος του επομένου έτους. Έχω ηλιακά πάνελ, έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχω μειώσει την κατανάλωσή μου και έχω φυτέψει και τα σχετικά δέντρα. Οπότε το αποτέλεσμα τελικά είναι ουδέτερο. Αλλά είναι πολύ εύκολο για ένα άτομο να το κάνει. Οπότε χρειάζεται κοινή δράση σε τρεις τομείς, σε τρεις μορφές. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές και να συνεχίσουμε προς τα εκεί και βεβαίως να αυξηθούν οι καταβόθρες και ο φινανδικός τρόπος ο βιώσιμος ε, διαχείρισης ε, του δάσους είναι απόδειξη πως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος ε, διαχείρισης είναι και... αυτό είναι κάτι το οποίο στηρίζω. Επίσης ε, χαίρομαι για το ότι υπάρχουν νέοι τρόποι δέσμευση του διοξιδίου του ανθρακά απευθεία από τον αέρα και αποτελεί πλέον πηγή άλλων προϊόντων. Και πρέπει να φυτεύουμε και δέντρα. Αναφέρατε ότι έχουμε κάποια εμπειρία συνεργασίας με λαϊκιστικά κόμματα. Ε, το μήνυμά μου είναι ότι και τα λαϊκιστικά κόμματα πρέπει να αναλαμβάνουν ευθύνε κυβερνητικέ. Και έτσι ε, έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Να αναλαμβάνουμε ευθύνες ε, και έτσι θα απαντήσουμε, θα δώσουμε και απαντήσεις στον κόσμο. Αναφέρατε Κύριε Σιλικιώτη. Το ότι ο Ιαλα, γνωστός Φιλανδός αριστερός, είπε στην κοινοβουλία μας πως ο καλύτερος φίλος των φτωχών είναι ο κελισμένος προϋπολογισμός. Έτσι θα φροντίσουμε τους πάντες σε κάθε χώρα, κάθε μέρα. Γι' αυτό στην Φιλανδία τα επιδόματα είναι τόσο υψηλά πέρα από την ε, εκπαίδευση βεβαίως που είναι ίδια για όλους τους πολίτες μας. Κύριε Ανταμάτο, το ποσοστό απασχόλησης συμφωνώ ότι είναι βασικό για να ισορροπήσει η οικονομία και βεβαίως στηρίζω όλες τις ε, δράσεις ε, που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι εξαντλήθηκε ο χρόνος. Με ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Eh, και ευχαριστώ και τώρα θα περάσουμε στη διαδικασία Κατσιάη. Πρώτος ομιλητής, μάλλον ομιλήτρια, είναι η κυρία Γιασλοβιάσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε ε, Πρωθυπουργέ, ε, θέλω να σας πω ότι η Προεδρία σας ε, είναι πολύ, ήταν πολύ ισόρροπη, μιλάτε πολύ για προστασία του περιβάλλοντος ε, και των πολιτών. Είστε Πρωθυπουργό ε, σε μια χώρα η οποία έχει το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη, για να μην πω παγκοσμίω. Ε, νόμιζα ότι θα μιλούσατε πολύ για εκπαίδευση, παρόλο που είναι ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν θα προτείνατε να επιβληθεί παντού το ε, φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα που προετοιμάζει σήμερα καλύτερα τους μαθητές και τους μελλοντικούς πολίτες. Ε, το κοινωνικό κεφάλαιο είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο ακόμα και στην οικονομία. Σήμερα έχουμε ρομποτοποίηση, αυτοματοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα πρέπει να προετοιμάζουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν ε, ε, θα είναι προτεραιότητα αυτή της Φιλανδικής Προεδρίας. Κυρία Καμπούλα Νάτρη. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ότι δεσμεύεται τόσο πολύ η μελλοντική Προεδρία προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, βλέπουμε παγκόσμιες προκλήσεις και μόνο ε, από κοινού μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Βλέπουν ότι από την άλλη πλευρά της μάχης προσπαθούν να πάρουν το δικό τους δρόμο, αλλά είναι πολλά τα προβλήματα ε, για να βρουν αυτό το δρόμο του Brexit στην πορεία τους. Επίσης, μας είπατε, κύριε Πρόεδρε, ότι ε, ε, δεν είμαστε ε, προετοιμασμένοι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Είναι κοινή η στόχη, είναι κοινά τα προβλήματα και ο κόσμος περιμένει από εμάς να είμαστε πρωτοπόροι στην προσπάθεια αυτή. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στη νέα οικονομία. Ο κύριος ε, Γιούγκερ ε, έχει αναφερθεί και ο ίδιος στη σημασία της Αρκτικής και της Βόρειας Ευρώπη. Δεν έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας μόνο προς Ανατολάς και προς Νότον, αλλά και προς την Αρκτική. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και ένα... Πρωθυπουργέ της Φιλανδίας, κύριε Σίπηλα. Ήθελα να σας θέσω το θέμα της κοινή αμυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, χθες είχαμε την θλιβερή επέτειο των Ιμίων. Τα Ιμία είναι μια περιοχή που ανήκουν στην Ελλάδα. Δύο νησιά που ανήκουν στην πατρίδα μου. Και όμως υπάρχουν οι προκλήσεις και οι αμφισβητήσεις της Τουρκίας. Μάλιστα αυτές τις ημέρες τουρκικά πολεμικά περιπολούν στην περιοχή. Η Τουρκία συνεχίζει τις παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, στα ελληνικά χωρικά ύδατα απειλεί την ελλάδα με κάζους μπέλι σε περίπτωση που η ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. ο ερντογάν θέλει να ανατρέψει τη συνθήκη της λοζάνης και θέλω μια δήλωση σαφέστατη πρώτον στήριξη της ελλάδος απέναντι στις απειλές του ερντογάν και της τουρκίας και δεύτερον τη θέση σας για να υπάρξει μια πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης που επιτέλους η ευρωπαϊκή ένωση θα στηρίζει την Ελλάδα σε περίπτωση αμφισβήτησης των συνόρων της από την πλευρά της Τουρκίας. Να υπάρξει στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σύνορα της Ελλάδος, τα οποία είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Και θέλουμε μια σαφέστατη τοποθέτηση από εσά, κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί θα είναι μήνυμα απέναντι στον Ερντογκάν, απέναντι στις απειλές της Τουρκίας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κατάινεν. Ναι, το έχω ανοίξει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Σίπηλα, ε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που στην ομιλία της η ομιλία σας μιλήσατε για τον πραγματισμό που χρειάζεται, για τον ρεαλισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δράσεις της. Η ακαιρεότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οικονομική της βιωσιμότητα δέχεται πιέσεις από πολλές διαφορετικές πλευρές και υπάρχουν, ε, υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη να ξαναδούν σε νέα βάση τις μορφές συνεργασίας τους. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη στο διεθνές προσκήνιο. Κύριε Πρωθυπουργέ, πώς νομίζετε ότι μπορεί να προωθηθεί η ιδέα, ας πούμε, ότι η οι κλιματικέ αλλαγέ και η κατανομή του βάρου του μεταναστευτικού φαινομένου θα πρέπει να γίνει πιο εξισορροπημένα μεταξύ των κρατών μελών. Διότι εγώ η ίδια βλέπω ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντί μα. Και αυτό φαίνεται και από το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τι επερχόμενε ε, ευρωεκλογέ. Και ελπίζω, κύριε Πρωθυπουργέ, στην ομιλία σας να διορθώσετε κάποιος ε, παρανοήσεις για την ε, φιλανδική δασοκομεία και το κατά πόσο μπορεί να είναι βιώσιμο και στο μέλλον. Πρόεδρος, θα δώσω το λόγο σε όλους όσοι ζήτησαν να παρέμβουν. Ωστόσο, θα πρέπει να σεβαστείτε το ένα λεπτό ομιλίας που έχει αποδοθεί στον καθένα σας. Ιδάλω θα είμαι υποχρεωμένος να διακόπτω τις παρεμβάσεις γιατί έχουμε και τις ψηφοφορίες κύριος Μπούκνερ. Κύριος Μπούκνερ, ευχαριστώ. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ. Εδώ και ένα χρόνο και πάνω από ένα χρόνο η κυβέρνησή σας μαζί με τη Γαλλία και 8 ακόμα χώρες μπλοκάρεται οποιαδήποτε πρόοδο στην καταπολέμηση εξαγωγής τεχνολογίας παρακολούθησης σε δικτατορίες. Πέρσι η δική σας κυβέρνηση μαζί με άλλες πήρατε θέση κατά της προστασίας ε, των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε είδη διτής χρήσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς το υπερψηφίσαμε με 92% πλειοψηφία και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέραμε μια πρόταση για να προστατέψουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, είστε η επόμενη Προεδρία. Μέχρι σήμερα το Συμβούλιο έχει δράσει τελείως ανεύθυνα. Παγκοσμίω δημοσιογράφοι, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρακολουθούνται και ε, συλλαμβάνονται, φυλάσσονται και θανατώνονται με δική μας τεχνολογία. Ελπίζω να πάρετε σοβαρά ε, τις ευθύνες σας και να το αλλάξετε αυτό. Η κυρία Κίλωνεν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί Ευρωπαίοι αισθάνονται ξένοι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, να λοιπόν, γιατί οι λαϊκιστές βρίσκουν γόνιμο έδαφος. Όχι, θα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πιο ανθρώπινα. Είτε μιλούμε για την απασχόληση, είτε για το κλίμα. Όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν, να δουν τι δυνατότητές τους, να μην αισθάνονται ξένοι. Τι μπορεί να κάνει η χώρα σας ούτως ώστε να υπάρξει περισσότερη ισότητα, δικαιοσύνη, ε, κοινωνική ένταξη. Όχι πολύ δηλαδή να ενστερνίζεται το, το θέμα ότι είναι, ότι είναι δική του η Ευρώπη. Μην έχουμε μόνο την Ευρώπη της οικονομίας και του χρήματος. Πρόεδρος Γιάκον κονσάρι. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα πρώτα καλώς ορίσατε Πρωθυπουργέ Σίπηλα ή στο Κοινοβούλιο. Μα ονομάζουν τη συνείδηση τη Ευρώπη γιατί ασχολούμεθα με ανθρώπινα δικαιώματα που τη σήμερα ημέρα είναι πολύ σημαντικό. Λίγο με απογοητεύσατε από όσα είπατε πάντω όσον αφορά τα οικονομικά. Τι γίνεται όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία μια που η Φιλανδία και πάλι έχει τοποθετηθεί εν μέσω των ε, νεοφιλελευθέρων. Και τι γίνεται και για την μετανάστευση. Μας λέτε για επαναπατρισμούς. Κάπου κάπως αλλάξατε νομίζω τον τόνο, αλλάξατε την κατεύθυνση των εξαγγελιών σας. θα πρέπει να συζητούμε όλα τα θέματα και όχι μόνο το πώ θα καταστεί δυνατόν να στείλουμε πίσω αυτού του ανθρώπου στην ε, χώρα του. Πάντω, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και την Κομισιόν και το Συμβούλιο που είπατε τα θέματα τη Αρκτική. γιατί και στην Αρκτική η συνεργασία με την Ρωσία πάει καλά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. πρόεδρο, λόγω στον ε, επόμενο. Ευχαριστώ, έχω δύο θέματα. Ναι, έχω δύο προτάσει προ τον Φιλανδό Πρόεδρο και τον ευχαριστώ πρώτα-πρώτα την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης σχετικά δηλαδή με αυτό το οποίο συμβαίνει σαν ένα σπουδαίο λαό, σε τον μεγάλο λαό της Βενεζουέλας όλα αυτά τα οποία τώρα υποφέρουν σχετικά με αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ε, μπορέσουμε να δείξουμε ότι ασπαζόμαστε δημοκρατία ε, η ειρήνη ούτως ώστε να υπάρχει ελευθερία, πολιτικά δικαιώματα για όλους, να προστατεύονται γυναίκες, ανήλικοι. Ε, εσείς τι πιστεύετε σχετικά με αυτό το πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να αναγνωρίσετε τον ε, νέο πρόεδρο της Βενεζουέλα. Τώρα κάτι άλλο όσον αφορά τον Τιντάμπη και όσον αφορά τον του ανταγωνισμό, την οικονομία και το διεθνές εμπόριο. Κατέστη δυνατόν να αποσπάσουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα και να μην χρειάζονται οι επιχειρήσεις μας περισσότερη πλαισίωση. Ιωάννα. Το μικρόφωνο σας λέει ο Πρόεδρος. Χαίρομαι κύριε Πρωθυπουργέ που σήμερα συζητούμε Ζήσας εσείς ως Φιλανδός Πρωθυπουργός και εγώ ως Ευρωβουλευτή, εκπροσωπώντας την χώρα που τώρα ασκεί την ε, Προεδρία του Συμβουλίου της ε, Ένωσης. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί πρόκειψαν διάφορα σκάνδαλα. Σκάνδαλα για κάποιες δηλώσεις που λέγατε ότι είσαστε έτοιμοι να λάβετε την Προεδρία κατευθείαν από τη Βουλγαρία και έτσι να βάλετε σε παρένθεση τη δική μας. Ναι, βεβαίως. Είδατε τις δηλώσεις μας ε, και είδατε ότι μόνο η κυβέρνηση μπορεί να εξασφαλίσει την Προεδρία. Δηλαδή θα πρέπει να λάβετε υπόψη μόνο τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και όχι άλλες δηλώσεις. Είμαι πεπισμένος ότι τώρα που παρήλθαν κάποιοι μήνες μετά από αυτές τις απρεπείς δηλώσεις ότι έχετε αλλάξει ρότα και έναν μήνα μετά την άλεψη της Προεδρίας η χώρα μας ήδη έχει κλείσει διάφορα σημαντικά ζητήματα. Το μήνυμά μου είναι η συνέχεια. Ελπίζω να συνεχίσετε το έργο της Ρουμανικής Προεδρίας. Ο Ευχαριστώ και συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προαγάγει μέσω τη εξωτερική πολιτική διάφορε αξίε, να προστατεύονται αυτέ τι αξίε όμω και στο εσωτερικό τη χώρα. Δεν θα πρέπει αυτέ οι αξίε να ερμηνεύονται αυθαίρετα, ούτε θα πρέπει ε, οι Βρυξέλλες να ε, υπαγορεύουν πώ θα υλοποιούνται αυτέ οι κοινέ αξίες αυτές που ενώνουν όλο τον κόσμο. Τώρα όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς, πιέζεται κάποια κράτη-μέλη να υιοθετήσουν ε, ε, κάποια μοντέλα φιλελεύθερα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Οι αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μας ενώνουν. Ε, θα πρέπει να μας φέρνουν πιο κοντά. Δεν θα πρέπει να θεωρείται ο μπαμπούλα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε ότι είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία, αλλά ενωμένοι δεν είμαστε στην πραγματικότητα. Ε, είμαστε διαφορετικοί και αυτό θα πρέπει να το αποδεχθούμε και θα πρέπει επομένως να βαδίσουμε με πηξίδα την επικουρικότητα. Ο επόμενος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στο κοινοβούλιο κύριε Πρωθυπουργέ. Συνήθως λέμε ότι είναι απλό Ε, να βλέπει κανείς το τι δεν πάει καλά στον απέναντί του. Ε, αλλά εδώ μιλήσατε για ισοσκελισμένο προπολογισμό και μιλήσατε και τις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την ε, μαθηματική προσέγγιση που θα έπρεπε να έχουμε στην καθημερινή διοργάνωσή μας. Η Φινλανδία θα πρέπει να βοηθήσει και την Προεδρία που έχει αναλάβει να προωθεί στο θέμα αυτό και θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τη Φινλανδία στην Προεδρία της. Ευχαριστώ η κυρία Χάουταλα. Kiitos ε, puhemies ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, Πρωθυπουργέ. Ο κύριος Πρόεδρος έχει πει ότι ακόμη και κάποιες από τις ιδρυτικές ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μάθουν ε, πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι χτίζεται στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θέλω να ρωτήσω δύο διαφορετικά πράγματα. Ποια είναι η φιλανδική στάση και τι δυνατότητες υπάρχουν για το πώς ε, θα εξετάζονται οι φορολογικές συμφωνίες μεταξύ χωρών. Ε, κάποιες χώρες δεν μπορούν να λάβουν μέτρα εναντίον άλλων που αποφασίζουν διμερώς να ε, έρθουν σε φορολογικές συμφωνίες. Όμως πρέπει να πατάξουμε και τη φοροδιαφυγή. Ξέρω ότι το συζητάτε το θέμα στο Συμβούλιο, όμως η Φιλανδία δεν φαίνεται να υποστηρίζει την κίνηση αυτή, διότι αντίκειται στην εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Και μετά υπάρχει και το θέμα τη εταιρική ευθύνη στην Φιλανδία. Είμαστε πολύ ενεργοί στο να υπάρχει μια νομοθεσία για τα θέματα τη εταιρική ευθύνη. Οι εταιρείε θα πρέπει να υποβάλουν εκθέσει για τι συνέπειε των δραστηριότητών του στο περιβάλλον και σε άλλα θέματα. Και είναι σημαντικό αυτό για να τεθεί ω προτεραιότητα στη Φιλανδική Προεδρία. Ευχαριστώ. Κύριε Κούνεν, ευχαριστώ Πρόεδρε, Πρωθυπουργέ. Ε, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα ε, τη χρονιά που προετοιμάζεται για την τρίτη της Προεδρία η Φιλανδία και είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις φιλανδικές προτεραιότητες. Πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει ενώ και απογοητεύτηκα λίγο. Γιατί δεν μιλήσατε πολύ για την έρευνα και για την εκπαίδευση, για την παιδεία. Το success story της Φιλανδίας ακριβώς εκεί βασίζεται. Στο πάρα πολύ καλό εκπαιδευτικό μας σύστημα, το know-how, την τεχνογνωσία και την επένδυση στην καινοτομία που μας έχει κάνει από τις πιο καινοτόμες χώρες. Αυτά ακριβώς χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, ε, ε, ανταγωνιστικότητα σε μια ψηφιακή οικονομία που αλλάζει τον κόσμο. Ε, ρομποτοποίηση, αυτοματοποίηση, αλλάζει ακόμα και αγορά εργασίας. Εκεί οι μεγάλες αλλαγές, οι μεγάλες προκλήσεις και γι' αυτό ε, αναφερθήκατε και στην κλιματική αλλαγή και την καταπολέμηση της. Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ ε, εστίαση στην παιδεία, στην τεχνογνωσία, στην ποιοτική έρευνα και αυτό είναι το μήνυμά μας και για την επόμενη Προεδρία. ήθελε το Κοινοβούλιο να αυξηθούν οι δαπάνες για την έρευνα. Η Φιλανδία έχει αυξήσει τις δικές της δαπάνες, αλλά τι γίνεται με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα συμφωνήσετε με την πρόταση του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις αυτές. Eh, Ευχαριστώ. πολύ κύριε Πρόεδρε και σήμερα συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης και νομίζω ότι έχουμε δύο επαναστάσεις οι οποίε πρόκειται να σημαδέψουν τη ζωή μας σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Η τεχνολογική, η ψηφιακή και η ενεργειακή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επομένως να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και όσον αφορά την ενεργειακή επανάσταση που θα μας ε, σημαδέψει θα είναι ένα ορόσημο για το, το, το, τα ταξίδια, την κατανάλωση θα πρέπει να δειχθούμε ε, φιλόδοξη επίσης για την αλλαγή του κλίματος. Κατά αυτή την ε, θητεία έγιναν πολύ σημαντικά βήματα και έτσι η Ευρώπη να γίνει πρωτοπόρα σε αυτή την ε, ενεργειακή μετάβαση ούτως ώστε να απαλλαγούμε από τον άνθρακα και να πετύχουμε τους στόχους για το κλίμα. Δεν θα πρέπει όμως να καταθέσουν τα όπλα ή να χαλαρώσουμε γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα και θα πρέπει η ανταπόκρισή μας να είναι συνεχής. Κατσέρσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει οικοδομηθεί και διαρκώς υπονομεύεται. Ε, υπάρχουν όμως και άλλες ε, θεμελίες λύθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η νέα αγορά, η αγορά εμπορευμάτων και ε, προσφοράς υπηρεσιών. Είναι σαφές ότι κάποιοι θέλουν να παραβιάσουν την ελεύθερη κυκλοφορία. και όμως Είναι σημαντική η ελεύθερη κυκλοφορία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται πέντε μέρε για να πάει ένα φορτηγό από τη Φινλανδία στην επικράτεια τη υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Φινλανδοί ευρωβουλευτέ ήδη ε, πλήρωσαν για να μην χρησιμοποιηθούν κατεξοδότηση πράξη στο πακέτο τη ε, κινητικότητα. Εσείς μπορείτε να υποστηρίξετε τη λύση του Συμβουλίου. Δεν θα περιορίζατε έτσι τις ελευθερίες των πολιτών, τις οικονομικές τους ελευθερίες. Δεν θα άρετε έτσι οικονομικούς φραγμούς, ενώ έχουμε πει πανελειμμένως ότι οι φραγμοί αυτοί πρέπει να έρθουν. Είναι πολλές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πρέπει να κλείσουν να κατεβάσουν ρολά. Οι Φιλανδοί καταναλωτέ θα πληρώσουν το τηλεπιτερή ε, για τα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρωθυπουργέ, ε, συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε. Ε, την συνοχή της ε, ενιαία αγορά, το κράτος δικαίου. Ήθελα εδώ όμω να θυμίσω κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τη χώρα σας. Είπατε ότι δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να υπάρξουν ε, νέα σύμφωνα για το κράτο δικαίου. Όμω στην χώρα σα δεν εφαρμόζεται πλήρω το κράτο δικαίου. Ξέρετε ότι βάσει τη φιλανδική νομοθεσία ε, υπάρχουν οικογένειε που έχουν πάρει τα παιδιά έχουν ε, προσφύγει στα δικαστήρια και δεν μπορούν να παρουσιαστούν ε, στην εκδίκαση της υπόθεσής τους. Εγώ έχω συντάξει σχετική υποστολή. Ε, τι μπορεί να γίνει όταν τέτοιοι Ευρωπαίοι πολίτες με ευρωπαϊκή θα γίνει άλλη της χώρας σα δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά των Φιλανδών πολιτών. Θέλουμε μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση στο θέμα αυτό. Και επίσης, τι προϋποθέσεις μπορείτε να δημιουργήσετε για το κράτο δικαίου στη χώρα σας, γιατί βλέπω ότι ανάλογα με τη χώρα ε, το προσδιορίζετε διαφορετικά. Ευχαριστούμε. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, η ομιλία σας ήταν ε, πολύ πραγματιστική. Ε, βασίζεται σε πολύ καλά στοιχεία και δίνει και μια πρόπτικη για το μέλλον. Μιλήσατε για τη δασοκομεία και τις προπτικέ της. Περίπου το 70% της Φινλανδίας καλύπτεται από δάση. Έχουμε λοιπόν ε, ιδιαίτερες γνώσεις στον τομέα αυτό και ξέρουμε και πώς να διαχειριστούμε με βιώσιμο τρόπο τα δάση. Τα δάση είναι πόρος για την Ευρώπη και την Αφρική. Ε, είναι πνεύμονας και επίσης ε, προσφέρουν θέσεις απασχόλησης και επιτρέπουν να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές. Σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο όμως θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας και προς την Αρκτική και τα θέματα της Σκανδιναβίας γενικότερα. Στην περιοχή της Αρκτικής όπου ζω εγώ ίδια υπάρχει τεράστιο δυναμικό και φοβερή φυσική πόρη ε, τρομερή τεχνογνωσία επίσης αλλά και εδώ Πρέπει να αξιοποιήσουμε τους πόρους. Πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή ε, προσέγγιση στα θέματα της Αρκτικής. Ευχαριστούμε, ο κύριος Πόλτσακ. Ο κύριος Λόπος Αγγιλάρ. Πρόεδρε, σα σας ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ Σιπίλα, που ήρθατε για να μας δείξετε ότι η Φιλανδία είναι μια ευτυχισμένη χώρα μετά από 25 χρόνια συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το 1% του πληθυσμού. Θέλω να μιλήσω για τον Πολ Αρί Σπακ που είπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά κράτη. Όλοι μικροί είμαστε για τις προκλήσεις. Απλώς μερικές χώρε ξέρουν ότι είναι μικρέ και κάποιες άλλες δεν το γνωρίζουν ακόμα. Αυτά έλεγε ο τότε Βέλγος Πρωθυπουργός από τους πατέρες ιδρυτές. Μιλήσατε για τις, ε, την πολιτική άμυνας που είναι πρόκληση για σας και πρόβλημα που είστε ουδέτερη χώρα, αλλά δεν μιλήσατε για τη μετανάστευση. Παρακαλώ, ενώστε τις δυνάμεις σας για να απεμπλακεί ο κανονισμός του Δουβλίνου, όπως ήταν εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται κοινή πολιτική, χρειάζεται αλληλεγγύη για τη μετανάστευση. Καμία χώρα δεν μπορεί να εθελοτυφλεί ε, και να γεννάει από την άλλη όταν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη μας χτυπούν την πόρτα. Η κυρία Γιατενμάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ Σίπηλα θα διαπιστώσατε ότι είστε πάρα πολύ ευπρόσδεκτο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί οι βουλευτέ έχουν τόσε πολλέ ερωτήσει και οι Φιλανδοί οι ίδιοι βουλευτέ. που ε, νομίζουμε ότι είμαστε στη Φιλανδική ε, Βουλή στην ώρα των ερωτήσεων του Πρωθυπουργού. Ε, Εμεί είμαστε εδώ ίσω πιο ευπρεπεί από του φιλανδού συναδέλφου, δεν φωνασκούμε. αλλά τι γίνεται με την υλοποίηση και την εφαρμογή των αποφάσεων. Συμφωνώ μαζί σα το είπατε κι εσεί. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάνουμε βήματα, παίρνουμε φιλόδοξες αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν ακολουθούν στη συνέχεια τα κράτη-μέλη ε, με την εφαρμογή τους. Τι θα πρέπει να γίνει. Πρέπει να αλλάξουν τακτική τα κράτη-μέλη. Πρέπει όλοι να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση των νομοθεσιών οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι αρκετά καλά προετοιμασμένες ε, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, ε, εκεί που συνεδριάζουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Γιατί είναι αρκετά περίεργο αυτό. Μετά από τα συμβούλια ε, βγαίνουν διάφορες δηλώσεις τι σπουδαίο ήταν η συνεργασία και τι καλά που τα συμφωνήσαμε και μετά γυρνάνε στις πρωτεύουσε τους και δεν δίνουν συνέχεια. Θα φροντίσετε αυτές οι κοινέ αποφάσεις να εφαρμόζονται. Κάντε ησυχία σας παρακαλώ ο Πρόεδρος στα αγγλικά και καθίστε κάτω down, please. Now, the speech, the conclusion. Και τώρα θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό της Φιλανδίας να κλείσει τη συζήτηση. Παρακαλώ κύριε Σίπηλα, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις σας. Είμαστε συνηθισμένοι σε υποβολή ερωτήσεων. Κάθε πέμπτη το κάνουμε αυτό στο κοινοβουλίο μα. Όλοι οι υπουργοί οφείλουν να είναι παρόντες. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Αλλά μετά τις ερωτήσεις ακολουθούν οι απαντήσεις και θα πρέπει να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις. Πρώτα-πρώτα για την παιδεία η ισότητα στην παιδεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και το δημόσιο σχολείο είναι το καλύτερο και για πλούσιους και για φτωχούς. Όλοι οι Φιλανδοί, όλα τα παιδιά όλων των Φιλανδών πάνε στα ίδια σχολεία. Έχουμε τους καλύτερους δάσκαλους στον κόσμο και θα πρέπει ένα εκατομμύριο Φιλανδών να περάσουν από το σχολείο τα επόμενα δέκα χρόνια. Αυτή η πρόκληση νομίζω ισχύει για όλες τις χώρες της ε, Ένωσης. Είναι θέμα τεχνητής νοημοσύνης, είναι θέμα των αλλαγών. Τώρα για την αλλαγή του κλίματος. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, για το ότι συμφωνήσατε με αυτά που είπα και για όσα έφυξα ένα από σένα στην ομιλία. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση αυτή για μας και ειδικότερα Ανησυχούμε. το uh, Διοξείδιο του άνθρακος και αυτό είναι κοινό διαπραγμάτευση με είπα και με Ρωσία. Οι χώρε αυτέ ε, ενδιαφέρονται κάτι να κάνουν και αυτέ για το κλίμα. Τώρα για τι επενδύσει πρέπει να γίνουν σωστά. Τώρα, όσον αφορά την ε, συνεργασία στην άμυνα, τη συνεργασία αυτή εξ αρχή εμεί ε, θεωρούσαμε ότι είναι καλή ιδέα και θεωρούμε θετικό το ότι υπάρχει πρόοδο σε αυτό το μέτωπο. Τώρα, για την Τουρκία. Περίπλοκα τα πράγματα είναι χώρα του ΝΑΤΟ και είναι και θέμα το κράτος δικαίου στην χώρα που μας ανησυχεί έτσι όπως είναι η κατάσταση και βέβαια και το τι θα γίνει σε σχέση με την Κύπρο για την Ρουμανία. Ανέκαθεν ήμουν βέβαιος ότι η Ρουμανία θα τα πάει άριστα ως Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είδατε αποδείξεις αυτών που σας λέω. Θέλουμε να υπάρχει δημοκρατία, εκλογές, ε, ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα και βέβαια η χώρα μας θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις και φυσικά θα κάνει για θα συμμορφωθεί με ό,τι αποφασίσει η Ένωση. Είχαμε πάρα πολλά τα οποία ρώτησαν οι συμπατριώτες μου, οπότε στα φιλανδικά θα σας πω τα υπόλοιπα. Πρώτα πρώτα, όσον αφορά τη βιώσιμη δασοκομεία. 70% ε, με 80% στη χώρα μας από τα δάση τα χρησιμοποιούμε και τέλος πάντων ε, φυτεύουμε περισσότερα από όσα κόβουμε πώς να είμαστε ε, αποτελεσματικοί και βέβαια την κατασκευή των προϊόντων από ξύλο προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει με τη χρήση του άνθρακα Τώρα για το πολιτικο δημοσιονομικό πλαίσιο είχαμε πολλές ερωτήσεις και ω επόμενη ή, επόμενη προεδρία επί τη βάση των όσων έχω πει με του συναδέλφου, θα μπορέσουμε να κλείσουμε έναν συμβιβασμό για τις παραδοσιακές κοινοτικέ πολιτικές και για τις νέες προκλήσεις. Επιδεικνύουμε ευελιξία στην πολιτική μας και ως Προεδρία νομίζω θα βρούμε τις πιο εύστοχες λύσεις όταν έρθει η ώρα. Για υλοποίηση ε, τα είπα στην αρχή στην ε, εισήγησή μου και η παράδοσή μας είναι ότι όταν συμφωνούμε για κάποιο ζήτημα ε, τότε τηρούμε τα υπεσχημένα από την αρχή ε, νομίζω και για αυτό υπάρχουν αποδείξεις. Όταν αποφασίσουμε το κάνουμε με οριμότητα και στη συνέχεια προχωρούμε στην υλοποίηση της απόφασης. Ε, αυτό είναι το πιο ζουμερό μήνυμα της ε, ομιλίας μου. Ε, ευχαριστώ πρώτα, ήταν μεγάλη μου ευχαρίστηση να παραστώ σε αυτή την συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Πάλι ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. Prime Minister, thank you for your answer. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ για την απάντησή σας και για τη θέση σας ε, για τη Βενεζουέλα. Η συζήτηση έχει λήξει. Μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες, σας παρακαλώ. Μια στιγμή κύριε Καστάλντο, το έχω υπόψη μου θα ήθελα προηγουμένω να καλωσορίσω, προηγουμένω είπαμε, σας παρακαλώ, θα ήθελα να καλωσορίσω αντιπροσωπεία της Βολής του Καζαχστάν. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο διπλωματικό ε, αντιπροσωπεία της Βολής του Καζαξάν ε, με επικεφαλή τον κύριο Μοκτάρ Χερμάν είναι εδώ στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην 16η ε, Μικτή Κοινοβουλευτική ε, Επιτροπή. Χαιρόμαστε που σας υποδεχόμαστε εδώ και αυτό είναι ένα μήνυμα υπέρ της κοινή μας προσπάθειας ε, προώθησης και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Σας εύχομαι εγώνιμες συζητήσεις και καλή παραμονή στην Ευρώπη. Ποιος θέλει το λόγο? Παρακαλώ. Uh, uh, ναι, Πρόεδρε. Βάσει του άρθρου 11.3 του κανονισμού, σύμφωνα με το πολίτικο, ο εκλεκτός συνάδελφος Έρμαν Μπροκ θεωρεί σκόπιμο και απαραίτητο να βγάζουμε λεφτά από τις ομάδες των επισκεφτών. Δεν του φτάνουν τα λεφτά του, ο μισθός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όσα παίρνει από τον Όμιλο Μπέρτελσμαν. Αλλιώς να κάνουμε έρανο για τον κύριο Μπρόκ. like set... Και ε, θα ήθελα να αρχίσω ε, τον έρανο πέντε, δίνοντας 5 cents ή 5 λεπτά του ευρώ. Δεν ξέρω κάποιος άλλος να θέλει να δώσει περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μιράντα. Point of order. Για διαδικαστικό κι εσείς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, ναι, διαδικαστικό βάση του άρθρου 22 του κανονισμού μας. Ο Πρόεδρος θα ε, διευθύνει ε, και θα προεδρεύει σε όλα τα όργανα, σε αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου και θα εγγυάται την ε, ομαλή διαδικασία. Ο κύριος Σταγιάννη είπε ότι μίλησε με τον ε, αυτοανακηρυχθέντα ε, πρόεδρο Γουαϊδό για να του ε, εξασφαλίσει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι προθύστερο και κατά του κανονισμού. Και θέλω επίσημη απάντηση, γιατί ούτε είχαμε αποφασίσει, ούτε είχαμε ψηφίσει τότε. Το σημειώνουμε. Θα ψηφίσουμε, αλλά πριν την πρώτη ψηφοφορία θέλει το λόγο ο κύριος Καστάλτο. Ναι, ναι, ζητήσατε το λόγο. Θα σας το δώσω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, βάσει του άρθρου 188 εδάφιο δεύτερο, θεωρώντας ότι μεταξύ των ε, τροπολογιών που ουσιαστικά καταργούν την ελευθερία των πολιτικών ομάδων για τη σύνθεσή του. Υπάρχει μια μυστική ψηφοφορία για τα θέματα ε, τη διαφάνεια στο πώς λειτουργούν τα θεσμικά μας όργανα. Διαφάνεια είναι ένα σύμβολο πολύ σημαντικό για την πολιτική μας δράση. Γίνεται λοιπόν φάρσα αυτή η ψηφοφορία. Γίνεται ένα θέαμα θλιβερό και σκανδαλώδες που ρίχνει και αμαυρώνει την φήμη του Κοινοβουλίου. Ως μέλος λοιπόν του Κοινοβουλίου δε, απαιτώ να γίνουν σεβαστές οι απαιτήσει των πολιτών που θέλουν την διαφάνεια και ως Ευρωπαίος πολίτης ζητώ η Ολομέλεια να σεβαστεί την πολυφωνία και τη δημοκρατία. Γι' αυτό εξ ονόματα της ομάδας και βάσει του άρθρου 100 σας παρακαλώ συνάδελφοι, ομιλώ βάσει του άρθρου 188 εδάφιο ε, δεύτερο ζητώ την αναπομπή του κειμένου αυτού στην αρμόδια επιτροπή διότι θα γίνει μπούμεραν το κείμενο αυτό και θα ε, έρθει να χτυπήσει το ίδιο το κοινοβούλιο. Και σας ευχαριστώ για τη μεγάλη ε, προθυμία που δείξατε για να φροντίσετε να ψηφιστεί κρυφά αυτό το κείμενο θα αναπευθεί στην, ε, θα δούμε αν θα αναπευθεί σε αυτή την επιτροπή. Υπάρχουν αντιρρήσει για αυτή την πρόταση. Κύριε Κόρμπετ, έχετε το λόγο. Ναι, θα ήθελα να μιλήσω κατά της πρότασης. Η έκθεση που είναι ενώπιό σα συζητείται εδώ και ένα χρόνο περίπου στην Επίτροπη Συνταγματικών Υποθέσεων, ΑΦΚΟ. Συναισθήθηκε ειδική ομάδα εργασία με εκπροσώπους από κάθε πολιτική ομάδα. Ήταν πολύ ψηλή η συνένεση και τώρα έρχεται στην Ολομέλεια προς ψήφιση. Όπως κάθε έκθεση που έρχεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια ε, μπορεί να τροπολογηθεί και θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες. Ήδη αναβλήθηκε από το Δεκέμβριο στην 1η του Ιανουαρίου και από την 1η στη 2η του Ιανουαρίου. Υποπτεύομαι ότι αν το αναβάλουμε για το Φλεβάρι θα πάει λέγοντας Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Σαν την Τερέζα Μέη μας τα λένε εδώ λίγο. Κύριε, ακούσαμε το αίτημα αυτό και το αντεπιχείρημα. Θα θέσουμε, μα ψηφίζουμε το αίτημα του κυρίου Καστάλτο. Υπέρ, κατά, αποχές. Κύριε Καστάλτο, το αίτημά σας απερίφθη. Θέλετε τώρα πραγματικά επαλήθευση. Ωραία, ας το ελέγξουμε. Ε, το επιθυμείτε. Άρχεται η ψηφοφορία. Με επί του αιτήματος του κυρίου Καστάλντο. Πέρας. Απορρίπτεται. Προχωρούμε. Με την ψηφοφορία. Κύριε Μπρόκ, έχουν αρχίσει ψηφοφορίες για την έκθεση Κόρμπετ. Κύριε Μπροκ, έχετε 30 δεύτερα για να απαντήσετε. Κυρία Πρόεδρε, οι αιτιάσει του συναδέλφου είναι κάτι για το οποίο θα αναγκαστεί να ζητήσει συγγνώμη μια μέρα. Δεύτερο, γνωρίζω ότι είναι η απάντηση για τη χτεσινή μου ομιλία στο Brexit. Ε, όταν αρχίζουν να στριμώχνονται, τι κάνουν, ε, προχωρούν σε συκοφαντίες. Ποτέ εγώ δεν πρόκειται να ε, ξεπουλήσω τα συμφέροντα της Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που και τα λεφτά τους να δεχτώ ακόμα θα ήταν ηθικά ανεύθυνο. Nous λοιπόν στην ψηφοφορία για την έκθεση Κόρμπετ. Έχουμε τις ε, τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής, ε, ομαδική ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ε, η τροπολογία 20 σε τρία τμήματα, τρίμα πρώτο, ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Le vote clos. Χρειάζονται πάνω από 376 βουλευτές, όντως. Ε, ε, δεύτερο τμήμα με μυστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Le vote est clos. Πέραση ψηφοφορία εγκρίνεται. S'il vous plaît, mes chers collègues, troisième partie sans discontinuer. Σας παρακαλώ, συνεχίζουμε με μυστική ψηφοφορία και το τρίτο τμήμα, χωρίς διακοπές. Le vote est clos. Πέρας, εγκρίνεται. 35. Appel nominal, le vote est ouvert. Η τροπολογία 35 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 36 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 37, ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 38, με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 39, ψηφίζουμε ονομαστικά πάντα. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 41D έρχεται η ψηφοφορία, ονομαστική. Πέρας. C'est adopté. 42 Εγκρίνεται 42 με ονομαστική ψηφοφορία και αυτή, άχτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 43 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Βατίκλου. Πέρας. Εγκρίνεται. 44 πάντα ονομαστική άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 54 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 55 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 63 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 5D υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ονομαστική 10. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 11. Με απλή πλειοψηφία μπορεί να εγκριθεί. Υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι πάρα πολύ σαφέ. αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Απόχε. Απορρίπτεται. Ωραία, να την ελέγξουμε. Την 68. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ε, ζητώ συγγνώμη. Δεν εγκρίνεται, όχι. Χρειάζεται ε, ψηφοφορία ενισχυμένη 376 ψήφων. Δεν εγκρίθηκε. Ωραία. Θα προχωρήσουμε τώρα στην τροπολογία 13 σε δύο τμήματα. Ονομαστικά το πρώτο τμήμα. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρασε. εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, ονομαστικά, αρχίζει η ψηφοφορία. Le Πέρασε, εγκρίνεται. 75 ψήφιπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86 και 87 D με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Όχι, απορρίπτεται. Και πάλι ήθελε 376 ψήφους. Για όλες τις τροπολογίες χρειαζόμαστε ε, ενισχυμένη πλειοψηφία, εκτός από την τροπολογία 11 και για την τελική ψηφοφορία. 88 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 81 με ε, ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. Προχωρούμε στην τροπολογία 30... 73, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. 73. Με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την 30. Ψηφί πέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 32D. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Με ονομαστική κλίση η τροπολογία 40. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την 84D και 85D με ονομαστική ψηφοφορία και πάλι αρχίζει τώρα. Πέρας ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την 76. Ψηφίπε. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Όχι, εγκρίνεται, λέει η Πρόεδρος. Η τροπολογία 89 αναθεωρημένη με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και τώρα. Για την πρόταση απόφασης έχουμε ε, αρκεί απλή πλειοψηφία. Αρχίζει η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Σελίμοβιτς, Ενωσιακός Τελωνιακός Κώδικας. Ονομαστική ψηφοφορία για την ε, τροπολογία 1 αρχίζει και τελειώνει αμέσως. Εγκρίνεται. Έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Έκθεση Σικέρσκη. Ε, άμεσες πληρωμές και πάλι είναι μια ενιαία ψηφοφορία αυτή που αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται ολοκληρώνεται η πρώτη αναγνώση. Έκθεση Hannibal, πρώτη για τη Δομινικανή Δημοκρατία, ε, με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα, μία ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερη έκθεση Hannibal, η Σημερινός και Ουκρανία, με ονομαστική κλίση, αρχίζει ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτη έκθεση της κυρίας Χάνιμπολ για την Ονδούρα με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτη έκθεση Χάνιμπολ, Λευκορωσία και Ουσμπεκιστάν. Ε, ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα. Μία ψηφοφορία και αυτή. Πέρας. Έκθεση Πόγκα με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα. Για τις υπερπόντιες χώρες και τα εγκρίνεται. Έκθεση Μαρινέσκου. Ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων κλπ. Αρχίζει τώρα η ενιαία ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Πέρασε. εγκρίνεται. Έκθεση Φέντερλε με ονομαστική κλίση, τροπολογία 46, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία, υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτά του επίπεδου .eu. εγκρίνεται και η πρώτη αναγνωσή του Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται εδώ. Έκθεση Γκολτιέρη, εναρμόνιση του ΟΕΠ, τροπολογία 2, με ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Εγκρίνεται και ολοκληρώνεται η πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Προχωρούμε στην αντίρρηση για τη γενετικά τροποποιημένη ελαιοκράμβη. Ε, πρέπει να πω και τα νούμερα. MS8, ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα, RF3 και MS8. Πέρασε. εγκρίνεται. Αντίρρηση για το γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο 5307 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα πάλι για τον αραβόσιτο μόνο 87403 ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Αντίρρηση είναι και αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τέλος, αντίρρηση για το γεννητικά τροποποιημένο βάμβακα ε, με ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα, GHB 614. Πέρας. Εγκρίνεται. risoluzione. Περνάμε στην πρόταση ψηφίσματο κοινή τεσσάρων πολιτικών ομάδων για τη Βενεζουέλα. Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Γκονσάλε Πόν. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά τη σύνταξη αυτού του κοινού ψηφίσματο, ο Ρονάλντο Ντρίγκε, ο Χωσέ Σαλά, ο Βατίστε Ντεμοντιέρ, ο Πιέρ Καραλέ, ο Γκονθάλο Ντομίγκεθ, ο Λεωναρδό Μπουνιό, ο Μαουρέν Μπαρίγα συνελήφθησαν και κρατούνται στη Βενεζουέλα. Πρόκειται για δημοσιογράφου οι οποίοι εργάζονται για δύο ΜΜΕ ευρωπαϊκά και έκαναν τη δουλειά του. Από ό,τι είπε ε, ο πρόεδρος του, ΕΦΕ, του πρακτορείου ΕΦΕ τώρα βρίσκονται ε, στα κελιά της μυστικής υπηρεσίας. Ε, όλοι, όλοι εδώ είμαστε υπέρ της ελευθερίας έκφρασης. Το ημικυκλή όλοι είμαστε υπέρ του να μπορούν να ασκήσουν τον νημερωτικό τους έργο με ελευθερία τα ΜΜΕ γιατί όλοι πιστεύουμε ότι η ελευθερία της ε, ενημέρωσης είναι η ουσία της δημοκρατίας οπότε Ακριβώ όπως και οι άλλοι που έχουμε συνυποβάλει το κοινό ψηφίσμα θέλουμε μετά το σημείο 4 να υπάρξει ένα σημείο 4α, παράγραφος 4α που να λέει ότι καταδικάζει την φυλάκιση των δημοσιογράφων που καλύπτουν την κατάσταση στην Βενεζουέλα και απαιτούμε την άμεση αποφυλάκησή του. Και ευχαριστώ. Υπάρχουν βουλευτές που έχουν αντίρρηση για αυτήν την προφορική τροπολογία. Πρέπει να σηκωθείτε, τουλάχιστον 40, ε, εάν έχετε αντίρρηση. Ιδάλλως ψηφίζουμε για την τροπολογία. Υπέρ της τροπολογίας Γκοντζάλες Πόντς. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 5, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 μετά την παράγραφο 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ειδηλογική σκέψη G, πρώτη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την ειδηλογική G, 2, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Με ικανοποίηση ανακοινώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τον Χουάν Γκουαϊντό ως νόμιμο μεταβατικό πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πρώτο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που το πράττει και ζητούμε από τα κράτη-μέλη και την ύπατη εκπρόσωπο να ε, πράξουν το αυτό το συντομότερο έτσι ώστε να έχουμε ισχυρή και ενιαία θέση. Ολοκληρώσαμε με την έκθεση Ρεμό για την ετήσια ε, ανταγωνιστική πολιτική, πολιτική ανταγωνισμού. Θα ψηφίσουμε στο κείμενο. Τι γίνεται εκεί. Ναι. 30 δευτερόλεπτα. Μετά την Βενεζουέλα υπάρχει κι άλλη χώρα που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν υπάρχει καμία δημοκρατία καταπιέζουν τα δικαιώματα των γυναικών και τους αντιφρονούντες τους ε, καθαρίζουν, τους κόβουν κομματάκια. Ε, η Σαουδική Αραβία είναι αυτή. Κάτι να ψηφίσετε και για τη Σαουδική Αραβία. Στο κάτω-κάτω Και εκεί χρειάζεται αλλαγή καθεστώτος Και εκεί έχει πετρέλαιο. Και εκεί έχει πετρέλαιο. Να αλλάξουμε το καθεστώ. Πολύ καλά. Καταγράφουμε την παρατήρησή σα. Περνάμε στην έκθεση Ρεμό, ε, τη έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού, παράγραφο 2, αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση, έρχεται η ψηφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, έρχεται. Πέρας Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ονομαστική κλίση. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 4. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Αρχικό κείμενο σε δύο τα Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρόπο παράγραφος 28 αρχικό κειμένο πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική κλίση τροπολογία 9 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο ε, 40. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Μάλλον ονομαστική κλίση. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 41 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά να Απορρίπτεται. Πρώτη τροπολογία. Ονομαστική κλίση. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφο 76, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 78 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφό 82. Αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ονομάστηκε κλίση για την τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψήφισμα στο σύνολό του. Ονομαστική, ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Και τώρα περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου σε λίγα λεπτά. <laughs> Αρχίζουν οι επεξηγήσεις ψήφου σε ένα λεπτό. Συναληθυπότε παρακαλώ, καθίστε. Ξανά καθίστε. Euh, Διευκολύνεται όσον αφορά το να μιλήσουν όσοι θέλουν. Έχουμε και την έκθεση Κόρμπετ. Φαντάζομαι θέλουν κάποιοι από εσά να μιλήσουν. Ευχαριστώ που βγαίνετε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Monsieur Castaldo se prépare. Monsieur ne Κύριε Καστάλτο, μη φεύγετε, θα πάρετε το λόγο ευθύ αμέσως. Tant pis. Non Ok, il veut pas. Très Πάμε τώρα σε επεξηγήσει ψήφου. Έκθεση Κόρμπετ. Όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Κύριε Καστάλτο, γιατί το λόγο, αλλά θα τον λάβει ο κύριος Γκόρνης. Monsieur Castaldo, vous prenez la parole finalement Pardon, monsieur Golnisch, monsieur Castaldo est revenu dans l'hémicycle. Je vous demande une. Α, ξαναγύρισε ο κύριο Καστάλντο. Έχετε το λόγο. Κύριε Γκόλνη, που λίγη υπομονή. Συγγνώμη, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Απλώ θα ήθελα να δηλώσω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχή και από πλευρά τη πολιτική ομάδα ότι τελικά επικράτησε η λογική στο ημικύκλιο. Η έκθεση Κόρμπετ ε, όντω έχει κάποια σωστά σημεία για τον κανονισμό. Αλλά δυστυχώς αμαυρώνεται από το εξή. Πρώτα πρώτα είναι το πρόβλημα της ε, διαφάνειας ε, οπότε αυτά ε, έχουν θέσει και με το ότι θέλει και η ψημιστική ψηφοφορία το ΕΛΚ. Εμείς είπαμε ότι αυτό δεν συνάδει με τις τροποποιήσεις θεωρούμε ότι πρόκειται για κατάχρηση εξουσίας, ότι δηλαδή επιβάλλεται στην αντιπολίτευση η πλειοψηφία. Αλλά τελικά η δημοκρατική εκπροσώπηση και ο πλουραλισμός επεκράτησαν ούτως ώστε να μην είναι συγκεντρωμένοι εκεί που ήταν η, εξουσία. Κύριε Γκόλνης, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εδώ και 30 χρόνια είμαι μάρτυρας του ότι συνεχώς καταπατούνται τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Εδώ όλο ένα και περισσότερο γινόμαστε ε, στρατιωτικοποιημένοι ούτως υπήν ε, και τελικά έχουμε αυτή την έκθεση Κόρμπελ που μας ε, που να μας ρυθμίσει σαν ήμασταν παιδιά οπότε θα πρέπει να κάνουμε μαθήματα να μάθουμε ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι πολύ κακό πράγμα να υπογράψουμε δηλώσεις δεν μπορούμε πια να δούμε από κοντά τους συνομιλητές μας ε, εάν δεν το δημοσιοποιήσουμε στο βωμό της διαφάνειας. εδώ. είμαστε δημοτικό σχολείο. Με μεγάλη μου χαρά θα εγκαταλείψω το κοινοβούλιο. Πάλι. Πάρα πολύ ε, χαίρομαι που έχουμε τώρα ε, την έκθεση Κόρμπετ του συναδέλφου. Μ' αρέσουν οι προτάσεις του, ιδίως για την τον κώδικα διοντολογίας και για τις κοινοβουλευτικές ε, ερωτήσεις που θα πρέπει μέσα σε 6, μήνες, εβδομάδες να απαντώνται. 32% των εγγράφων ερωτήσεων προς την Επιτροπή απαντήθηκαν μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Δεν ξέρω, πήγανε σχολείο αυτοί οι άνθρωποι. 32% ε, σαν βαθμός δεν είναι και τόσο εντυπωσιακό. Να τα πάνε καλύτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτές οι ερωτήσεις. Έτσι ε, κατοχυρώνεται η υποχρέωση λογοδοσίας της Κομισιόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρείται αυτό το όριο των 6 εβδομάδων. Πολύ χαίρομαι για το αποτέλεσμα που αφορά αυτή την έκθεση. Δεν μ' άρεσε ο περιορισμό για τις ε, πολιτικές ομάδες. Αυτό είναι περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών. Όμως, είναι αυθαίρετες αυτές οι προτάσεις. Και ορισμός. Τι θα πει ιδεολογική συγγένεια, συνοχή μάλλον των ε, ομάδων. Εάν εφαρμοστούν οι προτάσεις αυτές θα διελύονται κάποιες υπάρχουσες πολιτικές ομάδες. Μα τι γίνεται, πάει στο καλάθι των αχρήστων η ελευθερία της ε, άποψης. Είμαι δημοκράτησα, πιστεύω στο κράτος δικαίου. Δεν είναι όμως δημοκρατικά αυτά τα οποία προτείνονται. Περικόπτονται οι ελευθερίες και αυτές οι προτάσεις αποτελούν επίθεση κατά της δημοκρατίας. Κύριε Μαριά. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να δηλώσω για να γραφτεί στα πρακτικά εντελώς διαδικαστικά ότι στην έκθεση σε Σελίμοβιτς το μηχάνημά μου δεν λειτουργήσε. Εάν λειτουργούσε θα ψήφιζα αρνητικά. Τώρα σε σχέση με την συγκεκριμένη έκθεση θέλω να πω ότι απέτυχε η προσπάθεια των μεγάλων πολιτικών ομάδων επί της ουσίας να επιβάλλουν αυτό το οποίο ήθελαν δηλαδή να κρίνουν αυτές υπό ποιους όρους θα συγκροτούνται πολιτικές ομάδες διότι η έννοια της πολιτικής σχέσης του political affiliation δεν είναι κάτι το οποίο θα το ρύθμιζε η ίδια η ολομέλεια και αυτό ήταν κάτι το οποίο το ανέλησα και χθε. από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξουν και άλλες βελτιώσεις στον κανονισμό ιδίως όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο που ασκεί το προεδρείο σε σχέση με τις ερωτήσεις διότι υποβάλλουμε ερωτήσεις και τελικά το προεδρείο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ελέγχει αν αυτές είναι σωστές και τις απορρίπτει ή όχι. αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο και θα πρέπει να σταματήσει. ευχαριστώ. Ο κύριος Φαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ψήφισα υπέρ των τροπολογιών για την αλλαγή στο εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, διότι για να μην είμαστε όμοιροι ιδεολογιών, δεν θα πρέπει να υποχωρούμε και στι ομάδε πίεση. Πρέπει να εργαζόμαστε για το συμφέρον όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών για την ατομική ελευθερία και τη δημοκρατία. Γι' αυτό θα χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στην πληροφόρηση για το τι σχέσει έχουν οι ευρωβουλευτέ με τι ομάδε πίεση, τι επαφέ έχουν με του εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών και σε τι συνεννοήσει έρχονται. Αυτό είναι χρέο όλων μα. Διότι υπάρχουν διαφορέ απόψεων μεν για το πώ πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω θέλουμε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση που να του εκπροσωπεί όλου και να, εκπροσωπούμε το, να εξυπηρετούμε τον ε, σκοπό για τον οποίο εξελέγουμε. Θα πρέπει λοιπόν να ε, βρισκόμαστε όλοι στον οίκο της δημοκρατίας ε, με απόλυτη διαφάνεια και τη σωστή συμπεριφορά. Ευχαριστούμε κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ. Υποστήριξα τι τροπολογίε για την αλλαγή του ιστορικού κανονισμού στο Κοινοβούλιο τη Εκθέση Κόρμπετ παρά το γεγονό ότι η τροπολογία 20 θα ήθελε να έχει δώσει διαφορετικό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία. Ε, διότι θα ήθελα να υπάρχει υποχρεωτική ε, αποκάλυψη των στοιχείων για τι συνεννοήσει των Πρόεδρων και των και την... Ε, το τι θα γίνει με την ομάδα εργασία που εξετάζει το θέμα τη γενική αποζημίωση. Είναι μια δημόσια σφαίρα που το Κοινοβούλιο έχει προβολή προς την κοινή γνώμη και σε όλους είναι θέμα του πώ λειτουργούν τα θεσμικά μα όργανα. Η διαφάνεια ε, είναι κάτι που εκτιμούν οι ψηφοφόροι μα και είναι σημαντικό και για την εκλογική μα δράση. Επίση, να καταγραφεί ότι δεν συμφωνούσα με την κρυφή ψηφοφορία, τη μυστική ψηφοφορία που οργανώθηκε από το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να γραφτεί αυτό στα πρακτικά και θα ήθελα οι ψηφοφόροι μα να ξέρουν πώ ψήφισε ο καθένα μα. Επίση, για την τροπολογία που αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των ε, ε, σχετικών ε, διατάξεων για την καταπολέμηση τη παρενόχληση. Πιστεύω ότι η εκπαιδευτική αυτή εκπαίδευση πρέπει να γίνεται για όλου του ευρωβουλευτέ. Ευχαριστούμε το μικρόφωνο σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση του κυρίου Κόρμπετ είναι αντιφατική. Περιορίζει τα δημοκρατικά δικαιώματα. Απαιτεί από εμά δηλώσεις βάσει των οποίων θα πρέπει να δηλώνουμε σε ποιο κόμμα ανήκουμε και ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετούμε. Αυτό νομίζω αντίκειται στους κανόνες του Κοινοβουλίου. Δεν μπορεί κανείς να αποδείξει τη στιγμή που ε, συστήνεται σε σώμα μια ομάδα την πολιτική του προέλευση και να είναι υποχρεωμένο να την αποδείξει. Θα πρέπει λοιπόν να μην καλλιεργήσουμε τέτοιο εχθρικό κλίμα μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ο κύριο Μάμικιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συνάδελφοι, συμφωνώ ότι όσο περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία υπάρχουμε στη διαδικασία ελλείψη αποφάσεων, τόσο καλύτερα. Ωστόσο, δεν μπορώ να συμφωνήσω με την έννοια τη πολιτική προσχώρηση. Ε, της πολιτικής συγγένειας. Ο όρος συγγένεια δεν έχει κάποια πραγματική βαρύτητα. Όπως είδαμε εκ του αποτελέσματος, κάποιες φορές οι πολιτικές ομάδες μπορεί να έχουν ε, διαφορετικές απόψεις σε κάποια θέματα μεταξύ τους στα μέλη των ομάδων. Γι' αυτό έχουμε και την ελεύθερη ψηφοφορία ως διαδικασία. Θέλουμε να προσωπήσουμε τις ανάγκες, τους Ευρωπαίους πολίτες στις ανάγκες τους. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε από την ε, συγγένεια με μια πολιτική ομάδα, από το, από την ομάδα στην οποία έχουμε προσχωρήσει. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο πώ ε, διαμορφώνουμε την ε, κρίση μα και γι' αυτό απήχα. Ευχαριστούμε κύριο Χάναν. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ε, εδώ το θέμα είναι ότι θέλουν να δυσκολέψουν τη ζωή στις μικρές ομάδες που δεν είναι τόσο ορθόδεξες ομάδες. Όχι, ακόμα και οι φεντεραλιστές συνάδελφοι ε, ε, το καταλάβουν ότι εδώ και χρόνια αυτό επιδιώκει το Κοινοβούλιο. Παρά τα όσα αντίθετα ακούμε για την διαλλακτικότητα, βλέπουμε μια διαλαξία. Θα ήθελα όμως να πω ότι θέλω να σα επιστήσω την προσοχή στη 14 τροπολογία. Για, για το άρθρο αυτό που λέει ότι δεν θα πρέπει να υπονομεύεται η ελευθερία του λόγου του βουλευτού ε, και δεν θα επηρεάζει τις ε, συζητήσεις. Αυτό το καταργείται. Τι έγινε, αλλάζουν τα ήθη στην Ευρώπη γενικότερα. Μα τελικά το κοινοβούλιο τι είναι κοινό βούλιο είναι εκεί όπου ο καθένας μπορεί να μιλάει ελεύθερα κανονικά από την ετοιμολογία της λέξης. Ο κύριος Σόσνιερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τροπολογία, ε, μάλλον η τροποποίηση του κανονισμού ε, που, μάλλον η τροπολογία που είχαν κάνει οι πολιτικές ομάδες, οι μεγάλες, για να φημώσουν τις μικρές, κατέπευσε. Ε, κατέπεσε, καταψηφίστηκε. Ε, η δημοκρατία απειλείται στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να έρθει στο κοινοβούλιο για να το διαπιστώσει. Εδώ είναι οι μικρές ομάδες ε, και ε, τις κατηγορείται για ακροδεξιές, ακροαριστερές, φασιστικές κτλ. Πού είναι η ελευθερία του λόγου. θα υπάρχουν εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου κατά της διαφάνειας και δεν θα μπορεί κανείς να λογοδοτεί ε, στους συναδέλφους του ή στους ψηφοφόρους του. Ε, αυτά τα μέτρα καταστολής είναι τελείως απαράδεκτα. Ε, ε, ε, ανέκαθεν στην ιστορία οι πλειοψηφίες ήθελαν να ελέγχουν τις μειοψηφίες ή οι πλειονότητες τις μειονότητες και να ταπεινώνουν ε, τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Και η, ρητορική ε, του μίσου, να σας πω ποια είναι αυτή η ισότητα, τα περισσότερα των φίλων. Ε, είναι το μίσος κατά των ανδρών. Ο κύριος ε, Πόλτσακ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. πρέπει να σας πω ότι εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή, την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού. Να σας πω και για ποιο λόγο. για την ρητορική μίσους ε, δεν με βρίσκει σύμφωνο η συγκεκριμένη τροπολογία. Ε, χρειάζεται ε, μεγάλη ελευθερία έκφρασης για τους βουλευτές, δεν διαφωνώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί ο βουλευτής στο όνομα της ελευθερίας του λόγου να προσβάλλει τους συναδέλφους και να τους υβρίζει. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επανειλημμένα νομοδοτήσει. Και, και βγαίνει εδώ και μιλάει ο κύριος Σόσνιερτς. Ε, ξέρετε τι μας έχει σύρει ο κύριος Σόσνιερτς εδώ πέρα μέσα. Ε, και τώρα μιλάει για ελευθερία του λόγου. Θα πρέπει να ε, τηρούμε κάποια στοιχειώδη ευπρέπεια στο Κοινοβούλιο. Και θα πρέπει να είμαστε πραγματικά ε, πολύ τυπικοί σε ό,τι αφορά αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Κυρία Πρόεδρε, καλωσορίζω τις προτάσεις της έκθεσης αυτής. Κατανοώ ότι ήταν καλές οι προθέσεις τους, ιδιαίτερα στα πλαίσια των συναντήσεων με εκπροσώπους το λόμπι. Επειδή εγώ έχω εργαστεί σε αυτό το κλάδο, φοβάμαι όμως ότι θα είναι αναποτελεσματικά και επίσης φοβάμαι ότι εύκολα αυτές οι προφορίες που θα δημοσιεύουμε θα μπορούν να διαστρεβλώνονται από ανθρώπους που έχουν λιγότερο αγαθές προθέσεις. Παρακαλώ αυτή η ρήτρα να αναθεωρηθεί μετά από κάποιο χρόνο. Και... Συμφωνώ με τον κύριο Πάλμερ ότι θα πρέπει να απαντούμε σε ερωτήσεις πιο γρήγορα. Για το θέμα των πολιτικών ομάδων γνωρίζουμε ότι οι ομάδες τύπου UKIP έχουν καταχραστεί ε, του, του κανονισμού αλλά ε, δεν ήταν ε, το αποτέλεσμα αυτό που επιτεύχθη το επιθυμητό. Και για το ισότητα του φίλου συμφωνώ. Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου για την έκταση του κυρίου Μαρινέσκου. Η κυρία Σόιντροβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχουν νεότερα για τα οικονομικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η φράση είναι κοινή νοήματος, διότι δική μας δουλειά είναι να παρακολουθούμε την εκτέλεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θέλουμε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μας. Η δημοκρατία της Τσεχίας είναι γνωστή για την κατάχρηση και υπεξαίρεση δημόσιων κονδυλίων και το τι έχει γίνει ε, με τους ε, αξιωματούχους μας υψηλού επίπεδου για τα προβλήματα που έχουμε. Πρέπει ο αγώνα λοιπόν αυτό για την κακοδιαχείριση, κατά τη κακοδιαχείριση να συνεχιστεί. Βλέπω οι παρανομίε και παρατυπίε να μειώνονται χάρη στη δράση μα και γι' αυτό είμαι υπέρ τη έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε κυρία Νταμάτο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και την καταπολέμηση τη απάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τι πιέσει των μεγάλων λόμπι που με το φαινόμενο των περιστρεφόμενων πορτών, όπω έχει ονομαστεί, μπορούν να καλλιεργούν τη διαφθορά που εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Και βεβαίω ένα άλλο θέμα είναι η έλεγχη για τα οικονομικά μέσα, το τι γίνεται με του μεσάζοντε και με τι νομικέ υποχρεώσει των δικαιούχων. Επίση, η απάτη στον κοινοτικό ΦΠΑ κοστίζει περίπου 50 δις ετησίως στην Ένωση. Οι ατασταλίες και πρατεπίες από το 2017 δείχνουν ότι είναι δεδομένα, είναι ανησυχητικά τα δεδομένα. Ε, με απάτες λόγω χάρη στον τομέα της γεωργίας. Έχει αυξηθεί το φαινόμενο της απάτης κατά 125% σε αυτόν τον τομέα. Δεν θα έπρεπε λοιπόν όλα αυτά να εξετάζονται με ένα ενιαίο σύστημα. Δεν υπάρχουν και και στο γενικό εντοπισμό των φαινομένων απάτη. Το ερώτημα αυτό γίνεται πιο κατεπήγον, δεδομένου το γεγονό ότι κάποια κράτη δεν επισημαίνουν καμία μορφή απάτη. Πώ γίνεται Μπορεί κάποια κράτη μάλλον απλώ να φοβούνται του ευρωπαϊκού ελέγχου ε, και το πώ χειρίζονται τα κονδύλια του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Την οικονομική και κυβέρνηση που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και πάνε μονομερό να παρακολουθήσουν την ε, απάτη που υπάρχει στη χώρα του, αλλά τελικά δεν καταγράφουν τίποτα. Με αυτά τα τεράστια κενά και πώς πώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η άμεση δημοσίευση τη έκθεση για τα πορίσματα σε σχέση με το φαινόμενο τη απάτη και διαφθοράς. Δεν αφορά αυτό άμεσα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα των ελέγχων και το όλο σύστημα. Πρέπει να υπάρχουν δείκτες αυστηρότατοι και ε, ομοιογενή κριτήρια που να ισχύουν δεσμευτικά για όλα τα κράτη-μέλη και να εφαρμόζονται ε, ε, χωρί κανένα χωρί καμία εξαίρεση. Θα πρέπει να ε, ισχύουν αυτά σε όλη την Ευρώπη και η Όλαφ να έχει πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα για να μπορεί να καταρτήσει τι απαραίτητε ε, υποθέσει με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ευχαριστούμε, γι' αυτό ψήφισα υπέρ. Ευχαριστούμε, αλλά πρέπει να σα διακόψω, κύριο Μαριά. Η καταπολέμηση της απάτης που υπάρχει σε σχέση με τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων αλλά και το ΦΠΑ νομίζω ότι πρέπει να ενταθεί. σε αυτήν εδώ την αίθουσα έχουμε καταγγείλει το πάρτι το οποίο γίνεται από τις διάφορες μκο στην ελλάδα που πραγματικά ε, έχουν χρησιμοποιήσει τεράστια κονδύλια στο θέμα υποτίθεται της προστασίας των προσφύγων αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι οι πρόσφυγες τώρα το χειμώνα κρυώνουν. εδώ σε αυτή την αίθουσα έχω κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες ακόμη να έχουμε αποτέλεσμα από την όλαφ ακόμη να έχουμε αποτέλεσμα από την κομισιόν. το δεύτερο θέμα είναι οι απάτες στον τομέα της αγροτικής πολιτικής διότι αυτό που συμβαίνει είναι να βαφτίζονται ξένα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα ως ελληνικά, αυτά που λέμε ελληνοποίηση. Και έχουμε έτσι ελληνοποίηση γάλακτος που εισάγεται από την Αλβανία, ελληνοποίηση κρεάτων που εισάγονται από τα Σκόπια και πρέπει να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα. Είχε δεσμευτεί και ο κύριος Έντιγκεν ότι στο θέμα αυτό θα παρέμβει η Κομισιόν. Περιμένουμε ακόμη να ληφθούν μέτρα. Ευχαριστώ. Έχουμε νέα θέματα που προσθέτουμε στην εμείς διάταξη, οπότε πολλές φορές δεν υπάρχει ευκαιρία να γίνει αυθεντική συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε η συζήτηση να έχει γίνει αυτό τελώς. Άρα, για τα οικονομικά σχέδια της Ένωσης δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα θα μπορούσα να πω Πρώτα πρώτα υπάρχει απεσιοδοξία. Απεσιοδοξία γιατί το 17 σε σχέση με το 16 αναφέρθηκαν πολύ λιγότερες αντικανονικότητες. Και σε σχέση με το 16 είχαμε μισό δις ευρώ δηλαδή 20% αύξηση της αντιμετώπισης των παρατυπιών. Συμπαθάτε με κυρία Τζαμπάσκη. εντάξει, εντάξει. Κυρία Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση. Νομίζω ότι η εθνική κυριαρχία είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να προστατευτεί. Στην έκθεση λέει ότι όλες οι παρατυπίες που έχουν επισημανθεί το 2017 αποδεικνύουν ότι παρατυπίες 50.213 τον αριθμό δηλαδή λιγότερες από όσες την προηγούμενη χρονιά και έχουμε ένα σωρό αριθμητικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να εντείνουμε την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θεμητώ αυτό και συμφωνούμε. Όμως στην έκθεση αυτή έχει κάποιες ε, αντιφάσεις, δηλαδή κάποια στοιχεία τα οποία αντιβαίνουν στην αρχή της εθνικής κυριαρχίας. Ο επόμενος, Μαμίκινς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταπολεμήσουν ε, ε, ότι είναι αντίθετο στα οικονομικά συμφέροντα τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο είναι φυσικό και παντού γίνεται αυτό. Όμω η διαφορά δεν έχει σταματάει στα εθνικά σύνορα. Επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ε, έτσι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη του πολίτη στα θεσμικά όργανα και στη δημόσια διοίκηση γενικότερα. Θα πρέπει όλες οι διοικητικέ αρχές να διαβάσουν αύριο την έκθεση αντί να διαβάσουν εφημερίδα. Τα στοιχεία είναι ισοπεδωτικά. Έχουμε 50, 50 δις. Έχουμε ιδίω για τον ΦΠΑ μεγάλη ε, απώλεια εσόδων λόγω του Σαπάτης θα πρέπει στου 28 ή 27 να έχουν περισσότερη διευκόλυνση όσον αφορά την λειτουργία διοικητικών αρχών. Χάναν. Ναι, είναι προφανέ ότι θα πρέπει να προστατευτούν τα οικονομικά συμφέροντα τη ε, Ένωση. Και έχουμε και αυτό το έλλειμμα των 50 δι. Αυτό δεν θα είναι γεγονό. Σύμφωνα με όσα είπαμε χτε για το Brexit, χωρί συμφωνία δεν θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη θέληση να μην γίνει άτακτο Brexit. Μα ταυτόχρονα θα λέμε ότι περιμένει η Επιτροπή να καταβληθούν αυτά που οφείλει η Βρετανία ακόμα και αν δεν υπάρξει deal. Πότε δεν είπε όχι η Βρετανία για τις υποχρεώσεις της και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διευκολυνθούν οι μέλους στις θέσεις. Αλλά όταν είναι no deal, δεν κονάτε το δάχτυλο. Πολύ τσακ. Ευχαριστώ. Εγώ ψήφισα υπέρ. Γιατί πρώτα πρώτα θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου στο ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, δηλαδή τώρα έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό απάτης, λιγότερες παρατυπίες, αυτό είναι πάρα πολύ θετική τάση. Ακόμα και αν έχουμε κάποια σκαμπανεβάσματα νομίζω ότι η μακροπρόθεσμη τάση είναι θετική. Άρα να κάνουμε ό,τι μπορούμε να διεκπαιρεώσουμε όσο γίνονται περισσότερες υποθέσεις. Επίσης η τροπολογία που είναι υπέρ της ελληνική δημοσιογραφίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Είδατε ότι δολοφονήθηκαν ε, τέτοιοι δημοσιογράφοι σε Μάλτα και Σλοβακία και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα η διαπλοκή της πολιτικής με τα ΜΜΕ. Τότε δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Ευχαριστώ και περνούμε στις επεξηγήσεις ε, για την έκθεση του κυρίου Φέντερλε, πρώτη κυρία Σόντροβα. Κυρία Σόντροβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι η έκθεση αυτή ε, με βρίσκει σύμφωνη και την υπερψήφισα. Ακόμα και αν φαίνεται κάπως τεχνική, ε, είναι πάρα πολύ σημαντική για την ε, προβολή της ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη. Σήμερα το ίντερνετ συνδέεται με την ε, προστασία των δεδομένων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, πράγματα που ενδιαφέρουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να επεκταθεί σε όλο τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Είναι πολλές οι οικονομικές διασυνδέσεις στον ΕΟΧ και αυτό είναι ένα πράγμα ε, που αφορά και την ανάπτυξη την ίδια των κρατών μελών. Ο κύριος Στρογεύσκη. Ευχαριστώ. Μετά το τέλος της συζήτησης μου έχουν ε, γεννηθεί μερικά ερωτηματικά. Ας πούμε, ε, ποιο είναι το πεδίο ε, εφαρμογής του ονόματος τομέα ανωτά του επίπεδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε με ικανοποιητικό τρόπο. Έχουμε πολλά τέτοια domain names, δηλαδή ονόματα τομέων ανωτά του επίπεδου και ποιος τα διαχειρίζεται και ποιος ελέγχει πώς λειτουργούν υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε και που πρέπει να τονίσουμε. Πρέπει να ξεφορτωθούμε παροχημένους κανόνες και νομοθεσίες. Επίσης, πρέπει να ορίσουμε προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον σημερινό επιγραμμικό ψηφιακό κόσμο. Θα πρέπει επίσης να χαλαρώσουν οι κανόνες ε, καταχώρησης ε, ε, ονόματος τομέα, ανωτά του επίπεδου, domain name, και να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στις εταιρείες που καταχωρίζουν αυτές τις ε, ονομασίες και τα ίδια τα ονόματα. Ο κύριος Κέλλη, ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Φρέντερικ Φέντερλε για την εργασία του ε, και ε, για την έκθεσή του την οποία είχα χαρά να υπερψηφίσω. Ε, αυτό το .eu είναι γνωστή μάρκα εσύ στην αγορά. Το ψηφιακό το οποίο αλλάζει συνεχώς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ε, κανονικά να γίνεται η ενημέρωση και η επικαιροποίηση έτσι ώστε να είμαστε εξασφαλισμένοι για το μέλλον. Να υπάρχει μια ευέλικτη χρήση, ε, η ε, των ευρωπαϊκών αξιών, προστασία των καταναλωτών, της ιδιωτικής ζωής, της πολυγλωσίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προστατεύονται όλοι οι κάτοικοι και όλες οι εταιρείε που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το domain Και ε, όταν χρησιμοποιείται κακόπιστα να ε, μπορούν να τους το αφαιρούν κιόλας. χαίρομαι ε, και για τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία των φορέων με το Γραφείο Πνευματική Ιδιοκτησία. Ο κ. Μαμίκιν, σε ευχαριστώ. Καλωσορίζω την έκθεση του συναδέλφου Φέντερλε και την υπερψήφισα. Ε, ωστόσο, παρά το γεγονός ε, ότι το τελεία .eu λειτουργεί καλά. Ε, υπάρχει μια νέα ψηφιακή οικονομία, νέα ψηφιακή αγορά και πάντα θα πρέπει εμείς να σκεφτόμαστε ένα βήμα πιο κάτω, πιο μπροστά. Ε, το νομικό πλαίσιο λοιπόν χρειάζεται να προσαρμοστεί. Το όνομα τελεία .eu είναι και ένα κοινό στοιχείο της ψηφιακής μας ταυτότητας. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ ποιος θα το χρησιμοποιεί αυτό και πώς. Πολυγλωσία, προστασία των καταναλωτών, προστασία της ιδιωτικής ζωής, ε, βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να ε, τηρούνται ως κριτήρια για να δίνεται το .eu. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ελέγχει και να ορίζει κριτήρια και διαδικασίες για την καταχώρηση ενός ε, domain name. Κύριο Σόσνιρτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα της ευρωπαϊκής ιδεολογίας που πρέπει να μας ε, επιδεικνύει ό,τι διακυβερνά. Ακόμα και το ίδιο που το βάζει μετά από κάθε ιστότοπο και διεύθυνση και πραγματικά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις ευρωπαϊκές αξίες. Εάν είχαμε μια πραγματική συζήτηση θα έπρεπε να μιλάμε για τις πατάτες που προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες. Ο καθένας μπορεί να πάρει ένα όνομα προτευμένο ανώτατο, τομέα ανώτατο επίπεδου. Ε, τι σχέση έχει αυτό με την πολυγλωσία, τι σχέση έχει με τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Ίσως ε, μεταφράζονται όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. αν δεν υπήρχε τέτοιου είδους μετάφραση, τι σχέση θα είχε αυτό όμως με την αγορά του ονόματος τομέα. Είναι τόσο γελία όλα αυτά που πραγματικά μου προκαλούν γέλια. Ευχαριστούμε κυρία Μαγέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για τον Brexit, ε, η διεύθυνση τελεία EU θα χαθεί μέσα σε ένα βράδυ στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι μια διεύθυνση που εγώ χρησιμοποιώ και πολλοί άλλοι. Ε, θα είναι ένα πρόβλημα λοιπόν αυτών και θα έχει και οικονομικές συνέπειες. Εγώ καταλαβαίνω τις ε, οικονομικές πιέσεις σε τοπικές κυβέρνησεις χάνονται οι επαφές, οι συνεννοήσεις, τα στοιχεία. Τη κυβερνήσει. Όμω εδώ μα έχουν πρίξει με το Brexit και το ήπιο, το σκληρό, το ναι Brexit μηδενικό καθόλου πολύ. Ε, τι θα κάνουν οι τοπικέ επιχειρήσει, τι θα γίνει στα ανατολικά τη Αγγλία. Εδώ λοιπόν σα καλώ να σκεφτούμε κατεπηγόντω ότι είμαστε ένα διεθνή πρωταγωνιστή ε, στον τομέα τη παραγωγή, στι επιστημονικέ κοινότητε, στην έρευνα. Θα πρέπει να ε, κρατήσουμε τη διεθνή αυτή, αν θέλουμε να είμαστε πάλι ε, πρωταθλητέ στον κόσμο. Ευχαριστούμε. Περνάμε στι επεξηγήσει ψήφων για την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Ο κύριο Ιλουάγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη έχουμε ψήφισμα για την Βενεζουέλα. Όμως αυτές δεν βοήθησαν καθόλου την κρίση στη χώρα. Με την αναγνώριση του αυτών Γουαϊδό, εσεί τώρα αναγνωρίζεται ένα παραξικόπημα και θέλουν να φτάσουν ακόμα και σε εμφύλιο πόλεμο μέσω στρατιωτικής εισβολής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ενώπιον του ΟΗΕ να γίνει ουρά του Τραμπ για να υπάρξει παρέμβαση. Είναι διμερής αυτή η αναγνώριση που αποτελεί όμως λάδι στη φωτιά. Εξάμεινο έως ένα χρόνο ε, λέμε για εκλογές αλλά ε, λέει το Σύνταγμα της χώρας για 30 μέρες. Ε, θα πρέπει ο Πρόεδρος να εφαρμόσει το Σύνταγμα της χώρας που προεδρεύει. Θέλουμε διάλογο, θέλουμε δημοκρατία, ειρήνη και όχι να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά των πολέμων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα κατά, λέει η κυρία Μπερμό, για την Βενεζουέλα. Διότι δυστυχώς τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραβιάσει τις κόκκινες γραμμές όσον αφορά την τήρηση του ιδανούς δικαίου. Για άλλη μια φορά γινόμαστε ουρά τον ε, είπα. Ε, γινόμαστε και εμείς πολεμοκάπηλοι ε, γιατί πρόκειται για ένα πραξικόπημα ε, χτυπητό. Θα, δεν είναι δυνατόν ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα να δικαιολογήσουμε αυτά τα οποία κάνουμε. Σαουδική, Αραβία, Μαρόκο και άλλες χώρες με τις ευλογίες σας κάνανε τα ίδια για το πετρέλαιο γίνονται όλα μα ε, δεν σας νοιάζει να λερώ τα χέρια σας με αίμα ή με πετρέλαιο άρα έχουμε το, την, τον αποκλεισμό και θα πρέπει να υπάρχει επικοδομητικός διάλογος να υπάρξει η ειρήνη, να τηρηθεί το διεθνές ε, δίκαιο και να κάνουμε ό,τι επιτάσσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Κύριε Σπυράκη. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ένα σαφές και καθαρό μήνυμα. Στη Βενεζουέλα το καθεστώς Μαδούρο σκοτώνει ανθρώπους στο δρόμο επειδή διαφωνούν με τις απόψεις του. Στη Βενεζουέλα οι άνθρωποι δοκιμάζονται από τη στέρηση βασικών αγαθών και ελευθεριών. στη βενεζουέλα διώκονται και φυλακίζονται δημοσιογράφοι. στη βενεζουέλα δοκιμάζονται οι αξίες μας οι ευρωπαϊκές αξίες αυτές που μας ενώνουν και είμαστε εδώ. είναι λοιπόν απαραίτητο να πρωτοστατούμε ως κοινοβούλιο ζητώντας την αναγνώριση του ενδιάμεσου προέδρου της ενδιάμεσης ηγεσίας που θα οδηγήσει σε ελεύθερες δίκαιες και αξιόπιστες εκλογές είναι απαραίτητο να καλούμε το συμβούλιο να κινηθεί άμεσα και συνεκτικά. καμία αμφιβολία κανένας ενδιασμός καμία εκλεκτική συγγένεια με το καθεστώς μαδούρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να μειώσει την αποφασιστικότητα της ευρωπαϊκής ένωσης. ευρώπη και μαδούρο δεν πάνε μαζί. αυτό πρέπει να το ακούσουν όλοι οι πολίτες της βενεζουέλας νιώθοντας τη στήριξη της ευρωπαϊκής ένωσης. Ε, Κυρία ε, ε, Στην Ευρωπαϊκή Αριστερά καταψηφίσαμε το ψήφισμα του ΕΛΚ Σοσιαλδημοκράτων και Φιλελευθέρων για τη Βενεζούλα. Προφανώς, διότι είναι ένα ψήφισμα που αναγνωρίζει τον πραξικοπηματία Χουάν Γκουαϊδό ως πρόεδρο. Και γιατί το πράττει, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχουν ζώσει τα φίδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και γι' αυτό χρηματοδοτεί κέντρα βασανιστήριων για μετανάστες στη Λιβύη ε, φτιάχνει φράχτες ε, με ξηράφια ε, ή δεν αφήνει τα σκάφη να βγουν στη θάλασσα για να σώζουν τον κόσμο. Ανησυχεί πάρα πολύ, την έχουν ζώσει τα φίδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά στη Βενεζουέλα. Άλλο επιχείρημα για να αναγνωρίσει τον πραξικοπηματία είναι επειδή σέβεται πάρα πολύ και εκτιμά τη δημοκρατία. Και γι' αυτό έχει προτιμησιακή οικονομική συμφωνία με ένα μοντέλο τόσο ε, δημοκρατικό όπως η απολυταρχική δημοκρατία, βασιλεία συγγνώμη, της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα στηρίζεται ένα αυτοανακηρυχθέντα πρόεδρο έτσι, ε, χωρίς εκλογές και τίποτα άλλο, γιατί ο Μαδούρο είναι τύρανος και ε, αφήνει το λαό του να λιμοκτονήσει. Και όχι ο πρόεδρος του Σουδάν που έχουμε υπογράψει τόσες συμφωνίες του τελευταίους μήνες, που μόνο δύο εντάλματα σύλληψης εκκρεμούν εις βάρος του, από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και επίσης ανησυχούν πάρα πολύ, λέει, γιατί δύο εκατομμύρια Βενεζολάνοι ε, είναι στην εξορία. Αντίθετα, το Ισραήλ είναι σχεδόν ένα κόμμα με ε, με, κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχει μόνο 5 εκατομμύρια Παλαιστίνιους άνδρες και γυναίκες ε, πρόσφυγες η στήριξη του πρα, πραξικοπήματος δεν έχει καμιά σχέση με το πετρέλαιο, ούτε ότι είναι παρακολούθημα η Ευρωπαϊκή Ένωση των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε ε, ε μάλλον ότι έχει μια κυβέρνηση Βενεζουέλα που δεν ακολουθεί τις νεοφιλελεύθερες επιταγές τους. Ευχαριστώ. Κύριος... Ευχαριστούμε κύριο Σφαρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού. Ήμουν από τους συντάκτες διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 20 Μαΐου 2018 δεν είχε αναγνωρίσει την διεξαγωγή νόμιμων εκλογών στη Βενεζουέλα, οπότε δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει τώρα την νόμιμη ανάλυση της εξουσίας από τον κύριο Γουαϊντό και μαζί με τις υπόλοιπες ε, χώρες ε, μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την κατανόηση σε αντίθεση με την ε, Ρωσία, την Κίνα και τους υπόλοιπους που δεν αναγνωρίζουν. Ο κύριος Μαδούρο έχει αναλάβει από το 2015. Εδώ θέλουμε να επιστρέψει το κράτος δικαίου και η δημοκρατία στη χώρα, να πάψει η διαφθορά και να μην, επιτρέπει, να μην υποχρεώνονται οι πολίτες της χώρας να φεύγουν προς τα σύνορα για να σωθούν με τις οικογένειες και τα παιδιά τους. Θέλουμε η δημοκρατία να επικρατήσει και να μπορεί ο λαός να καθορίσει το πεπρωμένο δεδομένο το Δεν μπορούν οι εκκλήσει του λέω αυτό να αγνοούνται. Θα πρέπει ε, τα πολιτικά δικαιώματα, ε, όπω θέλει να τα αποκαταστήσει ο κύριο Γουαϊδό με το το Δικαστήριο, να ε, επιτραπεί και να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι που ε, συνελήφθησαν από τον κύριο Μαδούρο αυτέ τι μέρε. Μεταξύ των οποίων Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι. Ευχαριστούμε. Εγώ Να μην ψηφίσω κατά γιατί δεν ήθελα να υπερασπιστώ ένα κομμουνιστικό καθεστώ ακριβώς όπως έκανε η αριστερή πτέρυγα, η κόκκινη συνάδελφοι. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σας θυμίσω την Μολδαβία. Η κυβέρνηση στην Μολδαβία έκανε πραξικόπημα και το ίδιο έγινε και στο Σουδάν. Α μην έχουμε νομική πίστη των πραγμάτων, να είμαστε υποκριτές, γιατί το θέμα είναι η ελευθερία του λόγου και η περιστολή για τους ε, ευρωβουλευτές, ενώ δεν ισχύει αυτή η ελευθερία άλλου στον ε, κόσμο. Γιατί να κατεβόμαστε με όλα, ενώ δεν ξέρουμε τα θέματα. Ας κοιτάμε τα του οίκου μας καλύτερα. Πυρίνσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. It should be crystal clear. Θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο ότι ο μόνος τρόπος να λυθεί το σημερινό πρόβλημα, η σημερινή κρίση είναι διάλογος κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Αυτό το κείμενο που ψηφίσαμε πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Αντιβαίνει σε όσα έχει πει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Κόντρα σε όσα ε, λένε σε τα ΜΜΕ ότι ο πρόεδρος Μαδούρο προτίθεται να αρχίσει διάλογο. Έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά σε τρομερό βαθμό. Επικρίνουμε την κυβέρνηση για το ότι θέλει μονόπλευρες εκλογές και δεν, κάνει, δεν κανέναν για την διοργάνωσή τους και από την άλλη μεριά είμαστε υπέρ άλλων που θέλουν να κάνουν πάλι μονόπλευρα τις εκλογές ο άλλος πρόεδρος ε νομίζω ότι αυτό είναι πολύ λάθος του Κοινοβουλίου μας να λαμβάνουμε τέτοια απόφαση που απλώς κάνει την κρίση οξύτερη. Χάναν! Ευχαριστώ πολύ. Η προσέγγιση του Κοινοβουλίου στην τραγωδία της Βενεζουέλας είναι πάρα πολύ έντονη και η Προεδρία του κυρίου Ταγιάννη τα είχε επισημάνει αυτά. Εγώ μεγάλωσα το 1970 στην Νότια Αμερική και το 99 ε, ήταν πλούσια, πιο πλούσια χώρα η Βενεζουέλα, πήγαιναν όλοι εκεί πέρα, τότε που ανέβηκε σε εξουσία ο Τσάβες και τώρα έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια εκτροπισμένους έχουμε πληθωρισμό που είναι στο 10 εκατομμύρια της εκατό ετησίως και περίεργως υπάρχουν κάποιοι σοσιαλιστές και κομμουνιστές που τους ακούσαμε που ακόμα θέλουν να υποστηρίξουν το τυραννικό καθεστώς του Τσαβίστα Μαδούρο. Ε, πόσες φορές θα πρέπει να ξαναδούμε το ίδιο έργο πριν καταλάβουμε ότι το σοσιαλιστικό πείραμα είναι τόσο άτσαλο τυραννία, φτώχεια, καταστολή. Και τώρα, έκθεση Ρεμούν. Κύριος Μαριάς. Σημαντικός παράγοντας της πολιτικής ανταγωνισμού είναι οι λεγόμενες κρατικές ενισχύσεις. Και στο θέμα αυτό έχουν γίνει πραγματικά σημεία και τέρατα. Έχουν επιβληθεί πολλές ε, διατάξεις και πρόστιμα με αποτέλεσμα κυρίως η ναυπηγική βιομηχανία να έχει καταστραφεί η γνωστή ναυπηγική βιομηχανία στην ελλάδα τα ναυπηγεία σκαραμαγκά πρέπει να πληρώσουν για κρατικές ενισχύσεις 310 εκατομμύρια ευρώ. απαγορεύεται μέχρι στιγμής να χτίζουν εμπορικά πλοία. πού; στην ελλάδα όταν ο μεγαλύτερος εμπορικός στόλος έχει ελληνική σημαία. ταυτόχρονα ε, μια άλλη εταιρεία η larco αναγκάζεται με απόφαση του δικαστηρίου να επιστρέψει 135,8 εκατομμύρια ευρώ με αποτέλεσμα να κλείσει θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική γύρω από τις κρατικές ενισχύσεις να υπάρξει απαλλαγή στην ελλάδα και ιδίως σε αυτές τις επιχειρήσεις να μην επιστρέψουν τα κονδύλια αυτά και τέλος να υπάρξει ειδικό καθεστώς η ελληνική οικονομία είναι σε κρίση λόγω του μνημονίου να υπάρξουν ειδικέ ρυθμίσεις και ειδικό καθεστώς για την ελλάδα στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. ευχαριστώ. Uh, Madam President. This report rightly raises concerns about certain... Η έκθεση αυτή εγείρει ανησυχίες για την έλλειψη αντιστοιχειών μεταξύ των εθνικών φορολογικών στοιχείων και ε, συστημάτων και των στοιχείων που διαθέτουν. Πρέπει να πάψει αυτή η υποβάθμιση της ποιότητας. Οι φόροι είναι σημαντική για την επιβίωση των μεγάλων ομίλων, των μικρών ομίλων μάλλον, και όχι μόνο προς όφελος των Facebook, Amazon και ούτω καθεξής θα πρέπει ε, να είμαι, ε, θα μπορούσα να είμαι η τελευταία βουλευτής από τον Ηνωμένο Βασίλειο που θα πάρει το λόγο σε αυτή την Ολομέλεια. Θέλω λοιπόν να πω ότι είμαι υπερήφανη που πήρα μέρος στο μεγαλύτερο εγχείρημα Ειρηνή και ευημερία των ε, σύγχρονων καιρών. Και δεν θα πω ποτέ αντίο σα, αλλά εις το επανειδήν. Ο κύριος Σντρογεύσκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η ετήσια έκθεση για τον πολιτική ανταγωνισμού δεν ήταν τόσο κλασική όπως θα περίμενε κανείς, διότι αφιέρωσε ιδιαίτερη προσοχή σε πολλά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το ε, τη δημιουργία καρτέλ για την παραγωγή βαρέων οχημάτων που διοχετεύονται στην εσωτερική αγορά. Εδώ θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει όντως να καταπολεμά τις πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό όπως ε, την, ε, το πείραγμα των τιμών θα πρέπει ο ανταγωνισμός και η πολιτική του να βασίζεται στην αρχή της ίση μεταχείρισης όλων των κλάδων, όλων των τομέων, όλων των εταιριών. Το ίδιο και το, στον τομέα του άνθρακα. Θα πρέπει να έχουμε συμφωνίες ώστε μεγάλες εταιρείες ή αυτοί που ε, έχουν περισσότερες δυνατότητες να μην μπορούν να υποφελούνται από το σύστημα. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ. Εγώ απήχα στην έκθεση αυτή και στην ψηφοφορία, διότι κάποιε τροπολογίε ήταν μεν θετικέ, αλλά πιστεύω ότι ξεπερνά το πεδίο τη ε, έκθεση και του θέματο της πολιτικής ανταγωνισμού. Χρειάζεται η υλοποίηση του CCCTB και η πάυση της αρχής της ομοφωνίας της προφορίας σε φορολογικά θέματα στο Συμβούλιο. Πρέπει λοιπόν να ε, δώσουμε την απαραίτητη όθηση για να λάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση στα φορολογικά θέματα και να παραμείνει ζωντανή ισχυρή συνεργασία που υπάρχει και με το Κοινοβούλιο σε τέτοια θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ε, προστατεύσει καλύτερα τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ιδίω να τι προστατεύσει κατά των ε, αθέμητων πρακτικών. Ω μέλο του Ευρωκοινοβουλίου και τη Επιτροπή ε, Διεθνού Εμπορίου, πιστεύω ότι αυτά τα θέματα είναι ζωτική σημασία για, μια, ε, για ένα υγιέ περιβάλλον για το ευρωπαϊκό εμπόριο και να μπορούν οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να λειτουργούν ανεμπόδιστα σε αυτό. Ευχαριστούμε, κυρία Ροχόνεν Λέρνερ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε πολιτική του ανταγωνισμού είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ένα στόχο που θα πρέπει να τον επιδιώκουμε διαρκώ. Οι μεγάλε εταιρείε κοιτάζουν να φοροδιαφύγουν και έχουν πλεονεκτήματα τα οποία είναι αθέμετα σε σύγκριση με τις μικρομεσαίες. Φαίνεται να έχουν φτιάξει τους δικούς τους νόμους και να μπορούν να ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με παράνομες επιδοτήσεις ας πούμε. Όπως λέει και η έκθεση, η φοροδιαφυγή είναι κάτι το πολύ επιζήμιο για τα δημοσιονομικά των κρατών και για τους πολίτες τους ίδιους. Η εμπιστοσύνη στην Ένωση πλήττεται σοβαρά και ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε συστήματα που έχουν ωφελήσει τους πλουσίους και τις μεγάλες εταιρείες. Τα, τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να απαλείψουν αυτές τις αθέμητες πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εργαστεί για το θέμα αυτό μεν, για τις αθέμητε εμπορικέ πρακτικές και πρέπει να προβλεφθούν και κυρώσει στις περιπτώσει που διαπιστώνονται ατασταλίε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Θα ε, πω ότι υποστήριξα την έκθεση αυτή, διότι... Ε, διότι είναι σημαντικό, ε, πολλέ επιχειρηματικέ πρωτοβουλίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρήζουν ιδιαίτερε προστασίε. Πρέπει να υπάρχουν όμω γι' αυτό κοινοί κανόνε. Χρειαζόμαστε την ενιαία αγορά, αλλά και κοινού κανόνε. Θέλουμε να θαρρύνουμε του επιχειρηματίε, του νέου, του ανθρώπου που θέλουν να εργαστούν τίμια. Να θυμίσω εδώ το σκάνδαλο του πακέτου τη ακινητικότητα ε, για το θέμα αυτό. Είναι κατά του ανταγωνισμού, τη αρχή του ανταγωνισμού, του θεμητού ανταγωνισμού και θέλουν να πάρουν τι εταιρείε από κάποιου για να τι δώσουν σε άλλου αυτοί που θα εγκρίνουν. Ε, το πακέτο λοιπόν τη κινητικότητα, το πακέτο μακρόν όπω το έχουμε ονομάσει, θέλει να πάρει την ε, δουλειά από την ε, Ανατολική Ευρώπη και να την πάρει στην Κεντρική. Αυτό για μα σημαίνει τουλάχιστον μισό εκατομμύριο μετανάστε που θα φύγουν από τη χώρα αναγκαστικά για να δουλέψουν. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Και τελευταίο για να κλείσουμε, κύριο Πόλτσακ. Περιμένω το τέλο τη διερμηνία για να σα δώσω το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ε, θέλω να εξηγήσω πώς ψήφισα. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή. Εχθές στη συζήτηση για την πολιτική ανταγωνισμού συμφωνήσαμε ότι σε ε, ε, πολλές περιπτώσεις έχουμε πρόοδο και χαίρομαι γι' αυτό. Η ενιαία αγορά και ο ανταγωνισμό για την ενιαία αγορά κυριαρχούν στη συγκεκριμένη έκθεση. Θα πρέπει όμω να προστατεύουμε και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Καλό ο ανταγωνισμό, αλλά να προστατεύουμε του καταναλωτέ από τον αθέμητο ανταγωνισμό. Αυτό είναι ένα από τα καλά τη έκθεση. Στη συνέχεια. Εκφράζουμε την άποψη ότι οι αγορές οφείλουν να προσαρμόζονται στις ε, συνθήκες και να προστατεύουν το περιβάλλον. Δηλαδή υπάρχει και ένα στοιχείο βιωσιμότητας και αηφορίας, πάρα πολύ σημαντικό ε, και ιστοδυνικές. Δεν θα πρέπει να πούμε μετά από μένα στο χάος δηλαδή, για πυρημιχθή του. Ευχαριστώ. Τελειώνουν εδώ οι επεξηγήσεις ψήφου. Ε, τα πρακτικά θα διανεμηθούν και θα εγκριθούν στην αρχή της επόμενης συνόδου και αν δεν διαφωνείτε θα ε, διαβιβάσω αμελητή στους δικαιούχους και στους τελικούς αποδέκτες στα κείμενα. Διακόπτεται η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λέει τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ.